Uh, Αγαπητοί συνάδελφοι, θα ήθελα να συνεχίσουμε τη συνεδρίαση. Μια μισή ώρα είχαμε στη διάθεσή μας, ε, τώρα έχουμε μία ώρα και 20 λεπτά και νομίζω ότι είναι σημαντική η ακρόαση αυτή για το Brexit. Πρωτού προχωρήσουμε όμως στην ακρόαση. Ο πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου μου είπε να σας ενημερώσω ότι την επόμενη εβδομάδα θα γίνει διάσκεψη κορυφής ε, αρχηγών κρατών και κυβερνήσεων ε, Αφρικής Ευρωπαϊκής Ένωση 29 ε, και 30 Νοεμβρίου στην ακτή του Ελεφαντοστού. Και αυτό αποτελεί μοναδική ευκαιρία να ενισχύσουμε την εταιρική μας σχέση με χώρες της Αφρικής. Δεν νομίζω ότι χρειάζεται να αναπτύξω περαιτέρω το θέμα αυτό. Θα ήθελα όμως να σας ενημερώσω ότι η διάσκεψη των Προέδρων αποφάσισε αυτή η εβδομάδα να είναι εβδομάδα Αφρικής στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και αύριο θα πραγματοποιηθεί διάσκεψη υψηλού επίπεδου για την Αφρική στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο μία εβδομάδα πριν τη διάσκεψη κορυφής. Η συζήτηση θα έχει να κάνει με τη δημοκρατία, τη διακυβέρνηση, τα ανθρώπινα δικαιώματα. Αυτά είναι τα θέματα που άπτονται των θεμάτων της ΑΦΚΟ και θα είναι χρήσιμο να έχουμε τις ε, συνεισφορές σας ε, για την ε, συνάντηση αυτή και της επόμενης εβδομάδας. Ως ΑΦΚΟ δεν έχουμε θέματα που συνδέονται άμεσα με την Αφρική, αλλά είχαμε κάποιες συνεργασίες πάνω σε εκδηλώσεις που έλαβαν χώρα εντός του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και ελπίζω ότι στο μέλλον θα έχουμε ακόμα περισσότερες τέτοιες επαφές. Η ΑΦΚΟ είναι διατεθειμένη να συνεργαστεί με τους συναδέλφους μας ε, από την Αφρική, ε, όπου θεωρούμε ότι αυτό θα είναι χρήσιμο για την ανάπτυξη δημοκρατικών θεσμών. Μπορεί να θυμάστε ότι πριν κάποιο διάστημα η συντονιστές είχαν ε, συζητήσει το θέμα της ε, πολυεπίπεδης ε, διακυβέρνησης. Και στις ομοσπονδιακές εκλογές υπάρχουν ακριβώς οι υπερεθνικοί κατάλογοι. Είναι ένα από τα λίγα παραδείγματα στον κόσμο. Προχωράμε τώρα στο σημείο 6 της ημερήσιας διάταξης. Ε, πρόκειται για ακρόαση για το Brexit και το θέμα της δικαιοδοσίας όσον αφορά τη Συμφωνία Αποχώρησης και τη Συμφωνία Μελλοντικής Σχέσης μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και του Ηνωμένου Βασιλείου. Έχουμε δύο μελέτες που ανατέθηκαν από το Τμήμα Πολιτικής ε, για ε, τις συνταγματικές υποθέσεις ε, και έχουμε εδώ δύο καθηγητές, ε, τον κύριο Αντώνιο Φρανσίσκο Φερνάντες Τομάς, που έχει εκπονήσει τη μελέτη με θέμα επίλυση των διαφορών που προκύπτουν από την αποχώρηση του Ηνωμένου Βασιλείου από την Ευρωπαϊκή Ένωση και τον καθηγητή Steve Pierce, που θα μιλήσει σχετικά με τη δικαιοδοσία πριν και μετά την αποχώρηση του Ηνωμένου Βασιλείου από την οπτική της συνταγματικής τάξης του Ηνωμένου, Βασιλείου. Έχουμε πολύ λίγο χρόνο στη διάθεσή μας για τις παρουσιάσεις και για τη συζήτηση. Θα ήθελα λοιπόν να ζητήσω πρώτα από τον καθηγητή Αντώνιο Φρανσίσκο Φερνάντες Τόμας να μας παρουσιάσει τη μελέτη του. Κατόπιν θα ακούσουμε την βρετανική πλευρά από τον καθηγητή Steve Pierce. Κύριε Τομάς, έχετε το λόγο. Κύριε Πρόεδρε, κυρίες και κύριοι Ευρωβουλευτές, με μεγάλη ικανοποίηση και τιμή βρίσκομαι εδώ σήμερα στην Επιτροπή σας Συνταγμαστικών Υποθέσεων του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου προκειμένου να σας παρουσιάσω την έκθεση αυτή. Και είναι η δεύτερη φορά που έρχομαι εδώ στην Επιτροπή σας φέτος. Θα σας συνοψίσω την έκθεσή μου ξεκινώντας από τέσσερις διαπιστώσεις. Πρώτον, όπως είναι γνωστό, προβλέπεται η αποχώρηση του Ηνωμένου Βασιλείου είναι οδηγήσει σε δύο συμφωνίε. Η μία είναι η συμφωνία ακριβώ απόσυρση και η δεύτερη είναι η συμφωνία για τι μελλοντικέ σχέσει. Η κάθε μία από αυτέ αποτελεί ένα χωριστό τμήμα. Τώρα στη συνέχεια θέλω λιγάκι να ξεκαθαρίσω τους όρους της έννοιας. Σήμερα περιμένατε μια έκθεση συνεχεια θελω λιγακι να ξεκαθαρισω του ορου τι εννοιε σημερα περιμενατε μια εκθεση διχως αλλο για τη δικαιοδοσία και έχετε να κάνετε τελικά με μια έκθεση που αναφέρεται στην διευθέτηση διαφορών. Η δικαιοδοσία είναι κάτι πιο απλό, αλλά δεν μπορεί κανείς να προσφύγει σε αυτή σε διεθνές επίπεδο. Γι' αυτό και η έκθεσή μου είναι ευρύτερη και αναφέρεται στην δικαιοδοσία και σε άλλες διαδικασίες διευθέτησης διαφορών εν ώψη της αποχώρησης του Ηνωμένου Βασιλείου. Στη συνέχεια, όσον αφορά τη μεθοδολογία, αποφάσισα να χρησιμοποιήσω κάτι διαφορετικό από ό,τι χρησιμοποιούν συνήθως τα όργανα. Ξεκινάω λοιπόν την μελέτη μου από τη συμφωνία για το μελλοντικό νομικό πλαίσιο και όχι από τη συμφωνία απόσυρσης. Και αυτό γιατί έτσι πιστεύω ότι ξεκινώ από κάτι γενικότερο και πάω σε κάτι ειδικότερο. Μετά την αποχώρηση θα είναι μια τρίτη χώρα το Ηνωμένο Βασίλειο για την Ευρωπαϊκή Ένωση και οι σχέσεις της χώρας αυτής μαζί μας, γενικά μιλώντας, θα διευθετούνται από το Διεθνές ε, Δημόσιο Δίκαιο, εκτός από τις περιπτώσεις εκείνες που περιλαμβάνονται στη μεταβατική περίοδο και που θα αναφέρονται στην Συμφωνία Απόσυρσης. Και εκεί, κατ' εξαίρεση, θα εφαρμόζεται το δίκαιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Όμως, μόνο όσο ισχύει αυτή η μεταβατική περίοδος. Όμως, παρά την διαφορετική μεθοδολογία που ακολουθώ, κατά τα άλλα ακολουθώ ε, τις θέσεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Τώρα μετά από αυτά τα προκαταρτικά πρέπει να έχουμε υπόψη μας το θέμα της ασυμμετρίας. Είναι ένα γενικό πρόβλημα σε διεθνείς συμφωνίες που συνάπτει η Ευρωπαϊκή Ένωση. Και άρα έχει να κάνει και με τις δύο αυτές συμφωνίες που σας ανέφερα όσον αφορά το Ηνωμένο Βασίλειο. Είναι συμμετρική η σχέση διότι με την κατάσταση αυτή μια χώρα βρίσκεται για ένα διάστημα τουλάχιστον με το ένα από μέσα με το ένα έξω. Στις διάφορες διεθνείς συμφωνίες που έχει συνάψει η Ευρώπη με τρίτες χώρες δεν αναγνωρίζουν την ε, δικαιοδοσία του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου εκτός της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Αντίθετα, μέσα στην Ευρωπαϊκή Ένωση τέτοιες συμφωνίες περιλαμβάνουν το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο και έχει πλήρη δικαιοδοσία το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο για την εφαρμογή τέτοιων συμφωνιών. Μετά λοιπόν από αυτά θα περάσω στο σημείο 3 της σύνοψης. Λοιπόν, για τη σχέση αυτή, την μελλοντική, τη συμφωνία για τη μελλοντική σχέση, θα πρόκειται για μια διεθνή συμφωνία, όπω οποιαδήποτε άλλη διεθνή συμφωνία έχει η Ευρωπαϊκή Ένωση με τρίτη χώρα. Άρα εφαρμόζονται τα συνήθει σε τέτοιε συμφωνίε, που δεν περιλαμβάνουν τη δικαιοδοσία κανενό δικαστηρίου αλλά μόνο πιο ευέλικτα μέσα διευθέτησης διαφορών όπως είναι η διαιτησία. Κάτι αντίστοιχο θα συνέβαινε και κατά την τελική περίοδο ισχύω τη συμφωνία απόσυρση, δηλαδή όταν δηλαδή θα έχει τελειώσει η μεταβατική περίοδο. Και έτσι οδηγούμαστε στην διατήρηση της δικαιοδοσίας του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου στις διαφορές που μπορεί να απορρέουν από την εφαρμογή της Συμφωνίας Απόσυρσης κατά την μεταβατική περίοδο. Δεύτερον, και αυτό είναι αποφασιστική σημασία, το κλειδί έχει να κάνει με το αν ή όχι θα υπάρχει εφαρμογή του ευρωπαϊκού δικαίου στο Ηνωμένο Βασίλειο, ακόμα και όταν θα έχει αποχωρήσει από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Γιατί αν στη Συμφωνία Απόσυρση λέει ότι θα εφαρμόσετε το δίκαιο τη Ένωση, τότε αναγκαία αυτό μα οδηγεί στη δικαιοδοσία του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου τη Ευρωπαϊκή Ένωση. Άρα λοιπόν υπάρχουν δύο δυνατότητε. Η μία δυνατότητα, αν η συμφωνία Απόσυρση περιλαμβάνει μεταβατική περίοδο, τότε πρέπει να έχουμε τη δικαιοδοσία του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου. Και γιατί, γιατί δεν μπορούμε να διακρίνουμε το ευρωπαϊκό δίκαιο από τους μηχανισμούς που το εγγυώνται αυτό. Και όπως έχουμε πει, έχει πει πολλές φορές στην ομολογία του Ευρωπαϊκού Δικαστήριο, το Δικαστήριο του Λουξεμβούργου έχει το μονοπόλιο, την αποκλειστική δηλαδή αρμοδιότητα, να διασφαλίζει αυτόνομα, να ερμηνεύει ε, το δίκαιο στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Τώρα υπάρχει και μια δεύτερη δυνατότητα. Αν η συμφωνία ποσέση δεν περιλαμβάνει καμία μεταβατική περίοδο, αλλά παρόλα αυτά χρειάζεται ερμηνεία κάποιων διατάξεων του ανοσιακού δικαίου, για παράδειγμα των διατάξεων από τις οποίες απορρέουν οι υποχρεώσεις πληρωμών του Ηνωμένου Βασιλείου, τότε η αρμόδια αρχή θα εξακολουθούσε να είναι το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο. Κατόπιν τούτων τώρα έρθω στην Συμφωνία Μελλοντικής Σχέσης της Ευρωπαϊκής Ένωσης με το Ηνωμένο Βασίλειο. Τρία πράγματα έχω να πω εδώ. Πρώτον, μέσα στις συμφωνίες που συνάπτει η Ευρωπαϊκή Ένωση με τρίτες χώρες, ε, μπορούμε να διακρίνουμε διάφορες κατηγορίες. Αν η συμφωνία είναι με μια μακρινή χώρα και δεν δημιουργεί καμία ολοκληρωμένη δομή σχέσης, ας πούμε με τη Σιγκαπούρη, ή με τον Καναδά οι συμφωνίες με την Ουκρανία και τη Μολδαβία. Οι μηχανισμοί διευθέτησης διαφορών είναι ευέλικτοι και βασίζονται στις διαπραγματεύσεις, τη διαμεσολάβηση, τη διατησία. Η συμφωνία δεν έχει άμεσες επιπτώσεις. Η κοινή διακρατική επιτροπή έχει περιορισμένες αρμοδιότητες και εάν δεν καταφέρει να διευθετήσει την διαφορά, τότε το θέμα πάει σε ένα πάνελ διατησίας. Σε πολλές περιπτώσεις, Σιγκαπούρη, Καναδά, επιπλέον υπάρχει και μία ειδική διαδικασία για τη διευθέτηση διαφορών μεταξύ επενδυτών και χωρών. Άμεση διαιτησία. Ωραία, τώρα, το κατά πόσο διατάξεις αυτές είναι συμβατές, κυρίως το άρθρο 8 σίγμα τη της συμφωνίας με τον Καναδά, με τις ε, συνταγματικές συμφωνίες που έχουν να κάνουν και με θεμελιώδη δικαιώματα, αυτό έχει αφισβητηθεί από το Βέλικο Δικαστήριο που ζήτησε ε, προδικαστικό ερώτημα έστειλε στο δικαστήριο για να ε, πάρει απάντηση και έτσι φαίνεται ότι το θέμα των θεμελιωδών δικαιωμάτων των Ευρωπαίων πολιτών δεν λύνεται με τη συμφωνία αυτή με τον Καναδά και άρα θα πρέπει να υπάρχει ένας ανεξάρτητος δικαστής. Έπειτα, το κλίμα αυτό ευελιξίας δεν υπάρχει εφόσον η συμφωνία με τρίτη χώρα, κοντινές χώρες στην Ευρωπαϊκή Ένωση, δημιουργεί μία δομή ολοκλήρωσης με τρίτες χώρες και μέσα στη δομή αυτή τότε υπάρχουν ειδικοί μηχανισμοί διευθέτησης. Αυτό συμβαίνει για παράδειγμα στην περίπτωση του οικονομικού χώρου. Θα θυμόσαστε, και συμμετέχουν η Νορβηγία, η Ισλανδία κλπ. Τι έχουμε εκεί. Έχουμε ένα δικαστήριο που είναι το δικαστήριο το, του χώρου ελεύθερων συναλλαγών και το οποίο φέρει σε πέρα στην αποστολή του με εγγύσεις αντίστοιχες για τους πολίτες και τους διάφορους φορείς. Γιατί δεν υπάρχει ευελιξία σε αυτή την περίπτωση, θα με ρωτούσατε. Γιατί είναι αναγκαία η εφαρμογή ίδιων κανόνων σε δύο διαφορετικά πλαίσια, δηλαδή της Ευρωπαϊκή Ένωση και του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου. Και αυτοί οι κανόνες που πρέπει να είναι ίδιοι αλλά σε δύο διαφορετικά πλαίσια θα πρέπει να τυχαίνουν ίδιας ερμηνείας από όλους. Άρα λοιπόν ποιος θα μπορούσε καλύτερα να ερμηνεύσει με τον ίδιο τρόπο τα πράγματα από ότι το δικαστήριο αυτό. Τώρα το μια τρίτη χώρα ε, ρωτάει κάτι το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο, ζητάει μια ερμηνεία δηλαδή, όντα τρίτη χώρα, αυτό είναι μια εξαίρεση. Εξαίρεση στα όσα προβλέπονται στο άρθρο 267 της Εθήκης για την Ευρωπαϊκή Ένωση, που βάζει δύο προϋποθέσεις, όπως γνωρίζουμε, να είναι ένα δικαστικό όργανο και να είναι χώρας μέλους που στέλνει το προδικαστικό ερώτημα. Ο κανόνας αυτός όμως έχει κάποιες εξαιρέσεις. Στο πρώτο τμήμα της μελέτης μου ε, καταδεικνύω τρεις εξαιρέσεις. Πρώτο, το πρωτόκολλο 34, παράρτημα α για τον ε, ΕΟΧ. Η διάταξη που ισχύει για τον κοινό χώρο ε, Ευρωπαϊκής Αεροπορίας, που συμμετέχουν και τρίτες χώρες, και η συμφωνία σύνδεσης με την Ουκρανία και τη Μολδαβία. Σε αυτές τις περιπτώσεις ένα δικαστικό όργανο εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης ή ακόμα και ένα πάνελ διαιτησίας όπως της Ουκρανίας και της Μολδαβίας μπορεί να στείλει προδικαστικό ερώτημα στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Εξίσου. Γιατί, για να πετύχει μία ενιαία ερμηνεία ενός κανόνα που εφαρμόζεται σε δύο διαφορετικά πλαίσια. Στην πρακτική λοιπόν εφαρμογή συμφωνιών ε, με τρίτες χώρες έχουμε αυτές τις τρεις εξαιρέσεις. Οπότε γιατί να μην σκεφτούμε ότι θα βάλουμε και μια τέταρτη εξαίρεση για την περίπτωση του Ηνωμένου Βασιλείου εφόσον αποχωρήσει. Και αυτό εφόσον θα υπάρχει μεταβατική περίοδος κατά την οποία θα εφαρμόζεται στο Ηνωμένο Βασίλειο το Ευρωπαϊκό Δίκαιο. Αυτή είναι λοιπόν η εσωτερική λογική που ακολούθησαν τα ευρωπαϊκά θεσμικά όργανα. Αλλά είναι και η εξωτερική λογική εξαιτία των συμφωνιών τη Ευρωπαϊκή Ένωση με τρίτες χώρες. Δηλαδή να υπάρχει μια ερμηνεία για το δίκαιο και την ερμηνεία αυτή να την κάνει πάντα το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο εφόσον πρέπει να υπάρχει ενιαία ερμηνεία ενός κανόνα που εφαρμόζεται σε δύο διαφορετικά πλαίσια. Τώρα έρχομαι στη Συμφωνία Απόσυρσης. ακολουθώντας πάντα τα όσα λέει η περίληψη της εκθεσής μου. Στη μεταβατική περίοδο τώρα και ποιος είναι ο ρόλος του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου κατά τη διάρκεια αυτής. Υπάρχει λοιπόν, θα υπάρχει μάλλον, μάλλον μια μεταβατική περίοδος και εφόσον υπάρχει, γιατί θα υπάρχει, για να παρατείνει την περίοδο κατά την οποία ε, κάποιες ευρωπαϊκές διατάξεις όσον αφορά την ηθαγένεια, τον εσωτερικό χώρο κτλ. να εφαρμόζονται αυτά και στο Ενωμένο Βασίλειο. Να υπερισχύουν οι κανόνες αυτοί δηλαδή από οτιδήποτε άλλο αποφασιστεί με την απόσυρση. Να διασφαλιστούν δηλαδή εγγύησεις που προσφέρει το ευρωπαϊκό δίκαιο στους ιδιώτες, ώστε να μπορούν να επικληθούν το δίκαιο αυτό, αν έχουν κάποια διαφορά. Επίσης όμως, ο στόχος είναι να ε, διατηρηθεί η νομολογία του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου και να διατηρηθεί και σχέση συνεργασίας ανάμεσα στο Ευρωπαϊκό Δικαστήριο και τους δικαστές του Ηνωμένου Βασιλείου. Πάντα για να μπορεί να υπάρχει αυτή η δυνατότητα προδικαστικών ερωτημάτων. Και τρίτον, αυτό σημαίνει ότι διατηρείται η ισχύ του κανόνα που βάζει την ευθύνη στο κράτος εφόσον υπάρξει παραβίαση κανόνων της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Υπήρχε μια τέτοια περίπτωση παλιότερα. Το μήνυμα λοιπόν είναι ότι το καλύτερο για την Ευρωπαϊκή Ένωση και τους πολίτες της είναι να διατηρηθεί η νομολογία του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου και οι σχέση συνεργασίας ανάμεσα στα εσωτερικά δικαστήρια του Ηνωμένου Βασιλείου και το δικαστήριο του Λουξεμβούργου μέχρι το τέλος της μεταβατικής περίοδου. Δεύτερον, πώς θα μπορούσαμε να ενισχύσουμε τους στόχους αυτούς και με αυτό θα τελειώσω. Εξαρτάται βέβαια, αλλά κατά τη γνώμη μου, για να βελτιωθεί η θέση της Ευρωπαϊκής Ένωσης κατά τις διαπραγματεύσεις, το καλύτερο θα ήταν το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο να ζητούσε από το Δικαστήριο νομοδότηση... βάσει του 218.11. Και αυτό θα είχε πλεονεκτήματα αλλά και μειονεκτήματα. Το πλεονέκτημα θα ήταν ότι το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο έτσι θα μπορούσε να υιοθετήσει ε, τέτοια πρωτοβουλία υπέρ των Ευρωπαίων πολιτών απέναντι σε οποιαδήποτε χώρα. Θα μπορούσε να τα κατοβέλει οτιδήποτε άλλο. Αν κάποιος πρέπει να υποστηρίξει τα δικαιώματα των Ευρωπαίων πολιτών, προτιμότερο είναι να μπορεί να το κάνει αυτό το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο παρά μια χώρα, το Βέλγιο ή οποιαδήποτε άλλη. Δεν χρειάζεται όμως να περιμένουμε ένα τελικό κείμενο που να έχει υπογραφεί για τη Συμφωνία Απόσυρσης. Το δικαστήριο με τις πληροφορίες που έχει στη διαθεσή του μπορεί πάντα να αποφασίσει. Αυτό στο 1.09 του 2011 το είπε το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο. Οπότε, αν με ρωτήσετε πότε το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο μπορεί να ζητήσει τη γνωμοδότηση αυτή, στην πράξη, παρόλο που δεν το λέει αυτό η νομολογία του δικαστηρίου, μπορείτε να το κάνετε από τη στιγμή που υπάρχει ένας ε, πρώτος που το ζητάει. Τώρα, μετά θα μπορούσαμε να ζητήσουμε, να δούμε πώς συνάδει το περιεχόμενο της συμφωνίας απόσυρσης με τις συνθήκες που υπάρχουν ήδη συμπεριλαμβανομένων και των θεμελιωδών δικαιωμάτων. Στο 2.3 για την Σύμβαση Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων και την Ίστο Βαρκής Ένωσης εκεί υπάρχει ένα παράθυρο. Στην ομολογία του το δικαστήριο είπε ότι θα μπορούσε να αποφανθεί όχι μόνο για το περιεχόμενο της συμφωνίας, αλλά και για το τι θα έπρεπε να συμπεριλαμβάνεται σε αυτό που είναι κάτι πολύ ευρύτερο. Συνεπώς, είναι πολύ, ε, πολύ ευρύες οι δυνατότητες που δίνει στον εαυτό του το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο. Οπότε, με την ομολογία αυτή το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο θα μπορούσε να πάει ακόμα πιο μακριά εφόσον του υποβληθεί έτοιμα για γνωμοδότηση για να δει κατά πόσο στη Συμφωνία Απόσυρσης προστατεύονται τα δικαιώματα των Ευρωπαίων πολιτών. Τώρα, τα μειονεκτήματα. Αν ζητήσουμε γνωμοδότηση από το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο, αυτό σημαίνει ότι το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο βάζει κάποιε αυστηρέ κόκκινε γραμμέ και μπορεί να μην τι δεχτεί το Ηνωμένο Βασίλειο. Οπότε μπορεί να οδηγήσει αυτό σε αποτυχία τη συμφωνία απόσυρση. Όμω δεν είναι αυτό ο μόνο κίνδυνο που υπάρχει. Υπάρχει και άλλο πολιτικό κίνδυνο. Αν για να αποφύγουμε να έχουμε ε, την γνωμοδότηση αυτή του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου δώσουμε περισσότερα πλεονεκτήματα στην χώρα που φεύγει από ότι μειονεκτήματα, αυτό θα μπορούσε να προωθήσει άλλες δυσαρεστημένες χώρες να σκεφτούν και αυτές να αποχωρήσουν από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Μιλάμε για μια μεταβατική περίοδο που ο Υπουργός Εξωτερικών της Ιρλανδίας είπε ότι μπορεί να είναι πέντε χρόνια προχτές. Ο πολιτικός κίνδυνος λοιπόν υπάρχει και θα πρέπει να εκτιμηθεί κατάλληλα. Τίποτα άλλο. Ελπίζω να ήταν χρήσιμα τόσα. Σας είπα, σας ευχαριστώ πολύ για την προσοχή σας και είμαι στη διάθεσή σας για να απαντήσω σε ό,τι ερωτήσεις έχετε. Ευχαριστώ. Thank you. Ε, Ευχαριστούμε πολύ. Περνάμε αμέσω στον κύριο Στίβ για να μας παρουσιάσει τις δικές του απόψεις επί του θέματος. Εκτός μικροφώνου μιλητής. Ευχαριστώ πολύ που με καλέσατε. Ευχαριστώ. Αρχικά θα σας δώσω τις θέσεις της κυβέρνησης του Ηνωμένου ε, Βασιλείου, παρότι δεν βρίσκομαι εδώ εξ ονοματός τους, για να σας παρουσιάσω την νομική θέση στο Ηνωμένο Βασίλειο και γιατί η Βρετανική κυβέρνηση υιοθετεί τις απόψεις που υιοθετεί σε σχέση με τη δικαιοδοσία του δικαστηρίου. Η αφετηρία όμως τόσο απόψη ε, διεθνούς δημόσιου δικαίου και συνταγμάτος του Ηνωμένου Βασιλείου απόψη διεθνούς δικαίου είναι ε, ανεξάρτητο κράτος οπότε δεν έχει ε, μια διεθνή σύμβαση επιπτώσει στο, εσωτερικά στο Ηνωμένο Βασίλειο εκτός αν έχει μεταφερθεί η νομοθεσία συνήθως με ε, κοινοβουλευτική πράξη, ε, ενδεχομένως ως δευτερογενής νομοθεσία, όπως θα τις ονόμαζε το Ενωμένο Βασίλειο, τα αντίστοιχο των διαταγμάτων ή ε, κατεξουσιοδότηση πράξεων, όπως τις έχουμε στο Ευρωπαϊκό Νομικό Σύστημα. Αυτή είναι η αφετηρία. Αυτό σχετίζεται με την κοινοβουλευτική κυριαρχία. Η παραδοσιακή θέση του Ηνωμένου Βασιλείου είναι το δικαστήριο δεν μπορεί να αντιστρέψει ε, κοινοβουλευτικέ πράξει αντίθετα με άλλα κράτη όπου τα συντάγματα ε, βρίσκονται ε, είναι ανώτερα από τις κοινοβουλευτικές πράξεις οπότε μπορεί ένα δικαστήριο να απορρίψει κάποια απόφαση του Κοινοβουλίου για την αντισυνταγματικότητά του. Στο Ηνωμένο Βασίλειο δεν υπάρχει τέτοια δυνατότητα. εκτός εφόσον, στον βαθμό που απαιτείται από το ευρωπαϊκό δίκαιο εφόσον το Ηνωμένο Βασίλειο, για όσο χρόνο το Ηνωμένο Βασίλειο είναι μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Αυτή είναι η νομική ε, πτυχή και αυτό ισχύει και για τις διεθνείς συμβάσεις. Δεν έχουν νομικές, ε, νομικά αποτελέσματα στο εγχώριο δίκαιο του Ηνωμένου Βασιλείου χωρίς ε, κοινοβουλευτική πράξη. Το δικαστήριο δεν μπορεί να απορρίψει οι κοινοβουλευτικές πράξεις επειδή αντίκεινται στο διεθνές δίκαιο. Ενώ λοιπόν σε οποιαδήποτε άλλη, οποιαδήποτε χώρα έχει υπογράψει ε, συμφωνίες ε, με το ΕΒ, θα πρέπει να εμπιστευτεί το ΕΒ Βασίλειο ότι μέσω κοινοβουλευτική πράξη ή αλλιώ θα τηρήσει τι διεθνεί του υποχρεώσει και ότι δεν θα υιοθετήσει άλλη κοινοβουλευτική πράξη ε, ή δεν θα διατηρήσει υπάρχουσα κοινοβουλευτική πράξη που έχετε σε αντίθεση με τι διεθνεί του υποχρεώσει. Ω μέλο τη Ευρωπαϊκή Ένωση, φυσικά η θέση του ήταν διαφορετική όσον αφορούσε το ενωσιακό δίκαιο και τα Βρετανικά δικαστήρια τελικά βρήκαν ένα, μια συμφιλίωση μεταξύ της αρχή της κυριαρχίας ε, της υπερίσχυσης ε, του ενωσιακού δίκαιου και των αρχών του Βρετανικού Συντάγματος. Ο συμβιβασμό ήταν ότι τα εθνικά δικαστήρια μπορούσαν να απορρίψουν κοινοβουλευτική πράξη ε, που σχετιζόταν με ευρωπαϊκή νομοθεσία, αλλά για να το κάνουν αυτό χρειαζόταν κοινοβουλευτική πράξη. Αυτό σχετίζεται με την βασική αρχή της κοινοβουλευτικής κυριαρχίας. Αυτή η κοινοβουλευτική πράξη έχει, ε, με τέτοια κοινοβουλευτική πράξη έχει δοθεί η εξουσία στα δικαστήρια να μπορούν να απορρίψουν κοινοβουλευτικές πράξεις. Αλλά τα βρετανικά δικαστήρια έχουν διατηρήσει την άποψη ότι ακόμη και ως μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης μπορούν να δώσουν δικαίωμα στο Κοινοβούλιο να καταργήσει κάποια ευρωπαϊκή νομοθεσία εφόσον το επιθυμεί. Έχουν υπάρξει και άλλες αποφάσεις του Ανωτάτου Δικαστηρίου του Ηνωμένου Βασιλείου πρόσφατα χρόνια που μας κάνουν να πιστεύουμε ότι κάποιες βασικές αρχές του Βρετανικού συντάγματο πέραν τη κοινοβουλευτική αρχής δεν είναι κατώτερες από το ευρωπαϊκό δίκαιο. Οπότε τα Βρετανικά δικαστήρια, όπως πολλά από τα συνταγματικά και ανώτατα δικαστήρια σε άλλες χώρες, δέχονται το ενωσιακό δίκαιο αλλά με τον τρόπο με τον οποίο το έχουν προσαρμόσει στη δική τους παραδοσιακή κυριαρχία στο συνταγματικό τους δίκαιο. Προσπαθούν πάντα να υπάρχει ε, κάποιος συμβιβασμός, αλλά ποτέ δεν έχουν ε, ε, δεχθεί την, το να υπερισχύει το ενωσιακό δίκαιο όπω αυτό ισχύει στι αρχέ τη Ευρωπαϊκή Ένωση. Το ίδιο συμβαίνει και σε άλλε χώρε όπω στη Γερμανία ή στην Δανία. υπάρχουν άλλε εκδοχέ τη υπερίσχυση του ευρωπαϊκού δικαίου. Ε, οπότε ενδεχομένως να υπάρχουν ακόμα διενέξεις ε, σε κάποιες περιπτώσεις. Αυτά όσο το Ηνωμένο Βασίλειο είναι μέλος. Ε, μόλις γίνει το Brexit, το Brexit πρόθεση της Βρετανικής κυβέρνησης είναι να επιστρέψει στις Βρετανικές θέσεις όπου η ισχύς των συμφωνιών των διεθνών συμφωνιών, των συμφωνιών δημοσιο, ε, διεθνούς δημοσίου δικαίου εξαρτάται από τα μέρη. Αυτό δεν ορίζεται στην ίδια τη Διεθνή Συμφωνία. Το Ηνωμένο Βασίλειο ε, επιθυμεί να δεχθεί την διεθνή επίλυση διαφορών, όπως είπε ο καθηγητής Φερνάνδες Τόμας. Υπάρχουν πολλά παραδείγματα ε, ενωσιακών συμφωνιών με κράτη με εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης και αυτές καταδεικνύει το Ηνωμένο Βασίλειο, οπότε αυτή η αρχή του διτού χαρακτήρα θα βάσει αυτή τη αρχή θα δεσμεύεται σε διεθνέ ε, ε, επίπεδο το Ηνωμένο Βασίλειο, αλλά δεν θα δεσμεύονται τα, το Κοινοβούλιο και τα δικαστηριά του. η Βρετανική κυβέρνηση ανησυχεί για το ότι το δικαστήριο θα έχει άμεση δικαιοδοσία στο Ηνωμένο Βασίλειο μετά από τον Brexit και το απορρίπτει αυτό ισχυριζόμενο ότι δίνουμε δικαιοδοσία σε ένα τρίτο μέρος στο δικαστήριο, δικαιοδοσία επί της νομικής τάξης του Ηνωμένου Βασιλείου και πολλά κράτη δεν θα τον δέχονταν αυτό το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο και η νομολογία του για διεθνεί συμβάσει απορρίπτει αυτή την ιδέα όσον αφορά το ενωσιακό δίκαιο. Δεν είναι δυνατόν ε, οργανισμοί που έχουν ε, δημιουργηθεί βάσει διεθνών συμφωνιών να πούν στην Ευρωπαϊκή Ένωση πώ να εφαρμόζεται η Ευρωπαϊκή Νομοθεσία εντό Ευρωπαϊκή Ένωση. Ε, θα το βρούμε δηλαδή αυτή την αρχή, θα τη βρούμε αυτή την αρχή και αλλού. Οπότε δεν είναι τόσο εξωφρενικό ούτε ασυνήθιστο αυτή η θέση που υιοθετεί το όνομα Βασίλειο σε σχέση με άλλες χώρες. Πώς, ε, τι αποτελέσματα θα έχει αυτή η θέση του Ηνωμένου Βασιλείου στις ε, λεπτομέρειες ε, πρώτα απ' όλα του λογαριασμού αποχώρησης του Ηνωμένου Βασιλείου που βρίσκεται στο Κοινοβούλιο ήδη υπό εξέταση και έχουν γίνει διάφορες τροπολογίες πρέπει να περάσει και από τη Βουλή των Λόρδων όπου είναι πολύ πιθανό να ιτηθεί η κυβέρνηση στη θέση της ε, γιατί πρέπει και τα δύο ε, σώματα του Κοινοβουλίου να συμφωνήσουν. Θα χρειαστεί λίγος καιρός για να δούμε τι θα γίνει με αυτό το λογαριασμό αποχώρηση. Ε, αλλά αν δούμε αυτά που προτείνει η κυβέρνηση, το νομοσχέδιο αυτή, αυτό, συγγνώμη, το αποχώρηση, δεν ξέρουμε ακόμα τι θα περιλαμβάνει ακριβώς από άψη περιεχομένου ή όσον αφορά τη δικαιοδοσία ή τις τα νομικά αποτελέσματα της Ευρωπαϊκής Νομοθεσίας. Έχουμε το νομοσχέδιο αποχώρησης του Ηνωμένου Βασιλείου υπό εξέταση και τι συμβαίνει εκεί. Θα διατηρηθεί η Ευρωπαϊκή Νομοθεσία που υιοθετήθηκε μέχρι την ημερομηνία εξόδου, που μπορεί να μην είναι ίδια με την ημερομηνία της εξόδου του Ηνωμένου Βασιλείου, μπορεί να είναι διαφορετικές ημερομηνίες, αλλά όλη η Ευρωπαϊκή Νομοθεσία που έχει υιοθετηθεί ε, πριν από αυτήν την ημερομηνία και δεσμεύει το Ηνωμένο θα συνεχίσει να ισχύει επί της αρχής. Αυτό περιλαμβάνει την ομολογία του δικαστηρίου που έχει υιοθετηθεί μέχρι την ημέρα του Brexit. Στη συνεχεία το, Κοινοβούλιο του Ηνωμένου Βασιλείου ε, ή το εκτελεστικό σώμα ή το ανώτο δικαστήριο θα μπορούν να αλλάξουν την νομοθεσία αυτήν. το Ανώτατο Δικαστήριο δεν υποχρεούται να ακολουθεί αποφάσεις του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου. Και όλα αυτά μπορεί να επηρεαστούν από αποφάσεις του ε, Κοινοβουλίου ή από τους νομοθέτες γενικώ, όπου έχουν εξουσίες. Ε, και μετά στη Σκωτία, στην Ιρλανδία, στη Βόρεια Ιρλανδία και αυτοί θα έχουν την ελευθερία να νομοθετήσουν στους τομείς αρμοδιότητάς τους. Αυτό φυσικά διαφέρει από τη θέση του Ηνωμένου Βασιλείου ως μέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης όπου οποιαδήποτε ε, παράβλεψη αποφάσεων του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου ε, αποτελεί παραβίαση του Ευρωπαϊκού, ε, της Ευρωπαϊκής Δημοθεσίας που δεσμεύει το Ηνωμένο Βασιλείο. Οπότε αφετηρία είναι ότι διατηρείται το ευρωπαϊκό δίκαιο αλλά υπάρχει δυνατότητα να αλλάξει αυτό από πολιτικούς θεσμούς ή από δικαστήρια. Το νομοσχέδιο αποχώρησης λέει επίσης ότι το δικαστήριο του Ηνωμένου Βασιλείου μπορεί να λάβουν υπόψη την ομολογία του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου μέχρι την ημέρα εξόδου προαιρετικά. Είναι προαιρετικό δηλαδή. Μπορούν λοιπόν να νομοθετήσουν βάσει της ε, παραδοσιακής ευελιξίας που υπάρχουν στα Βρετανικά δικαστήρια. Να πούν ότι ας πούμε οι αποφάσεις του των ακόλουθων δικαιοδοσιών μπορεί να είναι ε, συμβουλευτικές και όχι δεσμευτικές, ε, όπως για παράδειγμα με τη ΣΥΠΑ, με τον Καναδά, για θέματα ε, common law ή χωρών όπως η Γερμανία με διαφορετικές παραδόσεις ή οποιασδήποτε συγκλήσεις τις οποίες έχει αναφερθεί το ανατολικό Δικαστήριο για θέματα ανθρώπινων δικαιωμάτων και όσον αφορά το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων όπως και το Δικαστήριο των Ηνωμένων Πολισιών για θέματα ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Υπάρχει πάντα λοιπόν αυτή η ευελιξία που έχει θεσμοθετηθεί ε, κατά τη διακριτική ε, ευχέρεια των Βρετανικών δικαστηριών. Αυτή είναι η θέση του Ηνωμένου Βασιλείου. Σε αντίθεση με αυτήν έχουμε τη θέση της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Δηλαδή αυτά που έχει πει το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο, αυτά που απαιτεί το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο στην ομολογία του. Εγώ την γνωμοδότηση 1.92 του ΕΟΧ και 1.2000 του ε, Ευρωπαϊκού Κοινού Χώρου Αεροπορίας. Όπως το καταλαβαίνω, δεν υπάρχει υποχρέαση επέκτασης της δικαιοδοσίας του Ευρωπαϊκού Δικαστήριου σε χώρα εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης. Δεν υπάρχει τίποτα σε αυτές τις αποφάσεις ε, του ECHR ή του Patent Court που να απαιτεί από χώρες που δεν ανήκουν στην Ευρωπαϊκή Ένωση να ε, τηρούν αποφάσεις του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου. Αυτό που ανησυχεί το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο είναι το να διατηρήσει την αυτονομία της Ευρωπαϊκής Ένωμης Τάξης. Δηλαδή, στα υπόλοιπα κράτη, στα παραμένοντα κράτη της Ευρωπαϊκής Ένωσης και τη σχέση τους με την Ευρωπαϊκή Ένωση ως θεσμικό όργανο και με την νομική τάξη της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Αυτό το ανησυχεί. Αυτό οδηγεί στις ε, ενστάσεις, ερμηνείες ε, του δικαστηρίου ή στα σχέδια διεθνών συμβάσεων για τα οποία καλείται να αποφασίσει. Έχω διαβάσει πολλές φορές τέτοιες αποφάσεις και ουδέποτε βρήκα οτιδήποτε που να απαιτεί από μια χώρα εκτός της Ευρωπαϊκής Ένωσης να δεσμεύεται από τη δικαιοδοσία του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου. Αυτό που έχει πει το δικαστήριο είναι ότι είναι εντάξει το να δίνουμε τη δυνατότητα στα κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης να δέχονται τη δικαιοδοσή του εφόσον το μη κράτος μέλος, εφόσον υιοθετήσουν τη λύση αυτή, θα συμφωνήσουν η απόφαση να είναι δεσμευτική για τα ε, εθνικά δικαστήρια του μη κράτους μέλους. Ε, δεν ε, μπορεί να δεχτεί το δικαστήριο να έχει μη δεσμευτικό ρόλο σε σχέση με τα μη κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Υπάρχει λοιπόν αυτή η λύση. Να πω κάτι ευρύτερο για το ίδιο θέμα. Ε, ως γενικό ρόλο στο ε, διεθνές δίκαιο δεν είναι δυνατόν ε, να θεωρήσουμε ότι η συνθήκη της Ευρωπαϊκής Ένωσης ε, περιέχει κανόνα που να λέει ότι το ΔΕΚ πρέπει να έχει δικαιοδοσία σε μη κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Εάν ερμηνεύει κανείς έτσι τις συνθήκες, αυτό σημαίνει ότι οι συνθήκες μεταξύ των κρατών μελών δεσμεύουν ένα μη κράτος μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Αυτό λοιπόν ε, είναι θεμελιώδες θέμα. Θα ήταν θεμελιώδες πρόβλημα το να πούμε ότι κάποιος ε, που δεν αποτελεί μέρος ε, της ε, συνθήκης να δεσμεύεται από τη συνθήκη. Αυτό νομίζω θα παραβίαζε άλλωστε και το άρθρο 50 της συνθήκες. Ε, όπως επίσης το να πούμε ότι οι αποφάσεις του δικαστηρίου θα πάψουν να ισχύουν για ένα κράτο μέλος ε, που επιλέγει να ε, αποχωρήσει. Η προφανής ερμηνεία λοιπόν του άρθρου 50 είναι ότι εκτός αν υπάρξει συμφωνία για το αντίθετο, το δικαστήριο δεν έχει δικαιοδοσία ε, στο κράτος μέλος που αποχωρεί μετά την ημερομηνία αποχώρησης από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Επιπλέον, η πρώτη από τις αποφάσεις αποφάσεις ε, του δικαστηρίου που ανέφερα, η απόφαση 1 του 92 λέει ότι οι χώρες ΕΖΕΣ μπορούν να εφαρμόσουν ε, τμήμα της ευρωπαϊκής νομοθεσίας ε, χωρίς να χρειαστεί να δεχτούν τη δικαιοδοσία του δικαστηρίου με τον τρόπο που την δέχονται τα κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Μπορεί λοιπόν να υπάρξει αυτή η απόκληση μεταξύ κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης από τη μία, που δεσμεύονται πιο αυστηρά από τον ρόλο του δικαστηρίου, που διασφαλίζει την ε, ένωμη τάξη στην Ευρωπαϊκή Ένωση ε, και να έχουμε από την άλλη τα μη κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης όπου υπάρχει μεγαλύτερη ευελιξία ακόμη και αν εφαρμόζουν μεγάλο τμήμα ε, της νομοθεσίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης όπως οι χώρες ΕΖΕΣ άλλωστε. Έχουμε λοιπόν εδώ μια πιθανή σύγκρουση και να σας περιγράψω περί τίνος πρόκειται και γιατί ήταν δύσκολες οι διαπραγματεύσεις στο θέμα αυτό. Ε, η διαπραγματευτική θέση των 27 κρατών μέλων της Ευρωπαϊκής Ένωσης είναι ότι θα πρέπει να υπάρχει μεταβατική ε, περίοδος ε, και θα πρέπει να ισχύει τότε η δικαιοδοσία. Ωστόσο, υπάρχει η δυσκολία ότι αυτή η θέση διαφέρει από τη θέση το, του Ηνωμένου Βασιλείου που θέλει να αποκοπεί από το δικαστήριο και στην πράξη αποχώρησης να διατηρηθεί η νομολογία ε, του δικαστηρίου μέχρι ε, την ημερομηνία αποχώρησης, να υπάρχει όμως δυνατότητα να εξεταστεί ε, μια απόφαση στα εθνικά δικαστήρια εφόσον εκδοθεί μετά την ημερομηνία αποχώρησης. Και να υπάρχει επίσης η δυνατότητα τροποποίησης νομολογίας του δικαστηρίου πριν την ημερομηνία αποχώρησης και να εφαρμόζονται κάποιοι βασικοί κανόνες της ε, Ένωμης Τάξης Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ε, αναφερόμαστε στον ε, χάρτη των θεμελιωδών δικαιωμάτων, αν και αυτό θα ψηφιστεί σήμερα. Και υπάρχουν διάφοροι τρόποι με, τον οποίο, με, με τους οποίους περιορίζεται ε, ο αντίκτυπος ε, της εθνικής νομοθεσίας. Πώς λοιπόν μπορούμε να συμφιλιώσουμε αυτές τις δύο θέσεις. Από πλευράς του Ηνωμένου Βασιλείου θα δεχτεί ε, την διεθνή επίλυση διαφορών αλλά τα 27 ε, κράτη της Ευρωπαϊκής Ένωσης μπορούν να δεχτούν επίλυση διαφορών μόνο για κάποια θέματα και όχι για θέματα που άπτονται της νομοθεσίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Και από πλευράς του ΔΕΚ, όπως αναφέρεται στις υποθέσεις που σας ανέφερα, το δικαστηρίο ε, πάντα διαφωνεί με την ιδέα ένας διεθνής φορέας να λέει στα, ευρωπαϊκά, στα δικαστήρια των κρατών μελών πώς θα ερμηνεύουν την νομοθεσία της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Εάν λοιπόν υπάρχει παραπομπή στην ευρωπαϊκή νομοθεσία, όπως είναι πολύ πιθανό να υπάρχει σε μια μεταβατική περίοδο και σε σχέση με τα δικαιώματα υπηκών και την ε, οικονομική ρύθμιση, ε, αυτό δεν ε, η Ευρωπαϊκή Ένωση θεωρεί ότι αυτό δεν μπορεί να ρυθμιστεί με μια ε, διεθνή μέθοδο επίλυσης διαφορών, ενώ το ε, Ηνωμένο Βασίλειο υποστηρίζει ότι αυτό θα πρέπει να γίνει έτσι. Υπάρχει λοιπόν η γνωμοδότηση για τον ε, Ευρωπαϊκό Εναέριο Χώρο και το δικαστήριο μπορεί να δεχθεί μη κράτη-μέλη να μην δεσμεύονται από τις αποφάσεις του δικαστηρίου, του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου, εφόσον αυτό δεν επηρεάζει την αυτονομία του να αποφασίζει πώς θα εφαρμόζεται η Ευρωπαϊκή Νομοθεσία εντός της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Και αυτό μπορεί να γίνει είτε με ξεχωριστό δικαστήριο για τα μη κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή να υπάρχουν εναλλακτικές ρυθμίσεις ε, στην Συμφωνία για τις Αερομεταφορές αλλά αυτό να αναμειχθεί με ένα σύστημα επίλυσης διαφορών, τον οποίο να λαμβάνει υπόψη την αυτονομία της ε, νομοθεσίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ε, να περιορίζεται όμως από τον κανόνα στην επίλυση διαφορών, ε, να μην μπορεί να αλλάξει η αυτονομία της Ευρωπαϊκής Νομοθεσίας. Σε περίπτωση λοιπόν που να μην μπορεί να επιληθεί η διαφορά και να χρειαστεί μια πολιτική απόφαση ε, θα σημαίνει αυτό ότι μπορούμε να πλέξουμε διαφορετική λύση από τον ρόλο του δικαστηρίου. Και σίγουρα στον ε, ΕΟΧ το δικαστήριο ήταν διατεθειμένο να δεχτεί κάτι παρόμοιο με την πράξη αποχώρησης ε, του Ηνωμένου Βασιλείου από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Όπου θα πρέπει να λαμβάνεται υπόψη η νομολογία του δικαστηρίου πριν την ημερομηνία ε, της αποχώρησης. Αν λοιπόν κάνουμε κάτι παρόμοιο με το Brexit, αυτό μοιάζει λίγο με αυτό που έχει προτείνει το Ηνωμένο Βασίλειο. Ένα τελικό συμβασμό που μάλλον θα μπορεί να γίνει αποδεκτό από την Ευρωπαϊκή Ένωση και το ΔΕΚ είναι η πράξη αποχώρησης να λέει ότι ε, τα εθνικά δικαστήρια της, ε, του Ηνωμένου Βασιλείου θα πρέπει να λαμβάνουν υπόψη την ομολογία μετά την αποχώρηση του Ηνωμένου Βασιλείου. Ε, το Ηνωμένο Βασίλειο έχει δεχτεί αυτό να γίνει ε, στο αστικό δίκαιο σύμφωνα με τη σύμβαση του Λουγκάνο. Ο κανόνας του Λουγκάνο λέει ότι το Ηνωμένο Βασίλειο θα λαμβάνει υπόψη ε, την ε, νομολογία του Δικαστηρίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης και αυτό έχει γίνει αποδεκτό από το ε, Δικαστήριο Ευρωπαϊκής Ένωσης όσον αφορά τον ΕΟΧ και τον τομέα των αερομεταφορών. Το Ηνωμένο Βασίλειο έχει δεχτεί κάτι τέτοιο στον τομέα του αστικού δικαίου, οπότε είναι πολύ πιθανό να δεχτεί κάτι τέτοιο σε σχέση με την πράξη αποχώρησης, με τη συμφωνία αποχώρησης. Και αυτό μπορεί να θεωρηθεί ότι δεν παραβιάζει την κόκκινη γραμμή ε, της κυβέρνησης του Ηνωμένου Βασιλείου για μη άμεση ε, δικαιοδοσία του Δικαστηρίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Έτσι λοιπόν δεν υπάρχει υποχρέωση ε, παραπομπής στο δικαστήριο σχετικών υποθέσεων, αλλά θα πρέπει να, να λαμβάνονται υπόψη οι αποφάσεις του δικαστηρίου, χωρίς να πρέπει να ακολουθώνται σε κάθε περίπτωση. Και θα πρέπει κατόπιν να ε, υπάρχουν πολιτικές λύσεις αποδεκτές από το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο. Ε, προτείνω λοιπόν ε, έτσι να προχωρήσουμε και έχω ε, μια τελική εκδοχή της μελέτης μου. Ε, θα αναπτύξω περαιτέρω το θέμα αυτό. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Ευχαριστούμε κι εμείς. Σίγουρα θα είναι πολύ χρήσιμο για μας να έχουμε το έγγραφο που λέτε. Η Νταϊάννα James έχει τώρα το λόγο. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ πολύ κυρίες και κύριοι. Ευχαριστώ πολύ για την παρουσίασή σας. Ε, είχαμε και κατά το παρελθόν ανταλλαγή απόψεων. Πολύ θετικό. Τώρα, έχω κάποια ζητήματα που για μένα δεν είναι ξεκάθαρα μετά από αυτά που μας είπατε σήμερα. Από ό,τι αντιλαμβάνομαι, και εντάξει δεν είμαι νομικός δύο χρόνια σπούδασα ε, χωρίς να τελειώσω όμως, αλλά μπορείτε να μας εξηγήσετε η δικαστική αναθεώρηση του Ηνωμένου Βασιλείου πώς θα είναι μπορείτε να μας τη βάλετε σε ένα πλαίσιο και να μας πείτε πού θα είναι τα όρια οι κόκκινες γραμμές και δεύτερον σας άκουσα να λέτε ότι μία μη ευρωπαϊκή χώρα δεν δεσμεύεται από την ευρωπαϊκή δικαιοδοσία. Και νομίζω ότι 5-10 λεπτά είπατε το αντίθετο. Πολλοί Βρετανοί που ζουν σε χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, στη Γαλλία, την Ισπανία, για παράδειγμα, γιατί εκεί είναι οι περισσότεροι, μπορείτε να τους καθησυχάσετε ότι θα μπορούσαν να απευθυνθούν στα γαλλικά ή τα ισπανικά δικαστήρια και δεν θα πρέπει να απευθύνονται στα βρετανικά, ότι θα έχουν αυτή τη δυνατότητα. Ευχαριστούμε. Η Μαρτίν Άντερσον. Ευχαριστώ πολύ και εγώ για τις παρουσιάσεις σας για τις εκθέσεις σας. Ε, περιμένουμε να μας στείλετε ό,τι άλλο έχετε. Για την 213 υπόθεση. προκειμένου να προστατεύονται τα δικαιώματα των Ευρωπαίων πολιτών και πιο συγκεκριμένα για την περίπτωση της Ιρλανδίας γιατί αναφέρεστε στο γεγονός ότι η, αρλική, Ιρλανδική κυβέρνηση σωστά ανησυχεί για το τι θα γίνει. Έχουμε επικεντρωθεί πολύ στα θέματα των συνόρων, των θεσμών, που είναι όλα πάρα πολύ σημαντικά ζητήματα. Αν δούμε όμως το έγγραφο το οποίο διέρευσε από την Επιτροπή στη Βρετανική κυβέρνηση, για τον διάλογο όσον αφορά την Ιρλανδία και τις έξι αρχές. Γνωρίζουμε όλοι σε αυτό το στάδιο ότι οι συμφωνίες της Μεγάλης Παρασκευής είναι ένα έγγραφο το οποίο πέρασε από τον ΟΗΕ και που έχει μεγάλη ισχύ. Για κάποιους εδώ το αγνοήσατε λίγο. Λέτε ότι θα έπρεπε να εμπιστευτούμε τους Βρετανούς, αλλά από πλευρά της Ιρλανδίας είναι δύσκολο να μιλάμε για εμπιστοσύνη στους, ε, στη Βρετανική κυβέρνηση όταν μιλάμε για εφαρμογή συμφωνιών, υλοποίηση συμφωνιών στην Βόρεια Ιρλανδία 20 χρόνια μετά τη συμφωνία της Μεγάλης Παρασκευής ακόμα δυσκολευόμαστε να έχουμε κυβέρνηση και να εφαρμοστούν τέλος πάντων, να υλοποιηθούν αυτές οι συμφωνίες. Στις διαπραγματεύσεις για την συμφωνία της Μεγάλης Παρασκευής αναγκαστήκαμε να παρετεθούμε τα σημεία 2 και 3 του συντάγματός μας που μιλάνε για έξι κομιτείες, για το σύνολο της Ιρλανδίας δηλαδή. Και παραιτηθήκαμε για το πνεύμα της Μεγάλης Παρασκευής προκειμένου να βοηθήσουμε και έτσι υπήρξαν οι διατάξεις αυτές για την ενότητα. Και στις 29 Απριλίου είπαμε ότι αν ενωθεί η χώρα θα εξακολουθούν να ισχύουν οι διάφορες διατάξεις στην Βόρεια Ιρλανδία. Εδώ δεν μπορούμε να πούμε είμαστε Ευρωπαίοι πολίτες που ζούμε σε τρίτη χώρα. Δεν ισχύει αυτό. Εξαιτία τη πράξη του 1998, των συμφωνιών τη Μεγάλη Παρασκευή κλπ. Οπότε στις συνομιλίες μιλάμε για τα σύνορα κλπ. Δεν μιλάμε όμως γι' αυτό, για τα δικαιώματα των ε, πολιτών στη Βόρεια Ιρλανδία και για την δικαιοδοσία και την χάρτα θεμελιωδών δικαιωμάτων που θα έπρεπε να εφαρμόζεται στους πολίτες της ε, Βόρειας Ιρλανδίας. Οπότε εδώ δεν είναι η κατάσταση έτσι ωραία που όλοι κοιτάμε, στρεφόμαστε προς την Βρετανική κυβέρνηση και το θέμα είναι οι με τη Βρετανική κυβέρνηση. Όχι, πρέπει να φροντίσουμε να υπάρχουν και διατάξεις που να προστατεύουν τον κόσμο στη Βόρεια Ιρλανδία, που είναι Ευρωπαίοι πολίτες, Ιρλανδοί, είμαστε όλοι και να διασφαλίσουμε ότι ό,τι αλλάξει, ότι άλλαξε μάλλον με τα άρθρα 2 και 3, δεν πρέπει να μας οδηγήσει σε κακή πίστη. δυνατόν να βλέπουμε το Ηνωμένο Βασίλειο σαν ένα σύνολο χωρίς να λάβουμε υπόψη μας τι λένε οι συμφωνίες της Μεγάλης Παρασκευής και πώς παρετεθήκαμε από τα άρθρα 2 και 3 του συντάγματος προκειμένου να πετύχουμε κάτι που τώρα όμως ε, μας ε, στερείται. Οπότε πρέπει να λάβουμε υπόψη μας τα δικαιώματα και την προστασία των Βόρειο Ιρλανδών. Δεν μπορούμε να πούμε ότι θα είμαστε Ευρωπαίοι πολίτες που ζούμε σε τρίτη χώρα. Δεν γίνεται. Και όταν μιλάτε για ευελιξία και ότι χρειάζονται λύσεις με ευελιξία κλπ. Μην ξεχνάτε ποτέ την Βόρεια Ιρλανδία. Ευχαριστούμε. Αμών Χορανκή. Ευχαριστώ πολύ. Πρώτα απ' όλα ευχαριστώ πολύ τους δύο ειδικού για τις εξηγήσει που μας δώσαν. Πρέπει να ομολογήσω ότι παρόλο που είμαι νομικός, σπούδασα, είναι τόσο περίπλοκη η κατάσταση που με ξεπερνάει. Ειλικρινά και έχω ερωτήσεις που θέλω να τις συνδέσω με την πολιτική διαδικασία. Εγώ καταλαβαίνω ότι έχουμε δύο σημαντικές στιγμές στην όλη διαδικασία. Πριν από το Μάρτιο του 2019 υπάρχει μια συμφωνία αποχώρησης του Ηνωμένου Βασιλείου που θα συνδυαστεί κατά πάσα πιθανότητα με μια μεταβατική συμφωνία. Θα πρόκειται για την ίδια συμφωνία κατά πάσα πιθανότητα. Η αποχώρηση και συγχρόνως οι προϋποθέσεις μετάβασης που θα κρατήσουν 2, 5, δεν ξέρω πόσα χρόνια. Και εδώ έρχεται η πρώτη μου αμφιβολία, γιατί νομίζω ότι δύο ειδικοί μας έδωσαν μια διαφορετική ερμηνεία για την ρύθμιση δικαιοδοσίας κατά το διάστημα αυτό. Από ό,τι κατάλαβα, ο καθηγητής Φερνάντες λέει ότι για την περίοδο αυτή τη μεταβατική η δικαιοδοσία του δικαστηρίου του Λουξεμβούργου ισχύει. Το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο αποφασίζει λοιπόν για τις ερμηνείες των μεταβατικών συμφωνιών που λέει ας πούμε ότι θα παραμείνει στην εσωτερική αγορά με τις τέσσερις ελευθερίες στο Ηνωμένο Βασίλειο και με τις προϋποθέσεις για την ηθαγένεια που καθορίζονται επ' αυτού το αρμόδιο δικαστήριο είναι το Λουξεμβούργο. Αυτή είναι, αν κατάλαβα καλά, η θέση του ειδικού παρόλο που υπάρχουν και άλλες δυνατότητες. Θα ήθελα λοιπόν αυτό οι δύο εμπειρογνώμονες μεταξύ τους να το ξεκαθαρίσουν, γιατί ο άλλος εμπειρογνώμονας μας είπε κάτι διαφορετικό. Το δεύτερο, όταν καταλήγουμε σε νέα συμφωνία για τη σχέση της Ευρωπαϊκής Ένωσης με το Ηνωμένο Βασίλειο μετά τη μεταβατική περίοδο, μετά από 5-2 χρόνια. Σε αυτή τη συμφωνία ο μηχανισμός δικαιοδοσίας είναι αυτός που αντιστοιχεί κανονικά και στον Ευρωπαϊκό Οικονομικό Χώρο. Μπορούν να το συμφωνήσουν οι δύο πλευρές ελεύθερα μεταξύ τους, σωστά. Οπότε ρωτάω. Η επίλυση διαφωνιών ανάμεσα σε επενδυτές και χώρες που στην φωνία θέτα με τον Καναδά διευθετήθηκε και προβλέπει ένα σύστημα ιδιωτικό δι... ετησίας με δημόσιους δικαστές, πιστεύει ο καθηγητής Φερνάντες ότι θα ήταν ο σωστός μηχανισμός για τέτοιες περιπτώσεις. Η συμφωνία με τον Καναδά προβλέπει διαφορετικό μηχανισμό από αυτόν που είχαμε. Και ρωτήθηκε το δικαστήριο του Λουξεμβούργου, από ό,τι θυμάμαι, και στη ΣΕΤΑ λέει ότι υπάρχει ένα νέο σύστημα μηχανισμού επίλυσης ιδιωτικό με δημόσιους όμως ε, δικαστές. Τώρα, η διαβούλευση του Κοινοβουλίου μετά από το πρώτο πρόχειρο της συμφωνίας αυτής. Το Μάρτιο που μας έρχεται πιστεύω ότι θα έχουμε ένα πρώτο σχέδιο. Ας πούμε ότι το, το Κοινοβούλιο απευθύνεται στο Ευρωπαϊκό Δικαστήριο λοιπόν και ρωτάει για αυτά που αναφέρει η συμφωνία, το σχέδιο συμφωνίας. Και ας πούμε ότι δίνει την γνώμη του το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο. Από αυτήν δεσμεύεται η Ευρωπαϊκή Ένωση, σωστά, όπως έγινε όταν ε, ενταχθήκαμε στη Σύμβαση για τα Ανθρώπινα Δικαιώματα. τότε το δικαστήριο είπε κάποια πράγματα και δεν μπόρεσε τελικά να γίνει προσχώρηση αυτή. Οπότε ρωτάω τώρα, αν απευθυνθεί στο δικαστήριο το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και πάρει απάντηση από το δικαστήριο, δεν θα πρέπει να περιμένουμε αυτή την απάντηση του δικαστηρίου για να προχωρήσουμε, αφού αυτή θα είναι δεσμευτική. Ευχαριστώ πολύ, ο κύριος Μόρτεν Μέσερσμιτ. Ευχαριστώ και τους δύο μιλήτες ε, για τις πολύ ενδιαφέρουσες παρουσιάσεις. Και εγώ όπως και ο προλαλής σας ε, ανησυχώ, εδώ είμαι στα δεξιά σας, για το τι θα γίνει ε, μετά ε, και στο ενδιάμεσο ουσιαστικά πριν ολοκληρωθεί η διαδικασία. Θα υπάρξουν κάποιοι τομεί όπου θα χρειαστεί να υπάρχει κοινή νομοθεσία, κοινέ συμφωνίε, κάποιοι κοινοί κανόνε οι οποίοι θα εφαρμόζονται, για παράδειγμα, στην αεροπλοεία. Τα εργασιακά, η διέλευση τη μάχη, πολλά. Οπότε αυτό που φαίνεται ενδιαφέρον είναι πώς αυτά τα δύο ανεξάρτητα αλλά ακόμη συνδεδεμένα καθεστώτα θα εκπληρωθούν στην πράξη, πώς θα το περισσότερο και εκτιμένο σήμερα προκύπτει από αποφάσεις νομολογίας. Αν διαβάσει κανείς τις οδηγίες, ε, δεν δίνεται πλήρης ερμηνεία ε, της ε, νομικής κατάστασης ε, διότι μεγάλο κομμάτι βασίζεται σε αποφάσεις του δικαστηρίου εδώ και 50-60 χρόνια. Κάποια πράγματα επηρεάζουν όλες τις, τους κανονισμούς, τις οδηγίες όσον αφορά την εφαρμογή, τη σωστή εφαρμογή από τα κράτη-μέλη κτλ. Μπορεί να αναμένει κανείς ότι μετά την ενδιάμεση περίοδο οι τομεί αυτή όπου θα υπάρχει κάποιο είδου αναγνωρισμένη νομική βάση συνεργασίας ότι ξαφνικά μετά θα υπάρχουν δύο διαφορετικές ερμηνείες. Για παράδειγμα, αν υπάρχει μια συμφωνία για τα εργασιακά δικαιώματα, μπορεί να δεσμεύεται η Ευρωπαϊκή Ένωση από μια αρχή ε, ότι ο πολίτης ας πούμε έχει δικαίωμα αποζημίωση σε περίπτωση που το κράτος μέλος, ε, το ε, παραλείψει να τον αποζημιώσει με τον ένα ή τον άλλο τρόπο ενώ ας πούμε στο Ηνωμένο Βασίλειο θα ισχύει κάτι άλλο ε, ή για τα τεχνικά ζητήματα, κρίσιμα ζητήματα για την ή ότι μπορεί το δικαστήριο να ορίσει ένα πρότυπο για τις 27 χώρες ε, και που θα ισχύει για τον Ρωμανό Βασίλειο με κάποια Αμερική Συμφωνία και που μετά με την εξέλιξη της νομολογίας ε, από τη συνθήκη του Μάστριχτ και μετά μπορεί να οδηγήσει σε πολύ διαφορετικά νομικά πρότυπα μεταξύ των δύο οντοτήτων. Αυτή είναι η πρώτη μου ερώτηση και μετά εν συντομία τώρα όσον αφορά το νομικό καθεστώς ε, των αποφάσεων των ετοιμιγοριών του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου που από ό,τι κατάλαβα όπως λέτε δεν θα έχουν καμία απολύτως ισχύ στο Ηνωμένο Βασίλειο. Αυτό ισχύει εξίσου και σε αποφάσεις προδικαστικές προδικαστικές αποφάσεις και άλλες αποφάσεις του δικαστηρίου Αναφέρετε τη Δανία, την οποία εκπροσωπώ με περηφάνεια. Πρόσφατα ε, είχαμε μια απόφαση του Ενώτου Δικαστηρίου που καθορίζει τις διαφορές μεταξύ αυτών των δύο εντοτήτων και λέει ότι τα προδικαστικά ερωτήματα δεν έχουν την ίδια νομική ισχύση όπως πραγματικές αποφάσεις ε, του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου. Αυτό προβλέπετε. Πώς βλέπετε τη διαφορά αυτών των δύο ε, ισότιμων αλλά διαφορετικών δικαστικών καθεστώτων. Πώς θεωρείτε ότι θα εξελιχθούν. Ευχαριστώ. Ευχαριστούμε πολύ. Ε, επειδή δεν βλέπω να θέλει να μιλήσει κάποιο άλλος, να κάνω εγώ μια σύντομη ερώτηση. Είπατε ότι το νομοσχέδιο αποχώρηση συζητείται αυτή τη στιγμή στο Κοινοβούλιο και θα πάει και στο Βουλή των Λόρδων και θα δούμε ποια θα είναι η κατάληξη και από ό,τι κατάλαβα σε, με αυτό το νομοσχέδιο θα μεταφερθεί το μεγαλύτερο κομμάτι της ευρωπαϊκής νομοθεσίας ε, στο Εγχωριοδίκαιο. Ταυτόχρονα από πλευράς Ευρωπαϊκή Ένωση ακούμε πολύ καθαρά ότι επειδή δεν υπάρχει χρόνος ε, για διαπραγματεύσει συμφωνίας για τη μεταβατική περίοδο, το μόνο που μπορεί να υπάρξει θα είναι η παράταση ε, του υπάρχοντος κεκτημένου. Πώς θα λειτουργήσει αυτό, υπάρχει κάποιο κίνδυνος ε, σε αυτή την περίπτωση παράτασης του κεκτημένου. και με τη θέση ισχύ του νομοσχεδίου αποχώρησης ε, την ε, ημερομηνία που θα ε, σημάνει την αρχή της μεταβατικής περίοδου. Έχετε το λόγο, όποιος θέλει να μιλήσει πρώτος, παρακαλώ. Η ερώτηση της κυρίας Ζήμης προφανώς είναι για τον κύριο Πίρση. αλλά θα προσπαθήσω να απαντήσω στις άλλες. Γι' αυτό που ρώτησε η κυρία Άντερσον. Πρέπει να σας πω το εξής. Πρώτον, δεν έχω ασχοληθεί τόσο με τα θέματα της Ιρλανδίας. Είναι ένα θέμα για το οποίο θα υπάρξει χωριστή έκθεση. Όμως σας συστήνω να διαβάσετε την εργασία του καθηγητή Μακρούντεν, Μπόριες Ιρλανδίας και στη σελίδα 78 συγκεκριμένα, γιατί λέει κάτι ενδιαφέρον. Ότι πράγματι κατά τη γνώμη του Πρόκειται για διεθνή συμφωνία. Οι συμφωνίες της ε, Μεγάλης Παρασκευής, χωρίς όμως να έχει γίνει ενσωμάτωση στην ε, νομοθεσία. Οπότε δεν μπορεί κανείς να προσφύγει. Χωρίς αμφιβολία πρόκειται για μια πολιτική συμφωνία. Ποια θα είναι η κατάσταση μετά την αποχώρηση. Δεν θα μπορεί κάποιος, είτε πολιτικός, είτε πολίτης, είτε να πάει στα δικαστήρια. Είναι σίγουρα πολύ ενδιαφέρον, εξαρτάται όμως από τα Βρετανικά δικαστήρια. Εγώ νομίζω ότι θα έπρεπε να ενσωματωθεί πρώτα η συμφωνία της Μεγάλης Παρασκευής στο Βρετανικό Δίκαιο και μετά θα μπορούσαν να γίνουν όλα τα υπόλοιπα. Το άλλο που θα κάνω είναι ένα κάπως τολμηρό σχόλιο. Σίγουρα η Ιρλανδία, η Βόρεια Ιρλανδία δεν θέλει να θεωρηθεί αναπόσπαστο κομμάτι του Ηνωμένου Βασιλείου. Ωραία. Τι λύση θα υπήρχε αν ενωνόταν με την λεγόμενη Νότια Ιρλανδία. Να ακολουθήσουμε τη γερμανική λύση. Δηλαδή ένα τμήμα που ήταν ε, Γερμανία ενσωματώθηκε στην υπόλοιπη Γερμανία. Και τότε δεν υπάρχει πρόβλημα με τους πολίτες. Είναι πολιτικά τολμηρή μια τέτοια σκέψη. Αλλά αυτό σκέφτομαι τώρα για αυτά που ρωτήσατε για τη Βόρεια Ιρλανδία. Έρχομαι τώρα στις ερωτήσεις του κύριου Χαουραγκή. Πράγματι, έχουμε να κάνουμε με δύο πολύ βασικά στάδια στην όλη διαδικασία. Αν υπάρξει μεταβατική περίοδος, θα συμπεριληφθεί στη Συμφωνία Απόσυρσης, που θα αποτελείται από ένα στάδιο όπου θα εφαρμόσει τη μεταβατική περίοδος με συγκεκριμένους κανόνες και μετά θα υπάρξει μια άλλη ρύθμιση, γιατί δεν θα ισχύει πια το κοινοτικό δίκαιο. Αν ισχύει το ευρωπαϊκό δίκαιο, εποφελείται από τις τέσσερις ελευθερίες το Ενωμένο Βασίλειο. Παρετείνεται κατά κάποιο τρόπο. Ε, παρατείνονται τα δικαιώματά του. Γι' αυτό λέω ότι υπάρχουν ε, πλεονεκτήματα και μειονεκτήματα. Το μειονέκτημα για το Ηνωμένο Βασίλειο είναι η δικαιοδοσία του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου. Τώρα το πρόβλημα που είναι δύσκολο για τους μη νομικούς να καταλάβουν είναι ότι η δικαιοδοσία αυτή του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου είναι η τελική δικαιοδοσία. Η άμεση, η πρώτη, είναι του Εθνικού Δικαστηρίου. Οπότε αυτό το οποίο θα έπρεπε να διατηρηθεί είναι αυτός ο φάλιος λόρος κατά κάποιο τρόπο που υπάρχει ανάμεσα στα εθνικά δικαστήρια και το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο. Γι' αυτό και μιλάμε για προδικαστικά ερωτήματα, γι' αυτό μιλάμε για ερμηνεία. Πρόκειται για συνεργασία μεταξύ των δικαστών που ερευνούν αν έχουν κάποια αμφιβολία στέλνουν το προδικαστικό τους ερώτημα στο Ευρωπαϊκό Δικαστήριο. Όσον αφορά τώρα τον μηχανισμό διαιτησίας ανάμεσα στους ιδιώτες και το κράτος. Δύο τουλάχιστον από τις διεθνείς συμφωνίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης με τρίτες χώρες, εκείνη της Σιγκαπούρης και εκείνη με τον Καναδά, εκτός από την διαιτησία μεταξύ των δύο πλευρών, Ευρωπαϊκή Ένωση από τη μια και Σιγκαπούρη από την άλλη, Ευρωπαϊκή Ένωση από τη μια και Καναδά από την άλλη. Από την άλλη μεριά υπάρχει και ένα μηχανισμό άμεση επίλυση. Είναι δύο διαφορετικοί μηχανισμοί αυτοί. Και τι γίνεται με αυτόν τον άμεσο μηχανισμό και γιατί λέγεται άμεσος, γιατί ακριβώς παρακάμπτει τις διαδικασίες. Αλλιώς πρέπει να περάσουμε από το εθνικό δίκαιο και να περάσουμε από όλα τα βήματα ενώ αν πάμε κατευθείαν στη διατησία, δεν περνάμε από την τακτική δικαιοδοσία. Οπότε, ποιο είναι το ζήτημα. Είναι ο ιδιώτης ο οποίος μπορεί τελικά να έχει συνδεθεί με τον επενδυτή με κάποιο τρόπο και τελικά οι δικές του οι υποθέσεις σε αυτή την περίπτωση πάνε κατευθείαν για επίλυση σε μια διεθνή δικαιοδοσία. Στον τύπο έχουν ανακοινωθεί κάποια πράγματα, γι' αυτό μπορώ να σας τα πω, αλλιώ η απάντηση, η απόφαση του δικαστηρίου ακόμα δεν έχει δημοσιοποιηθεί. Οπότε το ερώτημα είναι, ο εν λόγω πολίτης έχει πρόσβαση στη δικαιοσύνη. Δεν ξέρω τι θα πει το δικαστήριο. Εγώ λέω πως όχι, δεν θα έχει. Γιατί η υπόθεσή του πάει κατευθείαν σε ένα διαιτητικό σύστημα σε διεθνές επίπεδο. Μηχανισμοί που λειτουργούν όπως η Παγκόσμια Τράπεζα ή άλλοι με μια πρακτική διαιτησίας που συνήθως δικαιώνει τον επενδυτή. Και η Βέλγικη, το βέλγικο ζήτημα που έχει θέσει δηλαδή το Βέλγιο είναι ποιος ορίζει τους υπεύθυνους στη διατησία, πώς πληρώνονται τι υποχρεώσεις έχουν για ενημέρωση, πληροφόρηση κτλ. Θα είναι αρκετά ικανοί οι άνθρωποι αυτοί που θα αναλάβουν τη διατησία όσο είναι ένας δικαστής. Και όσον αφορά το θέμα της διαβούλευσης τώρα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, και αν θα μπορούσε βάσει του 11 να προσφύγει στο ε, δικαστήριο, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και να ζητήσει γνωμοδότησή του. Πρώτον, το Κοινοβούλιο, και όχι μόνο το Κοινοβούλιο, όλα τα ευρωπαϊκά θεσμικά όργανα δεσμεύονται από την όποια απάντηση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Γιατί αυτό που λέμε εμεί γνωμοδότηση του δικαστηρίου, γνώμη του δικαστηρίου, ουσιαστικά είναι κάτι δεσμευτικό. Και τι θα γίνει λοιπόν αν πρώτα γίνει αποχώρηση του Ηνωμένου Βασιλείου και έρθει μετά η απάντηση του δικαστηρίου. Υπάρχουν πολλές περιπτώσεις. Στην περίπτωση του Καναδά προσωρινά εφαρμόζεται όλη η υπόλοιπη συμφωνία, αλλά το κεφάλαιο 8 θα μπορέσει να ισχύσει μόνο αφού έχουμε την απάντηση του δικαστηρίου. Οπότε μπορεί να γίνει εφαρμογή της συμφωνίας αφήνοντας απ' έξω ένα κομμάτι της για το οποίο δεν έχει απαντήσει το δικαστήριο. Τώρα για την ερώτηση του κύριου Μέσσερ Σμιτ. Για τη μεταβατική περίοδο. Αυτό το νομοσχέδιο για την αποχώρηση του Εμένου Βασιλείου που βρίσκεται στο Βρετανικό Κοινοβούλιο, αυτό το νομοσχέδιο προβλέπει τη διατήρηση του παράγωγου δικαίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της δικαιοδοσίας του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου τώρα, μέχρι να αποσυρθεί. Μπορούν να προβλέπονται εξαιρέσεις. Τι εξαιρέσεις βάζει το Ηνωμένο Βασίλειο? Βάζει ότι δεν μπορεί να υπάρξει πρόσβαση στα δικαστήρια βάσει της προηγούμενης απόφασης του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου σχετικά. Οπότε αν περάσει το νομοσχέδιο αυτό, δεν θα μπορεί να ισχύει η δικαιοδοσία του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου. Τώρα, το ανώτατο δικαστήριο της Δανίας. για το κατά πόσο πρόκειται για ερμηνεία ή όχι και τι είναι πάνω από το άλλο. Δεν ξέρω ποια ακριβώς είναι η νομολογία, τι ισχύει ακριβώς ε, στο ανώτατο δικαστήριο της Δανίας και μπορεί να υπάρξει σύγχυση, γιατί οι περισσότεροι εσωτερικοί δικαστές σε μια χώρα δεν έχουν υποχρέωση να υποβάλουν προδικαστικό ερώτημα στο Ευρωπαϊκό Δικαστήριο. Δεν είναι υποχρεωμένοι. Μπορούν να το κάνουν, αλλά δεν είναι υποχρεωμένοι. Αν φτάσει το πράγμα στον νότο το δικαστήριο και δεν μπορεί να αποφανθεί, τότε ναι. Αναφέρθηκαν και κάποια πράγματα για την Ευρωπαϊκή Συμφωνία Αεροπορίας ε, συμφωνίες με την Ουκρανία και την ε, Μολδαβία, η συμφωνία με τον ΕΟΧ. Μπορεί να μην είναι σαφή τα πράγματα, αλλά εδώ ο αξιότιμος καθηγητής Πίρς επίσης αναφέρθηκε σε αυτά. Αλλά τι σημαίνει αυτό η διαιτησία στην περίπτωση της Ουκρανίας και της Μολδαβίας. Σπάνια σε τέτοιες περιπτώσεις πάνε προδικαστικά ερωτήματα στο Ευρωπαϊκό Δικαστήριο για Ερμηνεία. Πρόκειται πάντα για την προσέγγιση των ε, διατάξεων. Είναι ίδιες οι διατάξεις. Είναι. Το θέμα είναι το πώς εφαρμόζονται στη μία και την άλλη χώρα. Η ερμηνεία μπορεί να διαφέρει δηλαδή, όχι η ίδια η ουσία. Τώρα για την ερώτηση της Προέδρου, αν και απευθύνεται μάλλον στον καθηγητή Πύρση. Κατά τη γνώμη μου, εφόσον δεν υπάρχει χρόνος για το περιεχόμενο της συμφωνίας, όντως πιστεύω και εγώ ότι το ευρωπαϊκό κεκτημένο θα παραταθεί. Τέσσερις ελευθερίες, δικαιώματα πολιτών, θέματα αρμοδιότητας κλπ. Ο κύριος Πίρς, ευχαριστώ. Ευχαριστώ για τις ερωτήσεις. Θα προσπαθήσω να απαντήσω σε αυτές μία προς μία. Πρώτα απ' όλα, ο έλεγχος της νομιμότητας μιας αποφάσης του δικαστηρίου στο Ηνωμένο Βασίλειο δεν νομίζω θα λειτουργήσει αυτή η διαδικασία. Αυτό που φανταζόμαι ότι θα συμβεί μετά από την ημέρα του Brexit είναι ότι, για παράδειγμα, μια απόφαση του δικαστηρίου, ας πούμε, για την οδηγία ε, ας πούμε, χρόνο εργασία το Ιούνιο του 2019. Υποθέσουμε ότι έχουμε κάτι τέτοιο. Με το σχέδιο που έχουμε αυτή τη στιγμή, το νομοσχέδιο αποχώρηση δεν υπάρχει καμία υποχρέωση να ληφθεί υπόψη αυτή η απόφαση. Οπότε πιθανότητα αυτό που θα υποθεί θα είναι γιατί να ακούσουμε αυτή την απόφαση γιατί να τεθεί σε ισχύ από τα Βρετανικά δικαστήρια και τα συνδικάτα θα πούνε ότι μάλλον πρέπει να εφαρμοστεί και μετά τα Εθνικά Δικαστήρια του Νομού Βασίλειου θα αποφασίσουν ποιον θεωρούν πιο πιστικό και ποιον θέλουν να λάβουν υπόψη, αν θέλουν να λάβουν υπόψη το δικαστήριο. Αλλά θα έχουν και την επιλογή του νομοσχεδίου αποχώρησης όπου δεν λαμβάνεται υπόψη. Δεύτερον, τι γίνεται με τη δικαιοδοσία του δικαστηρίου, ε, κατά πόσο δηλαδή θα δεσμεύεται το Ηνωμένο Βασίλειο. Είναι περίπλοκο. Να ξαναπώ, να, ε, με άλλη διατύπωση αυτό που είπα, ίσως να είναι σαφέστερο τώρα. Πρώτα απ' όλα, ένα κράτος εκτός Ευρωπαϊκή Ένωση δεν μπορεί να δεσμεύεται να προσυπογράψει ε, στη δικαιοδοσία του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου. Ωστόσο, το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο θα εξακολουθήσει να είναι το δικαστήριο που θα έχει δικαιοδοσία για την υπόλοιπη Ευρωπαϊκή Ένωση όσον αφορά το ενωσιακό δίκαιο. Δεν υπάρχει ε, αντιπαράθεση μεταξύ των δύο, αλλά θα υπάρξει πρόβλημα συμβιβασμού αυτών των δύο θέσεων όταν η συμφωνία αποχώρησης στο μέλλον θα αναφέρεται σε του τη Ευρωπαϊκή Δομοθεσία. Εκεί θα υπάρχει ένα διεθνέ σύστημα επίλυση διαφορών που επί της αρχής δεν δημιουργεί πρόβλημα, αλλά το πρόβλημα είναι όταν αυτό το σύστημα επίλυση διαφορών θα αρχίσει να επιλύει διαφορέ ε, ενωσιακού δικαίου. Διότι το Ηνωμένο Βασίλειο δεν θα έχει πρόβλημα, αλλά η Ευρωπαϊκή Ένωση θα έχει πρόβλημα. Διότι θα λέει ότι αυτό το διεθνέ σύστημα επίλυση διαφορών δεν μπορεί να μα λέει εμά το δικό μα δικαστήριο τι να κάνουμε εμεί ω Ευρωπαϊκή Ένωση. Οπότε θα πρέπει να βρούμε μια λύση και εγώ πρότεινα στις λύσεις που έχει δεχτεί παλιότερα το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο που μοιάζουν με αυτά που λέει ήδη το νομοσχέδιο αποχώρησης. Το άλλο ερώτημα για τους ε, Βρετανούς πολίτες στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Η συμφωνία αποχώρησης θα υπογραφεί μόνο από την Ένωση. Οποιοςδήποτε λοιπόν ζει εντός της υπόλοιπη Ευρωπαϊκής Ένωσης μπορεί να πάει στα εθνικά δικαστήρια για να υπερασπιστεί μια υπόθεση και τα εθνικά δικαστήρια μπορεί να αισθανθούν ε, ότι δεν υπάρχει ανάγκη να απευθυνθούν ε, στο Ευρωπαϊκό Δικαστήριο για να ζητήσουν τι απόψει του. Αλλά αυτό είναι μέτρο τη Ευρωπαϊκή Ένωση. Αν το επιθυμούν όμω, αν το ανώτο δικαστήριο στη Γαλλία, στη Γερμανία ή στην Ισπανία ε, χρειαστεί, μπορεί να πάει να ρωτήσει το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο για την άποψή του. Αλλά δεν θα, δοθεί, δεν θα δοθούν ιδιαίτερε συνθήκε για του Βρετανού πολίτε, αν δεν δίνονται σε άλλου μετά η συμφωνία της Μεγάλης Παρασκευής. Εμπιστεύεστε τους Βρετανούς, αυτό είναι το θέμα. Ε, η έλλειψη εμπιστοσύνη που είχε η Ιρλανδική πλευρά προς τη Βρετανική ήταν ε, το εξή. Γιατί ε, ζητείτε να είναι μέλος η Βρετανία του ECHR και το ζήτημα του πώς θα επιληθεί το ζήτημα της Ιρλανδίας που εξετάζει το ECHR μας λέει ότι το Ηνωμένο Βασίλειο είναι μέλο του ECHR και θα πρέπει να το εφαρμόσει νομικά. Αυτή είναι η βασική ανησυχία. Όλα αυτά είναι ζητήματα εκτό ε, του ευρού τη επειδή εφαρμογή τη ενωσιακή ε, ε, νομοθεσία. και μετά τι γίνεται με το θέμα των τελωνίων και με τα γεωργικά πρότυπα. Όλα αυτά δεν απαιτούν απαραίτητα την αποφάση του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου. Λένε η Βρετανία πάρουμε τη Συμφωνία της Ελβετίας. Εκεί δεν εμπλέκεται το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο. Οι δύο πλευρές μελετώνει μια την άλλη, βλέπει η Ευρωπαϊκή Ένωση τι κάνει η Ελβετία, η Ελβετία βλέπει τι κάνει. Το ίδιο μπορεί να κάνει και το Ηνωμένο Βασίλειο. Όσον αφορά τη διαιτησία, δεν νομίζω ότι έχει να κάνει με συμφωνίε. Η ιδιωτική διαιτησία έχει να κάνει με επενδυτικέ ε, διαφορέ. Πολύ απίθανο λοιπόν να επεκταθεί σε άλλου τομεί ε. και μετά για το, η διαδικασία του άρθρου 218 το δικαστήριο μπορεί να το επιταχύνει ε, το 1994 όταν ο Παγκόσμιος Οργανισμός Εμπορίου ε, να το θέσει σε ισχύ είχε γίνει η ίδια διαδικασία μπορεί το ίδιο να γίνει αν καθυστερεί η, η συμφωνία αποχώρησης αυτό που δεν μπορεί να κάνει είναι δεν μπορεί να εφαρμοστεί αν ισχύει ήδη η, ε, η συμφωνία αποχώρησης. Εφόσον έχει ε, τεθεί σε, ε, δεν είναι πλέον το νόμο Βασίλειο, πρέπει να ξεκινήσει άλλη διαδικασία. Όπως είπε ο συναδελφός μου, καλύτερα να κάνετε ερωτήσεις νωρίς γιατί δεν ξέρουμε τι ακριβώς θα λέει η Συμφωνία Αποχώρησης. Μόλις θα γνωρίζουμε το περιεχόμενό της, τότε θα μπορούμε να ρωτήσουμε κάποια πράγματα στο Ευρωπαϊκό Δικαστήριο για να διευκρινιστούν νομικά ζητήματα τα οποία σχετίζονται με αυτή τη συμφωνία Αποχώρησης. Ευχαριστούμε πολύ. Να ευχαριστήσω και τους δύο καθηγητές που αποσαφήνισαν περισσότερο τις ανησυχίες μας, ε, τις επιφυλάξεις μας, τις σκέψεις μας. Θα θέλαμε να κλείσουμε τώρα αυτή την, ε, αυτό το κομμάτι της συνεδρίασης. Ευχαριστούμε αγαπητοί συνάδελφοι. Περνάμε στο πρώτο σημείο της απογευματινής ημερησίας διάταξης ε, ε, της Επιτροπής μας. Ε, θα κάνουμε την ψηφοφορία. Προετοιμαστείτε παρακαλώ για την ψηφοφορία. Αγαπητοί συνάδελφοι, θα ήθελα να δράξω την ευκαιρία να σας ενημερώσω σχετικά με τις αποφάσεις των συντονιστών. Οι συντονιστές συμφώνησαν η έκθεση για την ε, Συμφωνία Πλαίσιο για τις σχέσεις Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και ε, Κομισιόν ε, θα την αναλάβει ο Στέφαν Κοντζάλης από το ε, ΕΛΚ σχετικά με τον κανόνα, τον, το άρθρο 174 του κανονισμού και αίτημα του Προέδρου Ταγιάννη έχει προταθεί ο Ρίτσαρτ Κόρμπερτ ως εισηγητής. Η γνωμοδότηση για την μακροπροληπτική εποπτεία του χρηματοπιστωτικού συστήματος θα την αναλάβει το και Ντανούτα Χίπνερ, και όσον αφορά την παρακολούθηση της εφαρμογής ε, της νομοθεσίας Ευρωπαϊκής Ένωσης το 2016, προτείνεται να τον αναλάβει το ECR, εισηγητής ο κύριος ε, και όσον αφορά την ομάδα εργασίας ε, της ΑΦΚΟ για τον κανονισμό σχετικά με το άρθρο 50 του κανονισμού, και το αν ε, αυτό μπορεί να βελτιώσει τις ε, ε, περιπτώσεις συναπόφασης και το τελευταίο είχε να κάνει με τη διαφοροποιημένη και à συνεργασία πρόταση του κυρίου Μέσορ Σμιτ. Και συμφωνήθηκε αυτή η πρόταση να εξεταστεί στο πλαίσιο της συνέχειας που θα δοθεί στις εργασίες της ομάδας εργασίας. Αυτές λοιπόν ε, ήταν οι αποφάσεις τις οποίες ελπίζω να εγκρίνετε κι εσείς. Ε, next point on our agenda, which is the voting. Προχωράμε τώρα στο επόμενο θέμα της ημερησίας διάταξης, ψηφοφορία. Ένα θέμα έχουμε. Ε, ένα λεπτό πρέπει να καταλάβουμε πώς δουλεύει τη συσκευή, διότι διαφέρει από τις άλλες. Όπως και να έχει, ε, ε, μία δοκιμαστική ψηφοφορία. Παρακαλώ ψηφίστε δοκιμαστική ψηφοφορία για να δοκιμάσουμε τις συσκευές και τις κάρτες. Να βεβαιωθούμε ότι λειτουργούν σωστά. Ελέγχουμε απλά. One Κάποιος δεν ψήφισε, αλλά εντάξει, δεν πειράζει. Λειτουργούν ε, λοιπόν όλα. <laughs> Εγκρίθηκε η δοκιμαστική ψηφοφορία. Προχωράμε τώρα στον κατάλογο. Πρόταση κανονισμού του ε- Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου που τροποποιεί ε, την πρόταση σχετικά με τη χρηματοδότηση ευρωπαϊκών πολιτικών κομμάτων και ευρωπαϊκών πολιτικών ιδρωμάτων. Ε, τροπολογία 10 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. Τροπολογία 11 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. 12 διαγραφή. 12 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. 15 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. 14 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. Τροπολογία 13 με προφορική ε, τροπολογία. Έχει κάνει αντίρρηση στην προφορική τροπολογία, όχι. Ε, την ψηφίσουμε όπως έχει τροποποιηθεί. Υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. Τροπολογία 16, υπέρ, κατά, αποχές, απορρίπτεται. 17, υπέρ, κατά, αποχές, απορρίπτεται. 18, υπέρ, κατά, Αποχές απορρίπτεται. 21 υπέρ. Κατά αποχές απορρίπτεται. Ε, εγκρίνεται, εγκρίνεται, συγγνώμη. 22 υπέρ. Κατά αποχές απορρίπτεται. Συμβιβαστική α υπέρ. Κατά αποχές ε, εγκρίνεται. Οι 19 και 20 καταπίπτουν. 23 υπέρ. Κατά αποχές απορρίπτεται. 24 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 25 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 26 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 27 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 28 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται τροπολογία 1 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 29 υπέρ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 διαγραφή είναι. Αν ε, εγκριθεί πάμε στην 36. Απορρίφθηκε. Μερικές φορές έχω δίκιο λέει η Πρόεδρος. 35 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. 36 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. 38 υπέρ το πρώτο τμήμα. Ψηφίζουμε μόνο το πρώτο τμήμα υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται. Τροπολογία 3 υπέρ No, I don't have the second part. Well, if there is a first part, then I don't have. I'm sorry. Okay, It comes later on. So amendment 3, first part. No, sorry, amendment three in favor. Τροπολογία 3 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 39 με προφορική τροπολογία. Έχει κανείς αντίρρηση όχι. Ψηφίζουμε υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται. Τροπολογία 37 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 40 το πρώτο τμήμα, το οποίο είναι όμοιο με τμήμα της τροπολογίας 3. Ναι. 40 το πρώτο τμήμα, που είναι όμοιο με ε, τμήμα της ε, τροπολογίας 3, υπέρ. Καταπίπτει λέτε. Μπορεί η γραμματεία να το επιβεβαιώσει αυτό. 40 false. Η τροπολογία 40 καταπίπτει. Uh, I just need confirmation. Amendment 3 was adopted. Η τροπολογία 3 υιοθετήθηκε. Καταπίπτει. Ψηφίσουμε λοιπόν το δεύτερο τμήμα ή το σύνολο της τροπολογίας. Ψηφίσουμε το δεύτερο τμήμα. Υπέρ. Κατά. Νομίζω ότι απορρίπτεται η ηλεκτρονική επαλήθευση, παρακαλώ. Δεύτερο τμήμα της τροπολογίας 40. this. We have one EPP too much. One EPP too much, I am told. Can one EPP to... Yes, it's okay. And the... close the vote. Λήξη της ψηφοφορίας. Εγκρίνεται. 12 υπέρ 10 κατά. Εγκρίνεται. Δεν καταφέρατε να ψηφίσετε. Ναι, αλλά αυτό δεν αλλάζει το αποτέλεσμα. Ό,τι και να ψηφίζατε. Όπως και να έχει, δεν θα άλλαζε το αποτέλεσμα. Καταλαβαίνω τώρα. Τροπολογία 38, το δεύτερο τμήμα. Σωστά, υπέρ, κατά. Αποχές απορρίπτεται. Συμβαστική Β, υπέρ, κατά. Αποχές εγκρίνεται. Τροπολογία 40, κάτι... Ω, πού πάμε τώρα. 51. Ε, 51, υπέρ. Όλες οι προηγούμενες καταπίπτουν επειδή οθετήθηκε η συμβαστική. Τροπολογία 4 λέει ότι... Α, η τροπολογία 4 δεν καταπίπτει. Τροπολογία 4 ψηφίζουμε λοιπόν. Υπάρχει προφορική τροπολογία, έχει κανείς αντίρρηση. Όχι. Ψηφίζουμε την τροπολογία 4 με την προφορική τροπολογία υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. Τροπολογία 50 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. 51 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 52 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. 53 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 54 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 56 σωστά 56 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 57 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται τροπολογία 5 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται τροπολογία 60 με προφορική τροπολογία υπέρ. Έχει κανεί αντίρρηση. Όχι, ωραία, ψηφίζουμε υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται. 61 υπέρ. Κατά αποχές απορρίπτεται. 62 με προφορική τροπολογία. Έχει κανεί αντίρρηση. Όχι, ψηφίζουμε λοιπόν. 62 υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται. 63 υπέρ. Κατά αποχές απορρίπτεται. Τροπολογία 6 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 64 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. Ε, σοσιαλιστές και έλκοι ήταν κατά από ό,τι κατάλαβα. 65 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. Τροπολογία 7 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Τροπολογία 8 με προφορική τροπολογία, αν δεν έχει κανεί αντίρρηση, ψηφίζουμε όπως τροποποιήθηκε υπέρ, κατά αποχές εγκρίνεται. 9 με προφορική τροπολογία, αν δεν έχει κανεί αντίρρηση, ψηφίζουμε όπως τροποποιήθηκε υπέρ, κατά αποχές εγκρίνεται. 66 υπέρ, κατά αποχές εγκρίνεται. Η τελική ψηφοφορία είναι ονομαστική. Άρχεται η ψηφοφορία. Α, συγγνώμη, ένα λάθος έγινε. Ε, διότι δεν, ε, δεν είχε προγραμματιστεί για ονομαστική ψηφοφορία το μηχάνημα. Ονομαστική ψηφοφορία, λοιπόν, άρχεται η ψηφοφορία. Can you close the vote? Yes. Λήξη ψηφοφορίας. 19, 2 κατά, 2 αποχές εγκρίνεται. Και πριν προχωρήσουμε στην τελική ψηφοφορία που είναι απόφαση για την έναρξη διαπραγματεύσεων, θα ήθελα να σας ενημερώσω ότι ε, αυτή η ψηφοφορία θα γίνει με βάση την ε, έκθεση όπως τροποποιήθηκε. Επίσης εδώ απαιτείται απόλυτη πλειοψηφία και ε, αν εγκριθεί αυτό, ο εισηγητής, συνεισηγητής και εσκιώδης θα αποτελούν την διαπραγματευτική ομάδα. Ψηφίζουμε λοιπόν ονομαστική ψηφοφορία, όχι έναρξη της ψηφοφορίας. Πάλι έχουμε μία ψήφο παραπάνω από το ΕΛΚ από ό,τι θα έπρεπε. Κάνουμε ό,τι μπορούμε, τι να κάνουμε. Ναι, το ξέρω, ποτέ δεν είναι υπερβολικά πολλοί οι βουλευτές ε, του ΕΛΚ, αλλά συγγνώμη, ε, ε, συνεχίζει. Ένας πρέπει να αποσύρει την τη ψήφο του λήξη της ψηφοφορίας. Μπορούν να ξεκινήσουν οι διαπραγματεύσεις λοιπόν. Μετά από την Ολομέλεια φυσικά. Ναι, εντάξει, μια λεπτομέρεια είναι τώρα η Ολομέλεια. Σας ευχαριστώ θερμά. Και μπορούμε τώρα να προχωρήσουμε στο σημείο 9. Which is... Ο Κρίστιαν Πρέντα είναι ο εισηγητής μας στο σημείο 9 της ημερής σας διάταξης που είναι η, της έκθεση της Επιτροπής 2015 για την επικουρικότητα και την αναλογικότητα. Πρόκειται για γνωμοδότηση της Επιτροπής μας. Παρακαλώ, όσοι θέλετε να αποχωρήσετε, να αποχωρήσετε ησύχως. I think, Christian, you can just... Νομίζω, λοιπόν, ότι μπορούμε να δώσουμε το λόγο στον εισηγητή, αλλά προηγουμένως ησυχία στην αίθουσα. Αλλιώ, όσο πιο πολύ καθυστερείτε, τόσο πιο πολύ θα αργήσει και η συνεδρίαση για αυτούς που παραμένουν. Ωραία, ο κύριος Πρέντα. Ευχαριστώ. Μου αναθέσατε φέτος να ασχοληθώ με την γνωμοδότηση της Επιτροπής μας προς την Επιτροπή Νομικών Υποθέσεων που είναι και αρμόδια επί της ουσίας, όσον αφορά την ετήσια έκθεση. Έλμαρ, θέλεις κάτι? Λοιπόν, συνεχίζει ο κύριος Πρέντα για την έκθεση Επιτροπής της έκθεσης 2015 για την επικουρικότητα και την αναλογικότητα. Εγκρίθηκε 15 ε, Ιουνίου του 2017. Άργησε λίγο η δημοσίευση, γι' αυτό και τώρα πρέπει να ασχοληθούμε με δύο εκθέσεις, και αυτή του 2015 και του 2016. Υπάρχουν όμως κάποια μειονεκτήματα γι' αυτό. Το γεγονός όμως από την άλλη που εξετάζουμε και τις δύο εκθέσεις και για το 2015 και το 2016 μαζί, έχει και κάποια πλεονεκτήματα. Έτσι μπορούμε να δούμε πιο ξεκάθαρα τις τάσεις που εμφανίζονται όσον αφορά την τήρηση των αρχών της επικουρικότητας και αναλογικότητας, αλλά και το πώς εφαρμόζονται οι ελεγκτικοί μηχανισμοί που έχουν ε, καθοριστεί προς όφελος των Εθνικών Κοινοβουλίων. Με τον τρόπο αυτό, όσον αφορά τις αιτιολογημένες γνώμες που υιοθέτησαν τα Εθνικά Κοινοβούλια βάσει του πρωτοκόλλου αριθμός 2 για την εφαρμογή των αρχών της επικουρικότητας και της αναλογικότητας, Έχουμε ένα περιορισμένο αριθμό τέτοιων γνωμοδοτήσεων για το 2015, 8 μόνο. Διαπιστώσαμε όμως την επόμενη χρονιά, το 2016 δηλαδή, να έχουμε εκθετική αύξησή τους, πάνω από 700% αύξηση. Είχαμε 65 αιτιολογημένες γνώμες το 2016. Ο τρίτος μεγαλύτερος αριθμός που έχουμε από τότε που άρχισε να ισχύει αυτός ο μηχανισμός με τη συνθήκη της Λισαβόνας. Επίσης, στα πλαίσια του πολιτικού διαλόγου, πολύ συχνά στέλνουν ε, γνωμοδοτήσεις στα Εθνικά Κοινοβούλια. 350 είχαμε τέτοιες το 2015 και 620 το 2016. Τώρα βέβαια πρέπει να τεθεί το ερώτημα τι σημαίνει η αύξηση αυτή. Μάλιστα σε ένα πλαίσιο όπου υπήρξε μια γενική πτώση της νομοθετικής δραστηριότητας. Όπως ξέρετε, ο πολιτικός προσανατολισμός της Επιτροπής μας ήταν να ε, συγκεντρώσει την νομοθετική διαδικασία. Η αύξηση αυτή λοιπόν, κατά τη γνώμη μου, δεν δείχνει ότι έχουν αυξηθεί τα προβλήματα σχετικά με την επικουρικότητα. Όχι, απλώς εγώ πιστεύω ότι τα Εθνικά Κοινοβούλια θέλουν να συνεχίσουν να επηρεάζουν την Ευρωπαϊκή Νομοθετική Διαδικασία. Σίγουρα δείχνει ότι ενδιαφέρονται τα Εθνικά Κοινοβούλια όλο και περισσότερο για τις ευρωπαϊκές αποφάσεις και αυτό πρέπει να το χαιρετήσουμε. Αυτό φαίνεται και από την αύξηση των Εθνικών Κοινοβουλίων που υιοθετούν αιτιολογημένες γνώμες. 41 κοινοβούλια, 26 ε, ενέκριναν το 2016 αιτιολογημένες γνώμες, ενώ ήταν 8 τα κοινοβούλια που είχαν κάνει το ίδιο το 2015. Το ίδιο η σε ισχύει και με τον πολιτικό διάλογο. Και νομίζω ότι περισσότερο γι' αυτόν ενδιαφέρονται από ότι για την εφαρμογή τη επικουρικότητα και τη αναλογικότητα. Θέλουν να περάσουν την νομοθετική διαδικασία τα εθνικά κοινοβούλια, αλλά έχουν και όλα μέσα στη διάθεσή του, μέσα από τι κυβερνήσει του, που τα εκπροσωπούν στο Συμβούλιο. Το 2016 επίση είδαμε ότι άρχισε μια τρίτη διαδικασία βάσει το άρθρο 7 του πρωτοκόλου 2 που έχει να κάνει με την αναθεώρηση της οδηγίας για τους αποσπασμένους που είναι ιδιαίτερα επίμαχοι. Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο τελικά φαίνεται ότι αποτελεί ένα πραγματικό συνομιλητή των Εθνικών Κοινοβουλίων γιατί πολλές φορές πήρε αιτιολογημένες γνώμες και άλλη συμβολή στα πλαίσια του πολιτικού διαλόγου. Οπότε εμείς θα πρέπει να καθίσουμε να σκεφτούμε με ποιο τρόπο θέλουμε να βελτιώσουμε ακόμα περισσότερο τις συναλλαγές μας με τα Εθνικά Κοινοβούλια, προκειμένου να αντιμετωπίσουμε την ίδια την ουσία των νομοθετικών ε, προτάσεων. Κάτι το οποίο μπορεί να οδηγήσει σε εξορθολόγηση του τρόπου με τον οποίο γίνεται ο έλεγχος της επικουρικότητας και της αναλογικότητας. Εκ παραλίλου, συζητούμε και την έκθεση του συναδέλφου Πάρολα Ράντζελ ο οποίος συντάσσει έκθεση για τις διατάξεις που έχουν να κάνουν με τη συμβολή των Εθνικών Κοινοβουλίων. Έτσι λοιπόν, σε αυτά τα πλαίσια μπορούμε να βαθύνουμε περισσότερο στο θέμα και να τα βρούμε μεταξύ μας, να συμφωνήσουμε. Διακόπτει ο μιλητής. Προσπαθώ να μην πω πολύ σε αυτό το θέμα που έχει αναλάβει ο Πάολο Ράντσελ, παρόλο που δεν μπορούμε παρά αναφέρουμε κάποια ζητήματα. Ας πούμε την ιδέα να συνεχίσει ο προβληματισμός για την ιδέα της πράσινης κάρτας, για την ευελιξία στον μηχανισμό εγκαιρής προειδοποίησης. Και κάτι άλλο που αναφέρω σε αυτή την πρώτη εκδοχή είναι ότι η υπηκουρικότητα και η αναλογικότητα βρίσκονται στην καρδιά της λήψης αποφάσεων, όπως φάνηκε και από το πρόγραμμα της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και το Better Regulation, την καλύτερη νομοθέτηση. Ε, χρειάστηκε να περιοριστώ και ευχαριστώ την ε, ε, γραμματεία που με βοήθησε, αλλά εδώ θέλω να μιλήσω περισσότερο για τον έλεγχο της επικουρικότητας και της αναλογικότητας στα πλαίσια της καλύτερης νομοθέτησης. Υπάρχει καινοτομία για το ρόλο του ρυθμιστή, για το ρεφίτ, για τις προσπάθειες της Επιτροπής προκειμένου να τηρείται αναλογικότητα και επικουρικότητα. Όλα αυτά είναι στοιχεία τα οποία βελτιώνουν τους μηχανισμούς που έχουμε στη διάθεσή μας για καλύτερο έλεγχο των βασικών αυτών αρχών επικουρικότητας και αναλογικότητας. Τέλος, η γνωμοδότηση αναφέρει δύο άλλα στοιχεία. Τη δημιουργία πριν από λίγο καιρό μιας ε, task force για την επικουρικότητα και την αναλογικότητα και το κάνοντας λιγότερα ε, αλλά πιο αποτελεσματικά. Πιστεύω ότι αυτά θα πρέπει να παίξουν όλο και περισσότερο ρόλο στον προβληματισμό μας για το μέλλον της Ευρώπης. Σας ευχαριστώ πολύ για την προσοχή σας. Ευχαριστούμε πολύ. Να ρωτήσω την ε, κυρία Κλάδια Ταβδιέρες που είναι σκιώδης των σοσιαλιστών. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Αγαπητοί συνάδελφοι, κύριε Σιγητά, ευχαριστώ πολύ Ευχαριστούμε πολύ και για τη δουλειά σας. Είμαι πολύ χαρούμενη που σήμερα στην ΑΦΚΟ έχουμε την ευκαιρία να συζητήσουμε τις δύο ετήσεις εκθέσεις για το 2015-2016 διότι αυτά ήταν τα δύο πρώτα ε, χρόνια της Επιτροπής Γιούνκερ και εκεί μπορούμε να δούμε ε, σε ποιο βαθμό έχουν τηρηθεί αρχές της επικουρικότητας και της αναλογικότητας ως ε, συνεισηγήτρια για τους σοσιαλιστές και τους δημοκράτες στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο θα σας παρουσιάσω τη θέση της δικής μου πολιτικής ομάδας την οποία θα συμπεριλάβουμε στις ε, τροπολογίες μας που θα πρόκειται να υποβάλουμε. Ήθελα να επισημάνω κάποιες σημαντικές πτυχές που έχω εντοπίσει αυτή τη στιγμή στις δύο ευθές εκθέσεις. Πρώτα απ' όλα, όπως και εσείς κύριε Ισηγητά, δεν μπορούμε να παραβλέψουμε τη διαφορά μεταξύ των αιτιολογημένων γνωμοδοτήσεων που έχουν σταλεί στα Εθνικά Κοινοβούλια το 2015 και το 2016. Ε, το 2015 υπήρξαν λιγότερες τέτοιες αιτιολογημένες γνωμοδοτήσεις, 8 για το 2016 τα πράγματα είναι τελείως διαφορετικά, 65 αιτιολογημένες γνωμοδοτήσεις επί 4 μόλις προτάσεων της Κομισιόν. Η πρόταση που προκάλεσε τις περισσότερες αιτιολογημένες γνωμοδοτήσεις ήταν η οδηγία που αναθεωρούσε την οδηγία για την απόσπαση των εργαζομένων που ε, οδήγησε σε 14 αιτιολογημένες ε, γνωμοδοτήσεις και ενεργοποίησε τη διαδικασία κίτρινης κάρτες. Συζητήθηκε εκτενώς στα Εθνικά Κοινοβούλια ε, και στην Επιτροπή Τραν εδώ και στην Κομισιόν και στην Επιτροπή Τραν της οποίας εγώ είμαι μέλος. Αν δείτε πώς επηρεάστηκαν η ενιαία αγορά και ο τομέας των μεταφορών εδώ τίθεται το ζήτημα και θέλω να το πω και εδώ στην ΑΦΚΟ και στη Ρωμανία και στις άλλες ανατολικές ε, χώρες, ε, ε, χώρες της Ανατολικής Ευρώπης, τις πιο περιφερειακές χώρες για το πούμε έτσι, το διακύβευμα είναι πολύ υψηλό. Η οδηγία για την απόσπαση των εργαζομένων είναι εξαιρετικά σημαντική και ιδιαίτερα επίμαχη. Γέννησε ένα τεράστιο χάσμα μεταξύ Ανατολής και Δύσης σε θέματα αρχής και όσον αφορά την εφαρμογή της Ευρωπαϊκής Νομοθεσίας γενικότερα διότι η δεδηλωμένη ε, πρόθεση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής ήταν να βελτιώσει το ρυθμιστικό πλαίσιο για τα 2 εκατομμύρια ε, αποσπασμένων εργαζομένων. Δεν έγινε αυτό και την καλύτερη στιγμή και εξυπηρετεί περιορισμένο αριθμό χωρών, ουσιαστικά τις δυτικές. θα πρέπει να δούμε πώς θα μπορούσαμε να βελτιώσουμε την υλοποίηση των υπαρχόντων κανόνων και να υπάρξουν οι απαραίτητες κυρώσεις σε όσους δεν τις εφαρμόζουν. Δεν εφαρμόζουν. Έχουμε ένα συγκεκριμένο παράδειγμα που επισημαίνεται από την εθνική διαδικασία και χαίρομαι που ενεργοποιήθηκε η κίτρινη κάρτα από ε, τα εθνικά κοινοβούλια 11 κρατών μελών, γεγονός που αποδεικνύει ότι το σύστημα λειτουργεί και ότι τα εθνικά κοινοβούλια κατάφεραν να επισημάνουν τα προβλήματα ε, ε, σε έγκαιρα και να ενεργοποιήσουν τις διατάξεις προβλέπονται από τις συνθήκες. Μετά την ανάλυση αυτών των δύο εκθέσεων, πιστεύω επιπλέον ότι δίνουν περισσότερες προφορίες σε σχέση με την εκθέση που είχαμε το 2014 και αυτό είναι πολύ καλό όσον αφορά την τήρηση αυτών των θεμελιωδών αρχών της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Αυτό εξηγείται και από το γεγονός ότι από το 2015 και μετά η Κομισιόν έχει δημιουργήσει διάφορα μέσα που καθιστούν δυνατό για πολίτες και εθνικά κοινοβούλια να παρεμβαίνουν, να έρχονται σε επαφή με την νομοθετική διαδικασία σε διάφορα, σε επίπεδα στο στην Ευρώπη. Μαζί με το πακέτο Better Regulation αποκτήσαμε μεθόδους αξιολόγησης ε, της αναλογικότητας και της επικουρικότητας ε, βάσει παρατηρητών στην Ευρωπαϊκή Νομοθεσία. Τέτοιες πρωτοβουλίες βοηθούν στη βελτίωση της διαφάνειας σε ευρωπαϊκό επίπεδο για τους πολίτες. Επ' αυτού ήθελα να αναφέρω τις πλατφόρμες δημόσιας διαβούλευσης που δημιουργήθηκαν από την Κομισιόν όπως η REFIT που επιτρέπουν στα Εθνικά Κοινοβούλια να ε, εφαρμόζουν αυτές τις διαδικασίες πιο δραστήρια και που δίνουν τη δυνατότητα στους ε, συνηθισμένους πολίτες, στους όπλους πολίτες να έρχονται σε επαφή με την Κομισιόν όταν θεωρούν ότι έχει υπερβεί των αρμοδιοτήτων της. Ε, εγώ πιστεύω ότι με την εξέλιξη και περαιτέρω ρύθμιση της διαδικασίας θα μπορέσουμε να ακούσουμε πραγματικά αυτό που πιστεύουν οι πολίτες μας και τα τρία θεσμικά όργανα θα πρέπει να συμμετέχουν στη βελτίωση τη νομοθεσία. Και χαίρομαι που ακούω ότι το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και τα Εθνικά Κοινοβούλια θα συμβάλλουν στι εργασίε τη Task Force που αφορά ε, τι αρχέ τη επικουρικότητα και τη αναλογικότητα. Πιστεύω ότι μια τέτοια πρωτοβουλία θα διασφαλίσει καλύτερη συμμετοχή των τοπικών και περιφερειακών αρχών στην εξέλιξη των ευρωπαϊκών δημόσιων πολιτικών και ότι θα διασφαλίσει ότι αυτές οι πολιτικές οι πολιτικές που ε, πραγματοποιούνται καλύτερα σε εθνικό επίπεδο θα επισημανθούν σωστά. Θέλουμε η Κομισιόν να μας δώσει περισσότερες πληροφορίες ε, για τις αρμοδιότητες αυτής της ομάδας και το modus operandi που προβλέπετε. Αυτά ε, ευχαριστούμε για την προσοχή σας και όπως είπα νωρίτερα η πολιτική μας ομάδα θα υποβάλει διάφορες τρόπολογίες. Ευχαριστώ πολύ. Σας ευχαριστώ πολύ. Το ECR. Ο κύριος Καζημιάς Μιχάλης Ζετόφσκι. Ευχαριστώ πολύ. Θα σας μιλήσω εν συντομία. Σας ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστούμε πολύ ε, κύριε Ντεπρέδα για την εκθεσία αυτή, κύριε Νταμπρέδα ε, και σας ε, διαβεβαιώ ότι τα Εθνικά Κοινοβούλια ενδιαφέρονται περισσότερο για έναν πολιτικό διάλογο παρά για την εφαρμογή των αιτιολογημένων γνωμοδοτήσεων. αλλά δεν είναι ελεύθερη τους επιλογή εάν η διαδικασία της κίτρινης κάρτας δεν ε, πρόκειται να λάβει χώρα υπήρχε περίπτωση να έχει εφαρμοστεί με τρόπο πιο εκτενή από ό,τι γνωρίζουμε τώρα. δεν έχει νόημα για δεύτερη φορά. Ε, είναι μια διαδικασία που ήδη εφαρμόστηκε μία φορά. Σε αυτή τη νέα μορφή της οδηγίας για τους ε, αποσπασμένους εργαζομένους ε, έχουμε μία δεύτερη ε, περίπτωση με πολλές ε, ενστάσεις από πολλά κοινοβούλια και εκεί η Κομισιόν δεν άλλαξε τη θέση της ε, ή αν την άλλαξε την έχει άλλαξει ελάχιστα. Αυτό δυστυχώς δεν αποτελεί υπόδειγμα εμπιστοσύνης ούτε σωστής νοοτροπίας θεσμικής. Αυτός ο μηχανισμός θα συνεχίσει να υπάρχει και θα είναι υποφελής για όλους μας εφόσον εφαρμόζεται σοβαρά από την Κομισιόν. Αυτή την παρατήρηση είχα να κάνω. Έχουμε όλες αυτές τις τροπολογίες ε, που καθιστούν αυτό το σύστημα ε, προειδοποίησης ε, ευέλικτο. Ήθελα να κάνω μια ερώτηση. Ο κύριος Πράγκελ ανήκει στην ίδια, στον ίδιο πολιτικό σχηματισμό. Συνιστώ λοιπόν να λάβετε υπόψη τη συνοχή αυτής της ε, ε, γνωμοδότησης. Σας προτείνω να παρουσιάσετε και την έκθεση ενίσχυσης των Εθνικών Κοινοβουλίων δυνάμει της Συνθήκης Λισαβόνας, γιατί αυτά είναι θέματα ε, αλληλένδετα. Και καλό θα ήταν η ΑΦΚΟ να υποστηρίξει μια πιο δυνατή θέση των Εθνικών Κοινοβουλίων από ότι αυτή τη στιγμή αυτό θα είναι επωφελές και για την Ευρωπαϊκή Ένωση και για την καλή λειτουργία των ε, θεσμικών οργάνων. Ευχαριστούμε πολύ. Ο κ. Τσάρλ Γκέρεντς, όχι. Για την ΚΟΕ e δεν είναι κανένας. Από τους Πρασίνους, ο Μαξ Άντερσον. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Ευχαριστώ τον εισηγητή για τη δουλειά που έχει κάνει πάνω στο θέμα αυτό. Θα ήθελα να ζητήσω συγγνώμη που δεν ήμουν εδώ κατά την παρουσίασή του. Διότι συμμετείχα στη συζήτηση για την έκθεση ε, αυτή στην Γιούρη, που πραγματοποιήθηκε ακριβώς την ίδια ώρα. Θα παρακολουθήσω όμως εκ των υστέρων ε, την ε, μαγνητοσκοπημένη παρουσίασή του. Πάντως προσλέπω στις εργασίες πάνω στο θέμα αυτό. Δεν έχω πιστεί ακόμα ότι όλα τα εθνικά κοινοβούλια της Ευρωπαϊκής Ένωσης παίρνουν αρκετά σοβαρά το θέμα της επικουρικότητας. Πολλά από τα κοινοβούλια δεν έχουν στείλει ούτε μία περιστατωμένη γνωμοδότηση φέτος και νομίζω ότι ένας λόγος που δεν παίρνει το θέμα αυτό στα σοβαρά είναι ότι το σύστημα δεν λειτουργεί τόσο καλό όσο θα έπρεπε. Νομίζω ότι μακροπρόθεσμα θα πρέπει να εξετάσουμε προσεκτικά το κατόφλι. Μήπως είναι υπερβολικά υψηλό και αποθαρρύνει πολύ κόσμο να ασχοληθεί με το θέμα. Διότι είναι τόσο εύκολο να φτάσει κανείς στο κατόφλι. Θα πρέπει λοιπόν να σκεφτούμε πώς μπορούμε στο παρόν πλαίσιο να δώσουμε κίνητρα στα εθνικά κοινοβούλια ώστε να κάνουν σωστά τους ελέγχους επικουρικότητας και αναλογικότητας. Και ένας τρόπος να το πετύχουμε αυτό είναι να φροντίσουμε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή και εμείς να πάρουμε στο σοβαρά το θέμα αυτό. Προσβλέπω στη συνέχιση των εργασιών σας. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ θερμά, Μαξ. Ούτε και ο Φάβιο είναι παρόν. Ο Έλμαρ Μπροκ, παρακαλώ. Ευχαριστώ πολύ, κυρία Πρόεδρε. Ευχαριστώ πολύ, Κριστιαν Πρέντα. Ε, πολλά μου θύμισε με την έκθεση αυτή και θα ήθελα να κάνω κάποιες παρατηρήσεις, διότι Ήμουνα συντάχτης του άρθρου αυτού στην ε, συνταγματική συνέλευση. Δεν ε, αναφέρθηκε σήμερα η πορτοκαλί κάρτα. Ε, είναι όμως μια πρόταση που υποβάλαμε μαζί με τις κάτω χώρες για να ξεπεράσουν το αρνητικό αποτέλεσμα του δημοψηφίσματος. θα πρέπει καταρχάς ε, να γίνει η διάκριση ανάμεσα στην επικουρικότητα και την αναλογικότητα. Παρακαλώ, κοιτάξτε και το πρωτόκολλο. Ε, πολύ, έγινε πολύ συνειδητά αυτή η διάκριση ήδη τότε. Δεύτερη παρατήρηση, τι ακριβώς είναι η επικουρικότητα. Θα πρέπει να εξετάζονται οι προτάσεις, ε, αλλά άλλο το να μην αρέσει σε κάποιον ε, μια νομοθετική πρόταση και άλλο το να μην ε, πληρεί την αρχή της επικουρικότητας. Μπορεί λοιπόν να υπάρχουν και διαφορετικές απόψεις για το θέμα αυτό. Μπορεί να υπάρχουν καλές ή κακές ή λάθος αποφάσεις. αλλά Άλλο η επικουρικότητα, άλλο το αν συμφωνεί κανεί με το θέμα της ε, άλλο με το αν πληρείται η αρχή της επικουρικότητα, ή όχι. Αν ε, λέμε ότι δεν μας αρέσει, ότι δεν πληρεί την επικουρικότητα, αυτό θα σημαίνει ότι θα ακολουθήσουμε λάθος κατεύθυνση. Νομίζω λοιπόν ότι θα πρέπει να εξετάσουμε το περιεχόμενο του θέματος αυτού. Και όσον αφορά την πορτοκαλή κάρτα που εισάγαμε με την παράγραφο αυτήν, άρθρο 7, παράγραφος 3 δηλαδή. Άρθρο 7, παράγραφος 3. Εάν πλειοψηφία των Εθνικών Κοινοβουλίων πιστεύει ότι παραβιάζεται η αρχή ε, της επικουρικότητας, τότε μπορούν, χωρίς να το εμποδίσει αυτό η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, ε, το Συμβούλιο ή το Κοινοβούλιο να ε, δώσουν τέλος στη διαδικασία. Και αν πλειοψηφία των Εθνικών Κοινοβουλίων πει ότι αυτό αποτελεί παραβίαση της αρχής της επικουρικότητας, τότε το Συμβούλιο οι κυβερνήσεις μπορούν να δώσουν τέλος στη διαδικασία. Ε, αρκεί ένας να θέσει το θέμα. Και τον Φεβρουάριο του 2015, ε, ε, όταν ε, συνήθη η συμφωνία με το Ηνωμένο Βασίλειο, το Κοινοβούλιο είπε ότι σε τέτοια περίπτωση θα δώσει τέλος νομοθετική διαδικασία. Ε, με εφαρμογή δηλαδή της παραγράφου 3. Αυτό σημαίνει ότι δεν χρειαζόμαστε την πράσινη κάρτα. Η πράσινη κάρτα είναι μια αυτόματη διαδικασία. όπου δεν γίνεται διάκριση ανάμεσα στο αν υπάρχει παραβίαση της αρχής επικορικότητας ή αν δεν αρέσει σε κάποιον το περιεχόμενο. Έχουμε λοιπόν την πορτοκαλί κάρτα η οποία ακόμη δεν έχει χρησιμοποιηθεί. Θα έλεγα λοιπόν να βελτιώσουμε τις συνθήκες εργασίας για τα εθνικά κοινοβούλια, ώστε να μπορέσουν να χρησιμοποιούν την πορτοκαλί κάρτα. Εμένα αυτό μου φαίνεται λογική μέθοδος. Και στο σημείο 6 της έκθεσης του Κρίστιαν Πρέντα, νομίζω ότι θα πρέπει ε, να αναπτύξουμε πολύ περισσότερο την πρόταση αυτή. Το θέμα των 8 εβδομάδων είναι πρόβλημα το ότι είναι δηλαδή τόσο σύντομη η προθεσμία. Θα πρέπει να βρούμε τρόπους ώστε στην πράξη ε, να παραταθεί η προθεσμία. Να αρχίσει να μετράει ο χρόνος, για παράδειγμα, ε, τη στιγμή που θα υποβληθεί στην επίσημη γλώσσα του κράτους η πρόταση. Θα πρέπει να υπάρχει πρόταση σε κάθε επίσημη γλώσσα, ώστε τα εθνικά κοινοβούλια να μπορούν να εργαστούν πάνω στην πρόταση, να εξετάσουν την πρόταση και αυτό απαιτεί κατόπιν καμιά δύο εβδομάδες παραπάνω. Κάποια τέτοια θέματα να εξετάσουμε. Πώς μπορούμε δηλαδή να παρατείνουμε την προθεσμία των 8 εβδομάδων. ώστε να καταλήξουμε σε διάστημα 10 ή 12 εβδομάδων, ώστε να διευκολύνουμε τα εθνικά κοινοβούλια. Νομίζω επίσης ότι θα πρέπει να προσέξουμε το θέμα της αρχής της επικουρικότητας. Η αρχή της επικουρικότητας ε, έχει υποβληθεί σε διάφορες ερμηνείες. Εκπρόσωπος μεγάλης χώρας ε, θεωρεί ότι παραβιάζεται η αρχή της επικουρικότητα σε ένα θέμα που μπορεί να λύσει μόνο του, ενώ ένα μικρό κράτος δεν μπορεί να το λύσει αυτό μόνο του. Το ίδιο ισχύει ανάμεσα στις πλούσιε και τις φτωχέ χώρες. Υπάρχουν δηλαδή και διάφορες συμπεριφορέ ανάλογα με την καταγωγή κάποιου. Και νομίζω ότι και αυτό θα πρέπει να εξεταστεί. Κυρία Πρόεδρε, θα πρέπει να εξετάσουμε και το θέμα της βελτίωσης της νομοθεσίας. Υπάρχουν ε, κάποια, θέματα που πρέπει να, κάποια πράγματα που πρέπει να κάνουμε που δεν σχετίζονται με την αρχή της επικουρικότητας. Ε, για παράδειγμα, μελέτες αντικτύπου. για να πετύχουμε καλύτερη νομοθεσία. Αυτό δεν σχετίζεται με την αρχή της επικουρικότητας. Όλα αυτά λοιπόν χάνονται Μπερδεύονται όλα αυτά ε, ε, στην ίδια συζήτηση. Και κυρία Πρόεδρε, δεν ξέρω πώς έχει το χρονοδιάγραμμα. Ε, μήπως μπορεί ο κύριος Πρέντα να μας πει κάτι για το θέμα αυτό. Εγώ πάντως σε, αυτή τη φάση βρίσκω πάρα πολύ σημαντικό να έχουμε περισσότερο χρόνο και να καλέσουμε νομικούς εμπειρογνώμονες ώστε με βάση τις προτάσεις του κυρίου Πρέντα να έχουμε διάλογο ώστε να καταλήξουμε σε μια καλή πρόταση. Αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό διότι το θέμα αυτό είναι θέμα κλειδί. Και έχει να κάνει με το αν είμαστε ικανοποιημένοι με τις εργασίες μας, αν έχουμε ένα αξιόπιστο εργαλείο. Και ίσως θα μπορούσαμε να εξετάσουμε αν είναι δυνατόν να βρούμε μια βασική διαδικασία για τα θέματα αυτά και νομίζω ότι η πρόταση του Κρίστιαν Πρέντα αποτελεί πολύ καλή βάση να το πετύχουμε αυτό. Σας ευχαριστώ. Ευχαριστώ, Έλμερ. Να σας υπενθυμίσω ότι μιλάμε για την γνωμοδότηση. Έχουμε και την εκτίμηση Λοράντζο και την έκθεση βελτίωση της νομοθεσίας του Ρίτσαρτ Κόρμπετ ε, από τη Γιούρη, οπότε θα έχουμε περιθώριο για σχόλια. Ε, αυτά που μας είπε, Σέλμερ θα μπορούσαν να το τροφοδοτήσουν πολλά πράγματα, όχι μόνο τη γνωμοδότηση εδώ του Κρίστιαν. Μερσέδες Μπρέσο, έχετε το λόγο. Ναι, απλά λέω, ε, λέει η πρόεδρος, ότι δεν μπορεί να μπει σε τόσο λεπτομέρειε ε, σε τόσο ευρύ πεδίο όσο αυτό που θα θέλατε εσεί αυτό λέω. Ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε. Ήθελα να κάνω μία πρόταση στο συναδελφό μας τον κύριο Νταμπρέντα, ο οποίος ίσως να μην άκουσε τον καθηγητή Μαντούρο που σήμερα εδώ μας μίλησε για το ζήτημα της πράσινης κάρτας. Νομίζω ότι αυτός ήταν παρουσίασε ένα υποθετικό σενάριο της πράσινης κάρτας που αυτή τη στιγμή δεν θεσμοθετείται από τις συνθήκες. Να παρουσιάσει λοιπόν την πράσινη κάρτα ως ένα είδος ε, αντίστροφη αρχή της επικουρικότητας. Δηλαδή ότι κάποιο κοινοβούλιο ή κάποια ομάδα εθνικών κοινοβουλίων θα μπορούσαν να θέσουν στην Κομισιόν ε, το ερώτημα Ε, ότι κάποιο θέμα δεν το έχει αναλάβει η Κομισιόν ενώ θα έπρεπε βάσει τη αρχής της επικουρικότητας. Δηλαδή ότι είναι θέμα ευρωπαϊκής κλίμακας. Γιατί λοιπόν να μην χρησιμοποιείται η αρχή επικουρικότητας αντίστροφα για να επισημαθεί κάποιο ζήτημα που θεωρούν τα εθνικά κοινοβούλια ότι είναι προτιμότερο να εξεταστεί από τα θεσμικά οργάνα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, το Κοινοβούλιο, την Κομισιόν και το Συμβούλιο. Αυτό θα ήταν ενδιαφέρον αναμένοντας αυτή την ε, ε, περίφημη αναθεώρηση των συνθήκων που ακόμα συζητάμε να χρησιμοποιηθεί μια τέτοια διατύπωση ενδεχομένως που μπορεί να ακούγεται περίεργη αλλά ε, έχει κάποιο ενδιαφέρον. και κάποια άλλη τώρα σκέψη για το ζήτημα της κίτρινης και της πορτοκαλί Πιστεύω πράγματι ότι όπως λειτουργούν τα πράγματα τώρα δεν έχουμε καλά αποτελέσματα και ότι αυτό σχετίζεται κατά βάση με το γεγονό ότι η αναλογικότητα μπορεί να παραβιαστεί περισσότερο από οτιδήποτε άλλο. Καλό θα ήταν λοιπόν η Κομισιόν να κάνει μια πρόταση εντελώ εκτό των συνθήκων των εξουσιών τη. Ε, υπάρχει λοιπόν, όμως περίπτωση η έκταση που λαμβάνει μια οδηγία μετά από συζητήσεις ε, στο Συμβούλιο και στο Κοινοβούλιο να καταλήξει να παραβιάζει τις αρχές της αναλογικότητας, όχι απαραίτητα της επικουρικότητας. Και εκεί χρειάζομαστε κάποια βελτίωση πιστεύω, διότι μερικές φορές ε, και εμείς εδώ όταν αρχίζουμε να ασχολούμαστε με ένα ζήτημα πάντα ζητάμε κάτι παραπάνω και όλα να αυξάνουμε την ποσότητα περιεχομένου των κανονισμών και το μέγεθος των κανονισμών. Οπότε θα πρέπει να δούμε κατά πόσο δεχομένω τα Εθνικά Κοινοβούλια και τα Περιφερειακά Κοινοβούλια μέσω της ε, Επιτροπής των Περιφερειών μήπως θα μπορούσαν όλα αυτά οι φορείς να, να θέτουν το ζήτημα αυτό στις περιπτώσεις όπου το νομοθετικό κείμενο ε, έχει ήδη προχωρήσει. διότι η αρχή της αναλογικότητας ε, μπορεί να παραβιαστεί συνήθως προς το τέλος διαδικασίας, όχι στην αρχή, όταν έχουμε προσθέσει κάπως παραπάνω κείμενο από ό,τι επιτρεπόταν. Αυτό το ερώτημα θα μπορούσαμε να θέσουμε. Το θέμα της μελέτης αντικτύπου. Στη Διοργανική Συμφωνία έχουμε προβλέψει επαλήθευση του αντικτύπου στο τέλος ε, της νομοθετικής διαδικασίας με ενημέρωση του Κοινοβουλίου. Ε, εκεί μπορεί να διαπιστωθεί κάτι. Διότι και από τη δική μου εμπειρία ως ε, τοπική ε, πολιτικός ερετή στις λεπτομέρειες παρατηρείται η υπέρβαση της επικουρικότητας. Δεν είναι ο τομέας αλλά μερικές φορές οι υπερβολικές λεπτομέρειες ε, συνιστούν παραβίαση και υπερβαίνουν τις νομοθετικές ε, εξουσίες ε, και καταπατούν τις εξουσίες των τοπικών ή των περιφερειακών κοινοβουλίων. Εκεί θα πρέπει να δούμε κάποιο είδου νομοθετική αναθεώρηση ενδεχομένω. Κριστίαν, θέλετε να απαντήσετε ένα λεπτό. Ναι, κοιτάξτε. Να ευχαριστήσω όλους τους συναδέλφους που ε, συμμετείχαν στη συζήτηση. Είναι πολύ ενδιαφέρουσες οι προτάσεις. Εμείς ε, θα μελετήσουμε τις, ε, και θα εκπονήσουμε τροπολογίες, λαμβάνοντας υπόψη, ελπίζω, τις παρατηρήσεις σας και εντάσσοντες στις τροπολογίες. Τώρα όσον αφορά το χρονοδιάγραμμα, γιατί το ρώτησε ο Έλμαρ Μπρόκ, Σήμερα, ήταν η ε, Σήμερα έχουμε ως προθεσμία υποβολής τροπολογιών τη 15η Δεκεμβρίου. Ένα μήνα. Ε, λίγο λιγότερο. Και μετά οι τροπολογίες ε, λογικά θα είναι διαθέσιμες 10 Ιανουαρίου. Δηλαδή κατά τη διάρκεια των Χριστουγεννιάτικων διακοπών θα γίνει μετάφραση των τροπολογιών. Πιστεύω ότι εντάξει είναι. Ε, άνε το χρονοδιάγραμμα, όχι. Έλμαρ, πώς το βλέπετε, θέλετε περισσότερο χρόνο, γιατί 15 Δεκεμβρίου έχουμε την προθεσμία υποβολή τροπολογιών. Είναι αρκετό ο χρόνος, όχι. Εντάξει, δεν είναι. Επίσης, όπως υπόθηκε, θα επανέλθουμε. 15 Δεκεμβρίου είναι εντάξει. Θα ήθελα όμως να συζητήσουμε και με την Επιτροπή Νομικών Υποθέσεων να, μέσω μιας ακρόασης να λάβουμε κάποιες ε, ε, απόψεις, κάποια συμβουλή μαζί με τις νομικές υποθέσεις γιατί θεωρώ ότι είναι τόσο ύψης της σημασίας το ζήτημα αυτό. Δεν ξέρω, δεν είμαι μέλο τη Τζούρι. Ναι, να μιλήσουμε με τον πρόεδρο τη Επιτροπή Νομικών Υποθέσεων. Μπορεί να γνωρίζουν. Ή με κάποιον μπορεί να γνωρίζει το θέμα. Πρόεδρο, ναι, έχετε τελειώσει. Ναι, πράγματι. Ε, είναι αρκετό ο χρόνος για τι τροπολογίε όταν λέτε 15 Δεκεμβρίου. Επίση ξέρουμε ότι στην Τζούρι θα ψηφίσουν, ε, Γιούρι θα ψηφίσουν το Μάρτιο, οπότε έχουμε χρόνο, υπάρχει ευελιξία. Οπότε α κάνουμε τι τροπολογίε και μετά θα δούμε πόσο χρόνο θα χρειαστείτε. Ε, είστε πολύ ενθουσιώδει αυτή τη στιγμή, αλλά ίσω αργότερα να μην έχει τόσο πολλέ τροπολογίε, οπότε θα αφήσουμε κάποια ευελιξία. Μπορούμε να ψηφίσουμε και τέλη Φεβρουαρίου στην Επιτροπή μα. οπότε κύριε Μπρόκ. Κύριε Χιούμπνερ, δεν είναι δυνατόν το, το τρίτη φορά μαζί με την Επιτροπή Νομικών Υποθέσεων να κάνουμε μια ακρόαση επί του θέματος προσκαλώντας εμπειρογνώμονες. Ε, η ψηφοφορία είναι το Μάρτιο μόλις. Έχουμε χρόνο. Γνωρίζω τον πρόεδρο. Αυτό δεν σημαίνει τίποτα. Οι γραμματείε είναι πιο σημαντικέ δεν ξέρω κατά πόσο αυτό είναι εφικτό, γιατί ήδη έχουμε προγραμματίσει ακροάσεις για το πρώτο εξάμεινο του έτους, εδώ και καιρό. Ίσως υπό κάποια άλλη μορφή, κάποιο workshop ή κάτι τέτοιο. Δεν με ενδιαφέρει, λέει ο Μπρόκ. Ναι, ό,τι να είναι. Πρόεδρος, ναι, δεν θα μπορούσαμε να το εξετάσουμε κατά πόσο είναι δυνατόν. Να μιλήσουμε με την Γιούρη, να δούμε αν είναι διατεθειμένη. Κύριε Μπρόκ, δεν με ενδιαφέρει τι μορφή θα έχει η συνάντηση αυτή. But these experts. No, but Τους υπερογνώμονες δεν μπορούμε να τους πληρώσουμε. Πρέπει να έχουμε τοπικούς που δεν χρειάζεται να τους ε, πληρώσουμε. Η γραμματεία θα ελέγξει τι είναι εφικτό. Πάντως αυτοί που θέλετε να υποβάλλετε τροπολογίες να ξέρετε 15 Δεκεμβρίου είναι η προθεσμία. Στο μεταξύ εμείς θα... Τα δούμε αν έχουμε τη δυνατότητα να ακούσουμε και εμπειρογνώμονες. Ωραία. Καλώς. Περνάμε τώρα στην έκθεση Ραμών Χαουρέγγι. Πρόκειται για πρώτο κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου για την άσκηση του δικαιώματο εξέταση των πραγμάτων από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, προκειμένου να αντικατασταθεί η απόφαση 95-167. Είναι ένα αρκετά δύσκολο διαδικαστικά ζήτημα και ο Ραμόν θα μα εισαγάγει στο θέμα. Ευχαριστώ, ναι. Σύντομα, γιατί δεν θέλω να κουράσω τους συναδέρφους. Χτες έστειλα στους Κιώδης μία επιστολή ζητώντας τους να έρθουν σήμερα γιατί ήθελα να τους ενημερώσω, δεν μπόρεσα να βρεθώ με όλους, πάντως θα τους στείλω όλα ποια είναι η κατάσταση πραγμάτων. Λοιπόν, όπως ξέρετε, Έχουμε περίπου όλη αυτή την νομοθετική θετία, τρία χρόνια δηλαδή, προσπαθώντα να διαπραγματευτούμε με την Επιτροπή και το Συμβούλιο έκθεση που έγκρινε ήδη στα τέλη της προηγούμενης θητείας το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο την έκθεση David Martin, αλλά αυτό δεν πέτυχε. Όπως θα γνωρίζετε, η Επιτροπή και το Συμβούλιο για χρόνια, μέχρι το τέλος της προηγούμενης χρονιάς, οι διάφορες προεδρίες δεν κατάφεραν να καθίσουν το Συμβούλιο και η Επιτροπή μαζί μας να συζητήσουμε για την έκθεση αυτή. Στα τέλη της προηγούμενης χρονιάς η Σλοβακική Προεδρία μας πρότεινε μία λύση. Η λύση ήταν σε συνάντηση που είχαμε κύριε Χούμπνερ και εγώ με τη Σλοβακική Προεδρία του Συμβουλίου και μας πρότεινε λοιπόν οι νομικές υπηρεσίες των τριών θεσμικών εργάνων, δηλαδή Κοινοβούλιο, Συμβούλιο και Επιτροπής, να καθίσουν και να συζητήσουν άτυπα προκειμένου να εκπονήσουν ένα κείμενο το οποίο θα μπορούσε να οδηγήσει σε διάλογο μεταξύ των τριών θεσμικών οργάνων. Προκειμένου τα νομικά προβλήματα που τίθενται να μπορούν να λυθούν έτσι. Η διαδικασία αυτή δουλεύτηκε τους τελευταίους μήνες και ανάμεσα στον Ιανουάριο και τον Ιούνιο του 2017 οι νομικές υπηρεσίες των τριών θεσμικών οργάνων είχαν διάφορες συναντήσεις μεταξύ τους και τελικά κατάφεραν να καταλήξουν σε κάποιο κείμενο που να μπορεί να είναι το κατάλληλο κείμενο ώστε να λυθούν τα νομικά ζητήματα τα οποία τίθενται με το προηγούμενο η συμφωνία αυτή, η άτυπη έτσι, ανεπίσημη, ε, πετέχθηκε μεταξύ των τριών νομικών υπηρεσιών, των τριών θεσμικών οργάνων τον Ιούνιο. Τόσο η κυρία Χούμπνερ όπως και εγώ ενημερωθήκαμε για το ότι το κείμενο πήγε πια στους νομικούς συμβούλους. Έτσι, στους επικεφαλείς δηλαδή των νομικών υπηρεσιών των τριών οργάνων και πιστεύαμε ότι θα εγκρίναν το, τελικά το κείμενο αυτό τον Ιούνιο, τον Ιούλιο. Δεν έγινε όμως αυτό. Και όχι μόνο δεν έγινε, αλλά επιπλέον εξακολουθούμε να περιμένουμε οι υπεύθυνοι των τριών θεσμικών οργάνων να έρθουν και να μας πούν κατά πόσο συμφωνούν ή όχι με το κείμενο αυτό. Ζήτησα επανειλημμένα να έχουμε ενημέρωση. Φαίνεται λοιπόν ότι τα προβλήματα που έχει τόσο το Συμβούλιο όσο και η Επιτροπή δεν τους επέτρεψαν να συμφωνήσουν με αυτό το κείμενο το οποίο είναι τεχνικό και το οποίο διαπραγματεύτηκαν μεταξύ τους οι νομικές υπηρεσίες των ε, τριών θεσμικών οργάνων. Θέλω λοιπόν να πω και στου Κιώδη, αλλά και σε όλα τα μέλη της Επιτροπής μας εδώ, ότι εφόσον εγκριθεί το κείμενο αυτό από τα θεσμικά όργανα, η Επιτροπή μας, ΑΦΚΟ, θα έπρεπε να αποφασίσει ότι αυτό θα αποτελούσε τη βάση για να εγκρίνουμε ένα διαφορετικό κείμενο από εκείνο του David Martin, βάση τριμερούς διαλόγου για μια μετέπειτα συμφωνία. Όπως ξέρετε, Μόνο μια συμφωνία με το Συμβούλιο και την Επιτροπή θα μας επέτρεπε να πάμε το κείμενο στην Ολομέλεια να εγκριθεί οριστικά. Δεν χρειάζεται να σας υπενθυμίσω εδώ ότι πρόκειται για ένα κανονισμό. Άρα, πρόκειται για ένα νομικό κείμενο ιδιαίτερη σημασίας όπου αποφασίζονται οι αρμοδιότητες του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου όταν πρόκειται για επιτροπές μέσω των οποίων μπορεί να ασκήσει το δικαίωμά του εξέτασης των πραγμάτων το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Σας υπενθυμίζω ότι αυτό έγινε και με τα Panama Papers για τις εκπομπές ε, αυτοκινήτων, το περίφημο Dieselgate, που οδήγησε επίσης σε διερευνητική επίτροπη και θα μπορούσαν να δημιουργηθούν και άλλες επιτροπές στο μέλλον. Πρόκειται για μια πολιτική λογική. Αδιαφεσβήτητη. Προφανώς και ένα κοινοβούλιο πρέπει να μπορεί να ασκήσει το δικαίωμά του ελέγχου της εκτελεστικής εξουσίας και είναι δικαίωμα που έχουν όλα τα εθνικά κοινοβούλια. Πρόκειται λοιπόν για ένα δικαίωμα ερεύνησης, εξέτασης των πραγμάτων. Έτσι λοιπόν σήμερα ήρθα εδώ για να σας πω ότι δεν έχω απάντηση από τα θεσμικά όργανα και κατά τη γνώμη μου πλέον το ζήτημα γίνεται πολιτικό. Γι' αυτό και προτείνω τέσσερις πρωτοβουλίες που κατά τη γνώμη μου θα έπρεπε να θετήσει η Επιτροπή μας, ΑΦΚΟ. Πρώτον, να ενσωματώσουμε την, ε, το έτοιμά μας για απάντηση από την Επιτροπή και το Συμβούλιο στο κείμενο που θα στείλει ο Πρόεδρος του Κοινοβουλίου στους Πρόεδρους Επιτροπής και Συμβουλίου αυτό που ονομάζουμε κοινή δήλωση για το νομοθετικό πρόγραμμα του 2018. Το ετοιμάζω εγώ αυτό με ανακοινώσεις ΣΕΡΠΑΣ που ετοιμάζουν την δήλωση αυτή και η δικιά μου πολιτική ομάδα. Αλλά αυτό είναι ένα πράγμα που πρέπει να γίνει. Ότι δηλαδή η επιστολή του Προέδρου Ταγιάννη που θα πάει στους Προέδρους ε, Τούσκ και ε, Γιούνκερ να συμπεριλαμβάνουν το αίτημα αυτό. Το δεύτερο που προτείνω, Πρόεδρε, είναι η κυρία Χούμπνερ και εγώ ο ίδιος να μιλήσουμε τον κύριο Ταγιάννη για να το εξηγήσουμε πώς έχουν τα πράγματα. Κατά τη γνώμη μου έχουμε φτάσει σε μια ακραία πια κατάσταση και ο πρόεδρος του Κοινοβουλίου πρέπει να ενημερωθεί για το τι συμβαίνει και ποια είναι η θέση μας. Γιατί δεν θα ήταν καλό κύριο Σταγιάννη όταν βρεθεί με το Συμβούλιο στη Δέσκεψη κορυφή το Δεκέμβριο να μην γνωρίζει. Αντίθετα πρέπει να είναι σε θέση να μεταφέρει τη διαμαρτυρία μας στην Επιτροπή και το Συμβούλιο. Τρίτη μου πρόταση. Προφορική ερώτηση. Το Δεκέμβριο. Στην επόμενη δηλαδή σύνοδο, προκειμένου ο κύριος Τίμερμανς να απαντήσει για την πολιτική θέση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής όσον αφορά αυτή την κατάσταση πραγμάτων. Και η τέταρτη πρωτοβουλία που σας προτείνω είναι η δυνατότητα η Επιτροπή μας, κυρία Πρόεδρε, να ζητήσει από τη νομική υπηρεσία της Επιτροπής του Κοινοβουλίου μελέτη για τις δυνατότητες που έχουμε ε, πρόσβαση στο Ευρωπαϊκό Δικαστήριο προκειμένου εάν γίνεται να έχουμε μία νομική γνωμοδότηση του δικαστηρίου εφόσον δεν έχουμε απάντηση από την Επίτροπη Συμβούλιο ή επειδή δεν έχουμε συνεργασία από την Επιτροπή και το Συμβούλιο ή επειδή δεν έχουμε ικανοποιητική συνεργασία από την Επιτροπή και το Συμβούλιο. Να πούμε ότι το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο έχει αναλάβει πρωτοβουλία, όμως δεν έχουμε καμία απάντηση από τα δύο άλλα θεσμικά όργανα. Αυτά είχα να σας πω λοιπόν και περιμένω και τις δικές σας απόψεις. Ευχαριστώ. Ευχαριστούμε πολύ. Έχουμε μεγάλο κατάλογο και σχεδόν οι περισσότεροι δεν είναι εδώ, αλλά ο Χέλμουτ είναι εδώ, ο Μάξ είναι εδώ, οπότε αν θέλετε να πάρετε το λόγο πριν από τους υπόλοιπους, ε, παρακαλώ, Χέλμουτ Σόλτς. Θα είμαι σύντομο γιατί το ερώτημα το έθεσε και ο εισηγητής. Τον ευχαριστώ για τις παρατηρήσεις του. Επί της αρχής συμφωνούμε και εγώ ε, τον υποστηρίζω ναι, χρειαζόμαστε αυτό το δικαίωμα ε, για το Κοινοβούλιο. Χρειαζόμαστε διαβούλευση και να απαιτούμε εξηγήσει από το Συμβούλιο. Οπότε θα πρέπει εδώ να προσπαθήσουμε να ενισχύσουμε τη θέση μας ως Κοινοβούλιο. Διότι όπως είπατε, Panama Papers, Paradise Papers, Dieselgate, όλα αυτά τα πράγματα, αυτή είναι η καθημερινότητά μας, δυστυχώς. Και είναι δύσκολη η ενασχόληση με όλα αυτά. Ε, Όποτε Υποστηρίζω τον εισηγητή. Ευχαριστώ, Μαξ. Σημερίζομαι την εντύπωση του εισηγητή ότι το Συμβούλιο δεν παίζει δίκαια. Υποτιθώ ότι θα πρέπει να διαπραγματευόμαστε πάνω στο θέμα αυτό σύμφωνα με τη συνθήκη. και μπορεί το Συμβούλιο να έχει λόγου που να αξίζει τον κόπο να εξετάσουμε, αλλά φαίνονται απρόθυμοι ακόμη και να ξεκινήσουν τι διαπραγματεύσει. Και δεν είναι αυτό ο τρόπο που ότι πρέπει να γίνονται τα πράγματα αυτά. Συγχαίρω λοιπόν τον εισηγητή για την πολύ δύσκολη δουλειά του να καταφέρει το Συμβούλιο και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή να ε, συνεργαστούν μαζί μας και να κάνουν αυτό που πρέπει. Εύχομαι κάθε επιτυχία στις εργασίες μας, ε, στην προσέγγιση αυτή που νομίζω ότι αξίζει τον κόπο να προσπαθήσουμε να ακολουθήσουμε. Ευχαριστώ πολύ. Άλλος κανείς που να θέλει να πάρει το λόγο. Θα πρέπει να αποφασίσουμε τι θα κάνουμε τώρα. Νομίζω ότι η οι ιδέε του ΡΑΜΟΝ σχετικά με τα διάφορα βήματα μπορούν να υιοθετηθούν όλες. Θα, θα πρέπει λοιπόν να αφήξουμε το θέμα αυτό σε επίπεδο προέδρων των θεσμικών οργάνων. Πρέπει να χρησιμοποιούμε όλα τα κανάλια που σχετίζονται με, την, το πρόγραμμα εργασίας της Επιτροπής. Και η κυρία Βίκστρομ έθεσε το θέμα αυτό στον Πρόεδρο. Είχαμε λοιπόν το θέμα της ε, κοινή ε, δήλωση. Ε, μπορούμε να το ξαναζητήσουμε, αλλά φοβάμαι ότι δεν θα λειτουργήσει το θέμα αυτό. Και ο Ραμόν πολύ ευγενικά το είπε το τι κάνουμε τα τελευταία τρία χρόνια. Είχαμε πολύ δύσκολε συναντήσει με διάφορες προεδρίες. για μεταξύ άλλων και την εκπόνηση νέου εγγράφου. είναι θέμα που σχετίζεται και με το ρόλο της Προεδρίας στο Συμβούλιο. Και η εντύπωσή μου είναι ότι οι νομικές υπηρεσίες ασχολούνται με το θέμα αυτό εδώ και αρκετό χρόνο και έχουν ξεκαθαρίσει όλα τα δύσκολα θέματα. Όλα πλόκαραν στις γνωμοδοτήσεις των νομικών υπηρεσιών. Νομίζαμε ότι τώρα πια αυτό είναι σαφές, αλλά φαίνεται ότι οι γνωμοδοτήσεις τώρα σε κάποια θεσμικά όργανα, όχι στο Κοινοβούλιο, έχουν πάει σε πολιτικό επίπεδο. και φαίνεται το ότι αυτή η συζήτηση σε πολιτικό επίπεδο αποτελεί εμπόδιο για μας. Θα πρέπει λοιπόν να το θέξουμε απέναντι στον ε, Πρόεδρο Ταγιάννη. Αλλιώς δεν νομίζω ότι θα μπορέσουμε να προχωρήσουμε στο θέμα αυτό. Προτείνατε και προφορική ερώτηση. Να θέσουμε ερώτηση στην Ολομέλεια και προς το Συμβούλιο και προς την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Νομίζω λοιπόν ότι και αυτό είναι μια καλή ιδέα. Θα ζητήσουμε λοιπόν να γίνει αυτό. Και δεν ξέρω τι άλλο μπορούμε να κάνουμε στην παρούσα φάση. Ας προχωρήσουμε λοιπόν στην προφορική ερώτηση. Ας συνομιλήσουμε με τον πρόεδρο Ταγιάννη όσο γίνεται πιο σύντομα. Ή να προσπαθήσουμε οι πολιτικοί ηγέτες ή η διάσκεψη των πρόεδρων να ασχοληθεί με το θέμα. Ο κύριος Βίλαντ. να δούμε τη νομική οδό. Κατά πόσο δηλαδή το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο μπορεί να ζητήσει την άποψη του δικαστηρίου. Ας ρωτήσουμε την νομική μας υπηρεσία, αν νομίζετε κυρία Πρόεδρε, να ζητήσουμε από την νομική μας υπηρεσία να μελετήσει αυτή τη δυνατότητα. ίσως να τη συνδυάσουμε με τις άλλες ιδέες, έτσι. Ναι, ναι. Εμείς ως Επιτροπή δεν μπορούμε να το κάνουμε. Πρέπει να μιλήσουμε με τον Ταγιάννη. Γιατί μόνο ο πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου μπορεί να το κάνει αυτό. Οπότε πρέπει να αρχίσουμε από την προφορική ερώτηση, λέω εγώ, να μιλήσουμε με τον Ταγιάννη για την ιδέα αυτή. Να δούμε αν υπάρχει δυνατότητα να ζητήσουμε την άποψη του δικαστηρίου. Ωραία, ολοκληρώνεται αυτό το θέμα στην ημερήσια διάταξη. Εντάξει, δεν έχω άλλου ομιλητέ, κανεί κατά. Καλώ. Τώρα έχουμε ένα πρόβλημα όμω. Γιατί έχουμε εδώ του φίλου μα για τα δικαιώματα των ε, πολιτών ε, στο Ηνωμένο Βασίλειο. Ίσως δεν ξέρω Προβλέπετε για τις 5 και 20. Βέβαια εσείς είσαστε ήδη εδώ. Ας αρχίσουμε και ελπίζω ότι οι συνάδελφοι που θα εμφανιστούν αργότερα να μην έχουν αντίρρηση. Δεν ξέρω, θέλετε να αρχίσουμε τώρα ή να τους περιμένουμε. Να αρχίσουμε. Ωραία, δεν ξέρω πώς έχετε οργανωθεί, ποιος θα αρχίσει. Ρε, πάρτε το λόγο, όπως έχετε αποφασίσει εσείς, παρουσιαστείτε, πείτε μας ε, ποιες είσαστε. Αν θέλετε να περιμένουμε, να περιμένουμε. Ίσως είναι καλύτερα. Εμεί έχουμε χρόνο. Ναι, βέβαια υπάρχει και ο φόβος ότι θα φύγουν αυτοί που είναι εδώ και ίσως δεν έρθουν οι επόμενοι. Είναι λίγο επικίνδυνο θέλω να πω. Είναι μια φρικτή μέρα γιατί όλοι έχουν συγχρόνω πολλές και διαφορετικές συνεδριάσεις. Επίσης να ξέρετε ότι μεταδίδεται στο διαδίκτυο έτσι καλώς η συνάντηση, οπότε νομίζω και εγώ ότι είναι καλύτερα να αρχίσουμε τώρα. Α, ο Χέλμουτ όμως κάτι έχει να πει. Να περιμένουμε πέντε λεπτά. Πέντε λεπτά. Πέντε λεπτά να περιμένουμε και μετά να αρχίσουμε, γιατί κάποιος μπορεί να είναι στο δρόμο. Ελπίζω να έρθουν και άλλοι συνάδελφοι στο μεταξύ. Καλά, να ελπίσουμε, αλλά δεν ελπίζω και πολύ, λέει η Πρόεδρος. Ό,τι θέλετε εσείς. Αν θέλετε να περιμένουμε, να περιμένουμε. Αν δεν θέλετε να αρχίσουμε. You want to wait minutes Θέλετε να περιμένουμε πέντε λεπτά ή θέλετε να αρχίσουμε, συνάδελφοι. Τους, τους προσκεκλημένες μας ρωτάω. Ωραία. Αρχίστε. Παρακαλώ. Σας ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ. Θα ξεκινήσουμε. Πρώτα θα μιλήσει η οργάνωση British in Europe και κατόπιν θα μιλήσουν οι συνάδελφοί μας ε, από την οργάνωση τα 3 εκατομμύρια, το 3 million. Λέγομαι Jane Golding, είμαι πρόεδρος της British in Europe και για όσους από εσάς δεν μας γνωρίζουμε, είμαστε ε, ένας συνασπισμός 10 ομάδων πολιτών Βρετανών ε, που ζουν στα 27 κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης ε, και έχουμε περίπου 34.000 μέλη. Συνεργαζόμαστε στενά με τους συναδέλφους μας από την οργάνωση The 3 Million που εκπροσωπούν τη μεγαλύτερη ομάδα πολιτών της Ευρωπαϊκής Ένωσης στο Ηνωμένο Βασίλειο. 1,2 ε, εκατομμύρια Βρετανών βρίσκονται στο Ηνωμένο, ε, στην Ευρωπαϊκή Ένωση σύμφωνα με τους υπολογισμούς ε, και πολλοί από αυτούς είναι οικονομικά ενεργοί και το 27% στην Ισπανία και αλλού είναι συνταξιούχοι. πολύ μεγάλος αριθμός λοιπόν βρίσκονται σε ηλικία εργασίας ή είναι νεότεροι. Ε, συνεργαζόμαστε στενά λοιπόν με τους αδέρφους μας ε, ε, από την οργάνωση στα 3 εκατομμύρια. Το Brexit δεν είναι κάτι που επιθυμούσαμε και η πλειοψηφία των ε, μελών μας, όπως ε, και των τριών εκατομμυρίων, ε, δεν έχουν ψήφο σχετικά με το μέλλον μας. Υπολογίζουμε ότι το 60% των British in Europe δεν είχαν το δικαίωμα ψήφου. Ε, πιστεύουμε όμως σε εσά, πιστεύουμε στην Ευρωπαϊκή Ένωση, πιστεύουμε ότι θα προστατεύσει τα δικαιώματά μας και επικροτούμε την προσέγγιση της Ευρωπαϊκής Ένωσης στις διαπραγματεύσεις και τις βασικές αρχές σχετικά με τα δικαιώματα των πολιτών. Οι διαπραγματεύσεις ε, ξεκίνησαν ε, και μοιραία. Αυτό οδήγησε σε επιδείνωση της ε, κατάστασης όσον αφορά τα δικαιώματα των πολιτών δεδομένων των προτάσεων του Συμβουλίου του Ηνωμένου Βασιλείου. Αυτή τη στιγμή δεν έχουμε πολύ εμπιστοσύνη στο Ηνωμένο Βασίλειο όσον αφορά την υπεράσπιση των δικαιωμάτων μα, διότι πιστεύουμε ότι ο στόχο του είναι να προχωρήσουν στη δεύτερη φάση των διαπραγματεύσεων. Μάλιστα, πιστεύουμε ότι έχουν οπισθοχωρήσει σε μεγάλο βαθμό κατά τη διάρκεια τη πρώτη φάση. Τώρα λοιπόν βασιζόμαστε στην Ευρωπαϊκή Ένωση και σε εσά να συνειδητοποιήσετε ότι φαίνεται να έχουμε ανταγωνισμό προ τα κάτω ώστε να καταλήξουμε σε μια κατάσταση UK Plus και Ευρωπαϊκή Ένωση μείον. Δηλαδή η βελτίωση της πρότασης του Ηνωμένου Βασιλείου και η επιδείνωση της ε, πρότασης ε, της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Και ε, φοβόμαστε ότι κάτι τέτοιο θα επιβεβαιωθεί τον Δεκέμβριο παρά τις δηλώσεις ότι ε, το Brexit δεν θα ε, επηρεάσει τη ζωή των ε, Ευρωπαίων πολιτών στο Ηνωμένο Βασίλειο και των Βρετανών στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Τα πράγματα κινούνται πάρα πολύ γρήγορα αυτή τη στιγμή. Έχουμε εξελίξεις κάθε εβδομάδα ή και πιο συχνά. Και η παρούσα θέση είναι ότι δεν θα υπάρξει κατάλληλη προστασία των δικαιωμάτων των πολιτών της Ευρωπαϊκής Ένωσης στο Ηνωμένο Βασίλειο αυτή τη στιγμή στις διαπραγματεύσεις μικρές προσαρμογές όσον αφορά διοικητικές διαδικασίες ε, δεν ε, αντισταθμίζουν τη βασική θέση ότι οι ε, πολίτες Ευρωπαϊκής Ένωσης θα ζητήσουν ένα καθεστώς αναγνώρισης σε εχθρικό περιβάλλον. Και μάλιστα υπάρχει και αμοιβαιότητα. Φοβούμαστε δηλαδή ότι χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης θα εφαρμόσουν ανάλογες διαδικασίες ε, μετα... μετανάστευσης ε, Βρετανών πολιτών στις χώρες τους. Και αυτά που συζητώνται αυτή τη στιγμή ε, σημαίνει όχι επιβεβαίωση των δικαιωμάτων, τα δικαιώματα αυτά θα εφαρμόζονται κατόπιν αιτήματος. Θέλουμε επίσης να υπάρχουν ε, ακόμη τα δικαιώματα ελεύθερης κινητικότητας και το δικαίωμα επιστροφής στο Ηνωμένο Βασίλειο, αλλά αυτά τα δικαιώματα δεν φαίνεται ότι θα διατηρηθούν αυτή τη στιγμή στις διαπραγματεύσεις. Όσον αφορά την αναγνώριση επαγγελματικών ε, προσόντων, ε, πάλι φαίνεται ότι κάποια επαγγελματικά προσόντα δεν θα αναγνωρίζονται και αυτά που θα αναγνωρίζονται όπως και τα οικονομικά δικαιώματα θα περιορίζονται στο κράτος κατοικίας. Επίσης ε, θα υπάρχουν περιορισμοί όσον αφορά την επανένωση οικογενειών και για τις δύο ομάδε, ε, και για τους ε, Βρετανούς στην Ευρωπαϊκή Ένωση και τους Βρετανούς υπηκόους που επιστρέφουν στο Ηνωμένο Βασίλειο και έτσι έχουν δικαιώματα σύμφωνα με το δίκαιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης κατά την επιστροφή τους όσο έχουν τα πράγματα αυτή τη στιγμή η θέση της Ευρωπαϊκής Ένωσης όσον αφορά την ελεύθερη κινητικότητα, τα ε, επαγγελματικά προσόντα και τα οικονομικά δικαιώματα ε, είναι πολύ δυσνόητα αυτή τη στιγμή και φαίνεται ότι θα επηρεάσουν τα δικαιώματα αυτή τη στιγμή φαίνεται. Οι πολίτες της Ευρωπαϊκής Ένωσης ε, που διαμένουν στην, ε, στο Ηνωμένο Βασίλειο φαίνεται ότι δεν θα αναγνωριστούν τα δικαιώματά τους όταν επιστρέψουν σε χώρες Ευρωπαϊκής Ένωσης μετά το Brexit. Και πολίτες Ε, Βρετανοί ε, που αποχωρούν ε, από την χώρα για μεγάλο χρονικό διάστημα μέχρι τώρα είχαν δικαίωμα επιστροφής στη χώρα τους, αλλά φαίνεται ότι και αυτό θα επηρεαστεί. Κατά τη γνώμη μας όλα αυτά μπορεί να αντιστραφούν όμως. Οι διαπραγματευτικές οδηγίες και οι βασικές αρχές που συμφώνησε η Ευρωπαϊκή Ένωση είναι αρκετά ευρεία ώστε να επιτρέψουν κάτι τέτοιο. Η παράγραφος 20 της διαπραγματευτικής οδηγίας στόχο έχει να προστατεύσει το καθεστώς και τα δικαιώματα που απορρέουν από την νομοθεσία της Ευρωπαϊκής Ένωσης κατά την ημερομηνία αποχώρησης συμπεριλαμβανομένων ε, αυτών που θα προκύψουν αργότερα, για παράδειγμα δικαίωμα ε, σύνταξης ε, καθώς και δικαιώματα που αυτή τη στιγμή αποκτώνται και οι βασικές ε, αρχές για τα δικαιώματα των πολιτών είναι ακόμα πιο σαφείς. Λέει ότι παρόμοιο επίπεδο προστασίας ε, καθορίζεται στην Ευρωπαϊκή Νομοθεσία για τους πολίτες Ευρωπαϊκής Ένωσης ε, στο Ηνωμένο Βασίλειο και για τους πολίτες τους Βρετανούς στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Με άλλα λόγια, τα δικαιώματα που υπάρχουν πριν την αποχώρηση των δύο αυτών ε, ομάδων ε, θα πρέπει να ε, διαφυλαχθούν. Επιπλέον, όσον αφορά το θέμα της ελεύθερης κινητικότητας, η προστασία της ελεύθερης κινητικότητας επίσης αναφέρεται ρητά στις διαπραγματευτικές οδηγίες στην παράγραφο 21 και αυτό δεν είχε συμπεριληφθεί στο αρχικό σχέδιο, προσθέθηκε στην τελευταία εκδοχή του κειμένου. Ζητάμε λοιπόν να υπάρξει πρόοδος μόνο εφόσον επιληθούν όλα αυτά τα θέματα. Αλλιώς τα δικαιώματα των ανθρώπων θα είναι απλά ένα θέμα μεταξύ πολλών ε, στην τελική φάση. Και θα έχουμε σημαντικό περιορισμό των ε, δικαιωμάτων αυτών. Και όταν τελικά ε, καταλήξουμε σε μια ολοκληρωμένη συμφωνία, θα πρέπει να υπάρχει τουλάχιστον μια ρήτρα διασφάλισης ώστε τα δικαιώματα αυτά να ε, συνεχίσουν να ισχύουν άσχετα από το ποιο θα είναι το αποτέλεσμα ε, των διαπραγματεύσεων σε άλλους τομείς ε, στην Συμφωνία Αποχώρησης. Πέρα από τα νομικά θέματα όμως, ποιες είναι οι κοινωνικές και ανθρώπινες διαστάσεις, κάτι που συζητήθηκε πρόσφατα στο Γκέτεμποργκ. Είμαστε παιδιά της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ένα εγχείρημα που στόχο έχει την επίτευξη της ειρήνης και της αλληλεγγύης. Ο Γερμανός πεθερός μου επέζησε στα 16 του τον βομβαρδισμό της Δέσδης ε, και ήλπιζε τα παιδιά του και τα εγγόνια του ε, να ζήσουν ε, σε έναν χώρο Ειρηνή και ελευθερία. Εμείς οι πολίτες λοιπόν έχουμε προχωρήσει τις αρχές πολύ πιο πέρα από ό,τι οραματίστηκαν οι ιδρυτές πατέρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Οι δύο οργανώσεις λοιπόν, ε, British and Europe και τα 3 εκατομμύρια, ε, είναι τώρα όμοιροι μιας κατάστασης. Ε, μας ζητήθηκε να βάλουμε κατά μέρο τις διαφορές μας και να εξετάσουμε τις ομοιότητές μας. Εάν λοιπόν μας απογοητεύσετε τώρα, θα θρηματίσετε τα όνειρά μας. Ε, και θα στείλετε έτσι το μήνυμα ότι το να υιοθετήσει κανείς την ευρωπαϊκή ηθαγένεια είναι κίνδυνος και μπορεί να επιβληθούν κυρώσεις σε όσους ε, το κάνουν αυτό. Η ευρωπαϊκή ηθαγένεια είναι ένα ε, θεμελιώδες καθεστώς και θα πρέπει να το προστατεύσετε τώρα. Αν όχι τώρα, πότε. Σας ευχαριστώ. Ευχαριστώ πολύ από ό,τι κατάλαβα. Τώρα για τους 3 ε, million θα μιλήσει η κυρία Λοντάνσκο. Καλησπέρα σας. Είμαι η Άννα Λοντάνσκο. Είμαι Γαλλίδα Επικός, ε, Ευρωπαία Επικός και συνειδητής των 3 million που δημιουργήθηκε τον Ιούλιο του 2016 μετά από τα αποτελέσματα του δημοψηφίσματος Έχουμε περίπου 35.000 μέλη. Δεν μπορώ παρά να επαναλάβω τα όσα είπε συναδελφός μου Τζέικ από τους British in Europe. Όλοι μας είμαστε παιδιά της Ευρώπης, πράγματι παιδιά του ευρωπαϊκού οικοδομήματος. Δραστήριοι Ευρωπαίοι που δώσαμε ζωή στο έργο αυτό 3 εκατομμύρια Ευρωπαίοι πολίτες αποκλείστηκαν από το δημοψήφισμα του Ιουνίου του 2016 παρότι πολλοί από εμάς κατοικούσαμε ε, εδώ και δεκαετίες στο Ηνωμένο Βασίλειο και είχαμε φτιάξει τις ζωές μας εκεί, πληρώναμε φόρους, συνεβάλαμε, ε, συμβάλαμε με διάφορους τρόπους στην κοινωνία του Ηνωμένου Βασιλείου και στα οικονομικά του Ηνωμένου Βασιλείου είχαμε περιορισμένη συμμετοχή στις διαπραγματεύσεις και ανησυχούμε ότι στη φάση 2 θα υπονομευθούν τα βασικά μας δικαιώματα. Από την άποψη των 3 εκατομμυρίων έχει σημειωθεί κάποια πρόοδο σε κάποιους τομείς, ωστόσο είναι σαφές ότι πολλά ζητήματα έχουν παραμείνει ανεπιλήτα. Αυτές οι πιθανές ε, ε, ε, δεινές συνέπειες για τους πολίτες ε, που κατοικούν στο ε, Ηνωμένο Βασίλειο μας οδηγούν σε προβλήματα σε τρεις ε, τομείς. Πρώτον, συνταγματικά. Το πρώτο πρόσκομα εδώ είναι η πιθανότητα προσφυγή στο δικαστήριο για κάποιες υποθέσεις αλλά αυτά που μάθαμε χθε ίσως είναι καλές ειδήσει. θα δούμε τι θα γίνει θα πρέπει να περιμένουμε να δούμε κατά πόσο θα υπάρξει κάποιο πλαίσιο και μετά χωρίς ε, τη, τη συμμετοχή του δικαστήριου υπάρχει περίπτωση να υπάρχουν διαφορετικές ερμηνείες και να υπονομευθούν τα δικαιώματά μας. Τώρα, όλα αυτά που λέει ότι θα επιβάλλει το ΕΒ σε Ευρωπαίους πολίτες στο ΕΒ θα χάσουμε τα δικαιώματά μας. Μιλάμε για απώλεια, για εξαφάνιση των δικαιωμάτων ε, με υποχρέωση ε, υιοθέτηση ενό νέου καθεστώτος με λιγότερα δικαιώματα. Κάτι πολύ δύσκολο να αναστραφεί. Από την άλλη, λυπούμαστε που η Ευρωπαϊκή Ένωση δεν έχει διαμαρτυρηθεί για αυτό το καθεστώς. Ε, πολλά προβλήματα θα υπάρχουν στην οικογενειακή επανένωση. Θα έχουμε την απώλεια δικαιωμάτων όσον αφορά την ελεύθερη κυκλοφορία. Για παράδειγμα, πολλά προγράμματα χρηματοδοτούνται από την Ευρωπαϊκή Ένωση, οπότε αυτή τη στιγμή αν ζω στο Ηνωμένο Βασίλειο μπορώ να συμμετέχω αν θέλω, αλλά αργότερα μετά τον Brexit δεν θα μπορώ. Σε θέματα απασχόλησης, ε, έργα απασχόλησης για παράδειγμα, οτιδήποτε χρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση θα πάψει να είναι ανοιχτό σε εμά. Η πρόσβαση στα δικαιώματά μας μέσω διοικητικής διαδικασίας, αυτό ε, στα μάτια μας δεν υπάρχει ακόμα απλουστευμένη διαδικασία για να, καταγραφούν, για να γραφούν ε, τα τρία εκατομμύρια πολίτες και δεν υπάρχει ακόμα το καθεστώς. Δηλαδή αυτό εμείς λέμε ότι αυτή η διαδικασία είναι τρομακτική. Μιλάμε για πάρα πολλά έγγραφα και το βάρος απόδειξη ε, βαρύνει τον ετούντα μάλιστα. Αλλά ένα απλοποιημένο καθεστώς, μια απλοποιημένη διοικητική διαδικασία δεν σημαίνει ότι το καθεστώς ε, θα είναι σωστό ή αποδεκτό. Πράγματι η διοικητική διαδικασία ε, παρουσιάζει διάφορα προβλήματα. Υπάρχουν πολλά παραδείγματα σήμερα σε σχέση με το νέο καθεστώς έλεγχη ποινικού μητρώου, έλεγχη ε, διαγωγής ε, που θα καλύπτουν ολόκληρο το διάστημα που έχει παραμείνει ε, κάποιος στο Ηνωμένο Βασίλειο. Επίσης, θύνται ζήτηματα δοκιμές έλεγχη εργασίας, επαρκής πόρη, όσον αφορά την ασφάλεια υγείας Χαιρόμαστε που η κυβέρνηση του Ηνωμένου Βασιλείου λέει ότι θα εξαιρούμαστε υπό το νέο καθεστώ. Ωστόσο, το ζήτημα των επαρκών πόρων δεν έχει αναλύθει επαρκώ. Ενώ γνωρίζουμε ότι χρησιμοποιείται ω βάση για διαταγέ απέλαση. Τι σημαίνει αυτό για του υπευθύνου φροντίδα ή για ανθρώπους με ασταθή έσοδα ή για άτομα με μακροχρόνιες ασθένειες. Τι μπορούν να αναμένουν, τι μπορούν να ελπίζουν αν όλα αυτά δεν διευκρινιστούν σύντομα. Μετά έχουμε το εχθρικό αυτό περιβάλλον, η κυβέρνηση του Ηνωμένου Βασιλείου. Όλο μας λέει ότι αυτό δεν αποτελεί ζήτημα. Αλλά αυτό δεν είναι αλήθεια. Διαρκεί, διαρκώς χρησιμοποιεί αυτό το παράδειγμα της απλουστευμένης διαδικασίας ως παράδειγμα καλής ε, βούλησης. Ταυτόχρονα όμως αγνοεί τις πολλές ε, περιπτώσεις ε, διαφόρων περιστατικών ξενοφοβίας και παρενόχλησης που ε, βιώνουν οι Ευρωπαίοι πολίτες ε, στην καθημερινότητά τους για να ανοίξουν λογαριασμούς τραπεζικούς, ε, στον τομέα της στέγασης, στην πρόσβαση, στην υγεία και μάλιστα το, η κυβέρνηση του Ρωμαν προσπαθεί να διερευνήσει, να βρει πού βρίσκονται όλοι αυτοί οι ξένοι και ποια είναι η κατάστασή τους. Επίσης όλα αυτά αγνοούν ε, τα νούμερα της κυβέρνησης για τα εγκλήματα μίσους ε, που έχουν σημειώσει τεράστια αύξηση ειδικότερα μετά από το δημοψήφισμα. Μετά από το δημοψήφισμα είχαμε ε, γεωμετρική αύξηση όλων αυτών των εγκλημάτων χωρίς να αναφέρουμε τους ανθρώπους που δολοφονήθηκαν μετά από το δημοψήφισμα πέρυσι τον Ιούλιο και τον Αύγουστο. Ο συμπέρασμα όπως είπε και Τζέιν, θεωρούμε ότι υπάρχει ελπίδα, ελπίδα στις διαπραγματευτικές ε, οδηγίες, ε, υπάρχει ελπίδα για ευελιξία και αυτό μας φέρνει στις βασικές αρχές. Μια βασική αρχή που φαίνεται να έχει χαθεί μέσα σε όλα αυτά, ότι το Brexit δεν θα πρέπει να αλλοιώσει τις ζωές μας και τα δικαιώματά μας. Δεν θα πρέπει τα δικαιώματά μας να επηρεαστούν από αυτό. Θα θέλαμε να περιχαρακώσουμε τα ε, δικαιώματά μας τώρα, ώστε να σταματήσουν όλα αυτά τα προβλήματα. Οι Ευρωπαίοι πολίτες σε τελική ανάλυση είναι αυτοί που εκπροσωπούν το ευρωπαϊκό οικοδόμο. Όλο αυτό αφορά τι ζωέ των ανθρώπων, όχι εμπορικέ συμφωνίε. Και όπω είπε η Τζέιν, αν δεν το κάνουμε τώρα, πότε. Ευχαριστώ. Thank you. Ωραία, σας ευχαριστούμε πολύ. Η τρίτη. Εσείς, α, εσείς δεν θα πάρετε το λόγο τώρα. Ωραία. Οπότε, Ζητά... Συγγνώμη, πρόεδρο είχε μια άλλη πολύ σημαντική συνάντηση, γι' αυτό ανέλαβα εγώ την Προεδρία. Ρίτσαρντ Και μετά εσείς. Ναι. ναι, σας ευχαριστώ πολύ και ευχαριστώ πολύ για αυτές τις δύο εξαίρετες παρουσιάσεις που εξηγούν τα διάφορα ζητήματα και από πλευρά δηλαδή των ε, Βρετανών στο, στην Ευρωπαϊκή Ένωση και των ε, κατοίκων της Ευρωπαϊκής Ένωσης, μάλλον και των υπηκών της Ευρωπαϊκής Ένωσης στο Ηνωμένο Βασίλειο. Βέβαια, φαίνεται ότι δεν υπάρχει μεγάλη πρόοδος, όχι αρκετή πρόοδος, δυστυχώς. Αυτό λέτε κι εσείς. Από τη δικιά μου άποψη, δεν είμαι βέβαια στο κυβερνών κόμμα του Ηνωμένου Βασιλείου και πράγματι λυπάμαι πάρα πολύ για την ελάχιστη πρόοδο που έχει επιτευχθεί από την ε, αρχή έλεγα ότι θα έπρεπε να διασφαλιστούν τα δικαιώματα των Ευρωπαίων που κατοικούν στον Ηνωμένο Το σημερινό αδιέξοδο στις διαπραγματεύσεις λοιπόν εξακολουθεί να υπάρχει αδιέξοδο. Όσον αφορά το δικαίωμα της επανένωσης οικογενειών που το αναφέρατε και άλλα ζητήματα η αναγνώριση προσόντων κλπ. Αν υπάρξει συμφωνία ποτέ, θα επιβληθεί. Και καταλαβαίνω γιατί οι πολίτες άλλων χωρών δεν εμπιστεύονται τον τρόπο με τον οποίο θα επιβάλλει μια τέτοια συμφωνία. Αν τελικά ο μόνος μηχανισμός που θα ισχύει θα είναι ο Βρετανικός που ήδη θυμόσαστε τις επιστολές που είχαν στείλει και μετά είπα όχι, συγγνώμη λάθος. Οπότε πράγματι υπάρχει θέμα εμπιστοσύνης από τις άλλες χώρες απέναντι στον Ομένο Βασίλειο. Τώρα αν τις επόμενες εβδομάδες, ελπίζουμε. Γιατί ίσως ε, τώρα αρχίζει να υπάρχει πίεση για συμφωνία. Εν πάση περιπτώσει, αν υπάρξει και αν είναι ικανοποιητική αυτή, το γεγονός ότι θα αποτελεί μέρος μιας συνολικής συμφωνίας, η οποία δεν θα επιτευχθεί παρά μετά από άλλον ένα, ένα, χρόνο, αυτό σημαίνει ότι παραμένει αβεβαιότητα για όλους τους ενδιαφερόμενους πολίτες και από τις δύο πλευρές, γιατί αν δεν υπάρχει συμφωνία τελικά υπάρχει κίνδυνος για όλου αυτούς. Τώρα, μπορεί να παρακαμφθεί αυτό με μια χωριστή συμφωνία για παράδειγμα το θέσαμε με τον κύριο Μπαρνιέ, με την Επιτροπή, με άλλους και η απάντηση νομικά μιλώντας είναι αρνητική. Όχι. Αυτό όμως δεν θα πρέπει να εμποδίσει τις δύο πλευρές να προσπαθήσουν να καταλήξουν σε μια πολιτική συμφωνία που θα τηρήσουν και οι δύο, εφόσον επιτευχθεί δηλαδή αυτή. Να κάνουν προσπάθειες να καταλήξουν σε κάποια πράγματα που και οι δύο πλευρές θα τηρήσουν και αν δεν υπάρξει συμφωνία για το άρθρο 50 να υπάρξει κάποιος άλλος μηχανισμός επίλυσης. Αλλά δεν σημαίνει ότι πρέπει να είμαστε καθυσυχασμένοι γιατί υπάρχουν διάφοροι στο Ηνωμένο Βασίλειο και υπουργοί ακόμα που θέλουν η Μεγάλη Βρετανία να εγκαταλείψει χωρίς άρθρο 50. Ξέροντας την εσωτερική αγορά, τους κανόνες της, δεν τα θέλουν ούτε τα περί ηθαγένειας. Θέλουν το Brexit να διαγράψει κάθε σχέση. Κάτι το οποίο θα ήταν καταστροφή σε πολλά μέτωπα. Για όλους. Και κυρίως για το Ρωμανοβασίλειο Βασίλειο. αλλά τι να πω, αυτή είναι η πτέρυγα του σκληρού Brexit στο Ηνωμένο Βασίλειο. Τώρα υπάρχει και μια άλλη διάσταση, ιδιαίτερα επικαιρή. Σήμερα το απόγευμα η Βουλή των Κοινοτήτων συζητάει το θέμα των, του χάρτη θεμελιωδών δικαιωμάτων και κατά πόσο θα πρέπει να παραμείνει στην Βρετανική νομοθεσία ακόμα και όταν θα έχει βγει από την Ευρωπαϊκή Ένωση το Ηνωμένο Βασίλειο. Αυτό συνδέεται και με τις συνέπειες της ε, απόφασης του δικαστηρίου Φρανκοβιτς που τελικά ενσωματώνεται στο δίκαιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης και έχει να κάνει με την μη σωστή εφαρμογή του ευρωπαϊκού δικαίου από μια χώρα και η απόφαση ακριβώς του δικαστηρίου λέει ότι υπάρχει δικαίωμα σε αποζημίωση σε αυτή την περίπτωση. Αλλά η απόφαση αυτή, λέει το Ηνωμένο Βασίλειο, δεν ισχύει πια για το Ηνωμένο Βασίλειο εφόσον αυτό έχει αποχωρήσει. Αυτό είναι άλλο ένα ζήτημα λοιπόν που δείχνει κακή θέληση από πλευράς της Βρετανικής κυβέρνησης. Η εικόνα δεν είναι και τόσο καλή δηλαδή. Άλλη μια πτυχή του Brexit που δεν μας το είπε καθόλου η εκστρατεία του Λίβ, της αποχώρησης δηλαδή ότι θα υπήρχε. Είναι πράγματα τα οποία το απέκρυψαν και οι Βρετανοί τα ανακαλύπτουν σιγά σιγά κάθε μέρα Ανακαλύπτουν δηλαδή όλο και περισσότερα ζητήματα και δυσκολίες που προκύπτουν στη ζωή τους και τα οποία αποσιώπησαν πλήρως όσοι υποστήριζαν τον Brexit στην ε, προεκλογική εκστρατεία. Συσσωρεύονται λοιπόν αυτές οι δυσκολίες και τα προβλήματα και φαίνεται ότι το Brexit είναι κάτι πολύ ζημιογόνο και επικίνδυνο για το Ηνωμένο Βασίλειο και για όλους τους πολίτες ανά την Ευρώπη τελικά. Ευχαριστώ. Ευχαριστούμε. Κύριε Σόλτς, απλά να σας ρωτήσω, έχετε κάτι γραπτό το οποίο μπορείτε να μας αφήσετε ε, σε σχέση με τις ομιλίες σας, γιατί δεν προλάβαμε να καταγράψουμε όλα τα προβλήματα τα γνωρίζουμε φυσικά, αλλά καλό θα ήταν να έχουμε τις δικές σας σκέψεις σε, μια, σε ένα κατάλογο. Ναι, μπορούμε. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Επειδή είναι σε ζωντανή μετάδοση η συνεδρίαση αυτή, θα μιλήσω στα γερμανικά. Διότι αυτό δεν αφορά μόνο τους Βρετανούς, αφορά όλους τους πολίτες των 28 χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, οι οποίοι πρέπει να καταλάβουν τι συζητάμε και πόσο σοβαρό και αποτελεί προτεραιότητα το ζήτημα αυτό είναι των ανθρωπίνων δικαιωμάτων στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Θα ήθελα λοιπόν να καταστήσω σαφές ότι είμαι ευγνώμων για ε, τις παρατηρήσεις ε, των εκπροσώπων των μη που ήρθαν εδώ σήμερα και που μας έδειξαν με πόση αφοσίωση ασχολούνται με το θέμα αυτό. Ε, οι άνθρωποι που επηρεάζονται από την κατάσταση αυτή είναι πάνω από 4 εκατομμύρια και θα ήθελα να πω ότι ε, όπως ε, είπε και το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο στο ψήφισμα του, οι πολίτες δεν αποτελούν αντικείμενο διαπραγματεύσεων. Θα πρέπει η πολιτική να έχει κατά νου τους ανθρώπους αυτούς και να καταλήξει σε μια ε, λύση καλή για αυτούς. Στην πολιτική μας ομάδα, την προηγούμενη εβδομάδα στο Στρασβούργο, είχαμε μια συνάντηση με τον ε, Μισελ Μπαρνιέ, όπου καταστήσαμε σαφές ότι Περιμένουμε θετικά βήματα πάνω στο θέμα αυτό και από τις δύο πλευρές, ώστε να διαφυλαχθούν τα δικαιώματα των πολιτών. Και θα πρέπει τα δικαιώματα των πολιτών, ε, όπως ε, και το θέμα της Βόρειας Ιρλανδίας, να βρίσκονται στο επίκεντρο των διαπραγματεύσεων. Προτού να προχωρήσουμε στη φάση 2 των διαπραγματεύσεων. και τίθεται το θέμα ε, τι ακριβώς είναι η σημαντική πρόοδος, πώς ορίζεται η σημαντική πρόοδος. Θα ήθελα λοιπόν να επαναλάβω αυτό που είπατε και εσείς εδώ σήμερα. Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο θα πρέπει σε ψήφισμά του και μάλιστα πριν τον Δεκέμβριο. Θα πρέπει λοιπόν να καταγράψουμε τι περιμένουμε ως σημαντική πρόοδο. Ε, πώς δηλαδή θα πρέπει να κλείσει η πρώτη φάση των διαπραγματεύσεων. Και θα πρέπει ε, να μην κάνουμε καμία υποχώρηση στο θέμα αυτό. Το θέμα της Βόρειας Ιρλανδίας ε, καθώς ε, και το θέμα της ε, οικονομικής ρύθμισης θα πρέπει να εξεταστούν και να αξιολογήσουμε τα στοιχεία που θα έχουμε στη διάθεσή μας από τις διαπραγματεύσεις. Και κατόπιν θα πρέπει να δούμε πώς θα προχωρήσουν τα πράγματα. Και νομίζω ότι και αυτό είναι προς συμφέρον και ε, της British in Million, ε, και το, το British in Europe και των ε, τριών εκατομμυρίων. Θα ήθελα να πω σαφώς ότι το Brexit δεν επιτρέπεται να διακυβεύσει τις συνθήκες διαβίωσης. Και αυτό που αναφέρατε εσείς σήμερα είναι ένα πολύ δύσκολο εμπόδιο. Είχαμε δημοψήφισμα, έχουμε τη θέση του Ηνωμένου Βασιλείου. Ε, θα πρέπει όμως και η Ευρωπαϊκή Ένωση ε, να ε, δεχθεί ότι ε, το Brexit επηρεάζει τις συνθήκες διαβίωσης των ανθρώπων, δεν επιτρέπει όμως να μειωθεί το επίπεδο η φάση 1 λοιπόν και η φάση 2 συνδέονται πολύ στενά μεταξύ τους. Κλείνοντας όμως ε, θα ήθελα να πω ότι έτσι όπως βλέπω εγώ το θέμα και ε, όπως το βλέπει και η πολιτική μου ομάδα θα προσπαθήσουμε όλες ε, τις πληροφορίες που λαμβάνουμε να τις διαθέσουμε στους πολίτες ώστε να γνωρίζουν ποιο είναι το αντικείμενο των διαπραγματεύσεων και που βρισκόμαστε. και θα πρέπει να δούμε πώς θα προχωρήσουν τα πράγματα το 2018 και πώς θα προχωρήσουμε στη φάση 2. Νομίζω ότι και αυτό είναι μια σημαντική σκέψη, την οποία θα πρέπει να συζητήσουμε μεταξύ μας. Σας ευχαριστώ πολύ. Thank you, Helmut. Ευχαριστώ, Χελμούτ. Θα ήθελα τώρα να δώσω το λόγο στον κύριο Χαραγέ Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Θα μιλήσω ισπανικά. Πρώτα απ' όλα, συμμερίζομαι απόλυτα τη σημασία των όσων μας είπατε. Και θέλω να σας πω επίσης ότι γνωρίζω ότι σε όλες τις χώρες υπάρχει ισχυρό κίνημα, ιδιαίτερα στην Ισπανία το γνωρίζω βέβαια, των πολιτών, των Άγγλων, των Βρετανών που ζουν στην Ισπανία. Μας μετέφεραν τις ίδιες ανησυχίες που μεταφέρετε κι εσείς. Και οι δήμοι πολλών ε, ισπανικών ε, πόλεων που έχουν πολλούς Βρετανούς ε, κατοίκους, 400.000 είναι συνολικά από ό,τι φαίνεται, το χειμώνα κυρίως, σε πολλές ισπανικές πόλεις, τις ακτές. Βλέπουμε λοιπόν, ως το είπαν ότι υπάρχει μεγάλο τέτοιο κίνημα. Και είναι σημαντικότατο σε αυτόν τον αγώνα. Και συγχαρητήρια που οργανώσατε την κοινωνία των πολιτών και ήρθατε εδώ να την εκπροσωπήσετε. Το πρώτο είναι ότι εδώ στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο υπάρχει θα έλεγα πλήρη συμφωνία να σας στηρίξουμε όπως είπε και ο κύριος Σόλτς, όπως είπε και ο Ρίτσαρτ Κόρπιν. Όλες δηλαδή οι πολιτικές δυνάμεις συμφωνούν. Και να ξέρετε ότι δεν είναι εύκολο να συμφωνούν όλες οι πολιτικές δυνάμεις εδώ, γιατί είμαστε διαφορετικές μεταξύ μα. Αλλά όλο περιέργως για το θέμα αυτό υπάρχει περίπου ομοφωνία να στηρίξουμε τα δικαιώματα των πολιτών, των τριών εκατομμυρίων και του ενό εκατομμυρίου, χοντρικά τέλο πάντων τα λέω. Εδώ συμφωνούμε απόλυτα. Επίση θέλω να σα μεταφέρω και την πεποίθηση ότι οι διάφοροι εκπρόσωποι των πολιτικών ομάδων με τον ε, κύριο Φερχόφσταθ που εκπροσωπεί το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο στη διαπραγμάτευση έχουν σαν κύριο ε, στοιχείο και αίτημα η προστασία των δικαιωμάτων των πολιτών μας. Πριν από μερικούς μήνες εδώ στην Επιτροπή αυτής Δεγματικών Υποθέσεων είχαμε κάποιους εμπειρογνώμονες που μας μίλησαν για τα κεκτημένα δικαιώματα. Και δυστυχώς η έκθεση των εμπειρογνωμόνων έλεγε ότι τελικά δεν υπάρχουν τέτοια δικαιώματα κεκτημένα στην περίπτωση του Brexit. Δεν υπάρχει δηλαδή η διεθνής δικαιοδοσία η οποία να λέει ότι τα δικαιώματα αυτά δεν μπορούν να παραβιαστούν, γιατί δεν υπάρχει κάτι τέτοιο. Αυτό βέβαια έρχεται σε αντίθεση με αυτά που θέλουμε και μας οδηγεί στο ότι η διαπραγμάτευση είναι αυτή η οποία πρέπει να θέσει το νέο νομικό πλαίσιο των δικαιωμάτων σας και όχι προηγούμενες συμφωνίες, γιατί δεν υπάρχουν. Αυτό είναι πολύ σημαντικό στις διαπραγματεύσεις αυτές για τον Brexit. Οπότε αυτό που κάνει το Κοινοβούλιο και αυτά που θα καθορίσει η συμφωνία είναι καθοριστικά. Η συμφωνία αποχώρησης του Ηνωμένου Βασιλείου και η συμφωνία μετάβασης, γιατί θα υπάρχει και αυτή η συμφωνία για τη μεταβατική περίοδο προκειμένου να παραμείνει στην αγορά δύο με πέντε χρόνια, στην εσωτερική αγορά δηλαδή το Ηνωμένο Βασίλειο. Αυτή η συμφωνία είναι καθοριστική για σας και τα δικαιώματά σας. Και όλες οι πολιτικές ομάδες εδώ στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο συμφωνούν μαζί σας. Μπορεί να μην είναι εδώ σήμερα, αλλά το λέω εκ μέρους και των άλλων πολιτικών ομάδων που δεν μπορούν να είναι εδώ, ότι, να ξέρετε, όλοι σκεφτόμαστε λίγο πολύ όπως εμείς, όπως ο Ρίτσαρντ, ο Χέλμοντ και εγώ. Είναι επίση σημαντικό στο τέλος αυτής της μεγάλης διαδρομής, γιατί θα είναι μακρύς ο αγώνας, θα πρέπει να λάβουμε υπόψη μας την, ε, τη Χάρτα Θεμελιωδών Δικαιωμάτων, τον Ευρωπαϊκό Χάρτη Θεμελιωδών Δικαιωμάτων που λέει ότι μπορεί κανείς να απευθυνθεί στο δικαστήριο του Στρασβούργου ή του Λουξεμβούργου και να αποτελούν χώρους στους οποίους να μπορεί κανείς να αποφανθεί για να υποστηρίξει τα προηγούμενα δικαιώματά του. Αυτά στο τέλος. Στο μεταξύ όμως σας λέω ότι είναι ένα σημαντικός αγώνας που δίνετε και καλά κάνετε και μέσα από τις οργανώσεις σας υποστηρίζετε τα δικαιώματα των πολιτών και πρέπει να ξέρετε το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο είναι στο πλευρό σας. Ευχαριστώ. Ευχαριστούμε. Μερτσέδες Μπρέσο. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Οι συναδέλφοι μου ήδη είπαν ε, όλα ήθελα και εγώ να πω όλα όσα υποστηρίζει και το Κοινοβούλιο παρότι εδώ είμαστε ελάχιστε ε, ομάδες το Κοινοβούλιο έχει δεσμευτεί για την υπεράσπιση των δικαιωμάτων των πολιτών θα έχετε δει και τα ψηφίσματα τα είπαμε όλα με μεγάλη σαφήνεια πρόσφατα ε, βρέθηκα στο Μάντσεστερ και στο Λονδίνο και συνάντησα εκπροσώπους και του κινήματος 3 ε, Millions ε, της ε, Ιταλικής κοινότητας και πρέπει να πω ότι όσο περισσότερο σας ακούω τόσο περισσότερο ανησυχώ διότι τα προβλήματα που αναδύονται λόγω των διάφορων περιστατικών που ακούμε όλο ένα και αυξάνονται και ακούμε όλο και περισσότερα περιστατικά όσο μιλάμε με κόσμο αυτό είναι πολύ ανησυχητικό, διότι η συμφωνία είναι τύπου που είπε μία από εσάς τις δύο ότι τα δικαιώματα δεν πλήττονται από το Brexit ε, παραμένουν όσοι είχαν προηγουμένως ή βάζουν μέσα σε αυτά διάφορα σε σφήνες ε, που μπορεί να οδηγήσουν σε υπονόμευση της κατάστασης, σε επιδείνωση των καταστάσεων. Οι αλλαγές που γίνονται σε μικρές λεπτομέρειες ε, στο ε, σημερινό καθεστώς που απολάβουν οι Βρετανοί πολίτες στην Ευρώπη και η Ευρώπη στο Ηνωμένο Βασίλειο, αυτές οι σφήνες μπορεί να δημιουργήσουν διενέξεις και συγκρούσεις παρότι στην αρχή το ζήτημα της δικαιοδοσίας φαινόταν να μην είναι τόσο σημαντικό, εγώ έχω αρχίσει να ανησυχώ, διότι όπως φαίνεται μπορεί να γίνει ιδιαίτερα σοβαρή η κατάσταση. Και ε, μέχρι να βρεθεί μια καλή λύση θα είναι δύσκολο να φανταστούμε τι θα γίνει στις διάφορες περιπτώσεις και θα υπάρξουν σίγουρα προσφυγές. Οπότε θα πρέπει να υπάρχει μια σαφή δικαιοδοσία και αυτό είναι πολύ ανησυχητικό όταν μιλάμε για εκατομμύρια ανθρώπου. Εκεί υπάρχει κίνδυνο καθυστερήσεων, ε, καταστάσεων που θα εκκρεμούν ε, για οικογένειε, για παράδειγμα. Γι' αυτό το λόγο πιστεύω ότι πρέπει να καταβάλουμε προσπάθειε ώστε το όλο πλαίσιο να γίνει όσο το δυνατόν πιο απλό και σαφέ. Και κυρίω ε, να δώσουμε να καταλαβούν όλοι οι συνομιλητέ ότι απαιτείται μια ειλικρινή, ε, ε, ανοιχτόμυαλη ερμηνεία με κατανόηση του γεγονότος ότι ε, όλο αυτό το θέμα αφορά τόσους πολλούς ανθρώπους πριν καταλήγει κανείς σε δικαστήρια να υπάρχει κάποια ερμηνεία ε, σαφής ε, από τις διοικήσεις και της Βρετανίας και της Ευρώπης. Γνωρίζουμε πολύ καλά ότι το ζήτημα της ελευθερής κυκλοφορίας ε, στις 27 χώρες πως έχει όταν κάποιος κατοικεί σε μία από αυτές τις χώρες. Αυτό είναι σαφές. Αυτό είναι σίγουρα ένα διαπραγματευτικό χαρτί ένα διαπραγματευτικό χάρτη που μπορεί να χρησιμοποιήσει η Ευρωπαϊκή Ένωση για να διατηρήσει και μια καλή συμφωνία για τους δικούς της πολίτες. Αλλά εγώ πιστεύω ότι κανείς από εμάς δεν φαντάζεται ότι είναι δυνατόν να κινητοποιήσουμε τον καθένα από εσάς σε μια χώρα χωρίς να το δίνουμε την ελευθερία κυκλοφορίας. Ε, οπότε είναι σαφές ε, πώς έχει αυτό το πρόβλημα. Το τελευταίο που ήθελα να πω, αυτό που ανησυχεί όλο και περισσότερο, και από ό,τι κατάλαβα ανισχύει και τον Ρίτσαρντ, είναι ο κίνδυνος να μην καταλήξουμε σε συμφωνία. Διότι αν υπάρξει συμφωνία μπορεί να έχει κάποια κενά, αλλά τα θεμελιώδη δικαιώματα θα προστατεύονται. Αλλά αν δεν καταλήξουμε σε συμφωνία, τότε ε, η κατάσταση θα, και τα πράγματα θα είναι πραγματικά σοβαρά. Εγώ πιστεύω ότι και εμείς ως Κοινοβούλιο ε, θα έπρεπε να αρχίσουμε να ε, λαμβάνουμε υπόψη μας και αυτό το ενδεχόμενο και να σκεφτούμε σε περίπτωση μη συμφωνίας πώς θα μπορέσουμε να βρούμε ελάχιστα εχέγγυα αν μη τι άλλο για τους ε, πολίτες αμφωτερών των μερών διότι η κατάσταση αρχίζει να μας ανησυχεί όλους. Πραγματικά, στην αρχή θεωρούσαμε ότι το ζήτημα ε, ήταν ζήτημα λεπτομεριών ουσιαστικά, αλλά όπως φαίνεται, όπως αποδεικνύεται, μπορεί η κατάσταση να αποδειχθεί ιδιαίτερα περίπλοκη και δυσχερής. Εσείς τα έχετε εξετάσει όλα αυτά, έχετε κάποιες προτάσεις. Εμείς προς το παρόν δεν τα λαμβάνουμε υπόψη, αλλά το σενάριο αυτό πρέπει να το έχουμε στο νου μας, πρέπει να μας απασχολήσει ώστε να μην βρεθούμε απροετοίμαστε επειδή ο χρόνος περνάει ε, δεν μένει πολύ και από την εντύπωση που έχουμε σχηματίσει το Ηνωμένο Βασίλειο φαίνεται να δυσκολεύεται να ξέρει τι θέλει και συνεπώς να διαπραγματευτεί με συνοχή φαίνεται να πηγαίνουν τα πράγματα πέρα δόθε λίγο βέβαια η θέση του Ηνωμένου Βασιλείου και καθιστά τα πράγματα εξαιρετικά απορρίπλοκα ο συνομιλητής μας φαίνεται να αλλάζει απόψη κάθε λίγο και λιγάκι ή να αλλάζει άποψη ανάλογα με το συνομιλητή του. Και αυτό μας ανησυχεί ιδιαίτερα. Μαζί λοιπόν με το ζήτημα της δικαιοδοσίας αυτό που με ανησυχεί περισσότερο είναι το κατά πόσο θα καταφέρουμε να επιτύχουμε μία ε, πάγια ε, συμφωνία ε, για την οποία θα δεσμευτούν οι διοικήσεις οι οποίες θα την εφαρμόσουν με τρόπο υπέρ των πολιτών, όχι υπέρ της διοίκησης, ούτε υπέρ του περιορισμού των δικαιωμάτων, υπέρ της ουσιαστικής ε, και όχι μόνο στα χαρτιά ε, προστασίας των δικαιωμάτων. Ευχαριστούμε. Ευχαριστούμε Μερτσέντες. Ήθελα να πάρω κι εγώ τον λόγο, αφού δεν θέλει κάποιος άλλο τον λόγο. Και ζητώ συγγνώμη καταρχάς ε, για την καθυστέρηση. Είχα ε, δουλειά σε μια άλλη κοινοβουλευτική επιτροπή και δεν μπορούσα να φύγω, οπότε ίσως τα πράγματα που θα πω να έχουν υποθεί ήδη. Εγώ ήθελα να ε, σημάνω τον κόδωνα του συναγερμού για αυτό το δικαίωμα των δικαιωμάτων των πολιτών. Ευχαριστώ ιδιαίτερα τους φίλους από τους 3 Million και τους British in Europe που πραγματικά ε, μάχονται με τρόπο αξιοθαύμαστο και πολύτιμο για ολόκληρη την Ένωση. Πολύτιμο διότι αφορά το ζήτημα των δικαιωμάτων της ελεύθερης κυκλοφορίας σε ολόκληρη την Ένωση. Το καμπανάκι του συναγερμού θα ήθελα να το σημάνω για δύο σημεία. Πρώτον για το ζήτημα της επαρκούς πρόοδου, του sufficient progress. στην πραγματικότητα γνωρίζουμε ότι η κατάσταση είναι περίπλοκη, διότι έτσι θέλουν. Θέλουν να είναι περίπλοκη. Όλοι γνωρίζουμε πολύ καλά όσον αφορά τους πολίτες τι θα πει επαρκής πρόοδος. Οι αρμόδιοι, οι διαπραγματευτές από την αρχή έχουν πει ότι το Brexit δεν θα πρέπει να αλλάξει την καθημερινότητα των πολιτών. και συνεπώς θα έπρεπε να δράσουν ανάλογα. Ενώ αυτό που βλέπουμε να διαπραγματεύονται τώρα είναι το settled status ε, που πρότεινε το Ηνωμένο Βασίλειο ένα καθεστώς δηλαδή ε, κατώτερο σε σχέση με αυτό που έχουν σήμερα οι Ευρωπαίοι πολίτες ε, στο Ηνωμένο Βασίλειο και οι Βρετανοί στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Συζητούν δηλαδή διάφορες διαδικασίες, τα, ε, δύσκολες λεπτομερείς ε, δαπανηρές. το οποίο δεν συνάδει με την αρχική ιδέα ότι δεν θα έπρεπε να αλλάξει το καθεστώς για τους πολίτες. Οπότε αυτή η επαρκή πρόοδο φοβάμαι ότι και στο δικό μας κοινοβούλιο σε μέρος του κοινοβουλίου μας ε, ε, λέμε ότι έχει γίνει κάποια πρόοδος ενώ δεν έχει σημειωθεί. Δεν είναι δηλαδή ότι θα είμαστε όλοι ομόφωνοι εδώ πέρα σε όλες τις ομάδες του Κοινοβουλίου. Το δεύτερο που ήθελα να πω είναι μια ερώτηση που θα ήθελα να απευθύνω στις φίλες εδώ ε, των British Europe και των 3 Millions. Αφορά μια μάχη που έχω πραγματοποιήσει εγώ από την αρχή μαζί σας ε, για την ε, περιχαράκωση των δικαιωμάτων των πολιτών. Για την ανάγκη αυτή να τους προστατέψουμε από τις συνέπειες των διαπραγματεύσεων, να τους ε, περιφράξουμε κατά κάποιο τρόπο. Κατά την άποψή μου θα πρέπει να εμβαθύνουμε στο εξής, να εμβαθύνουμε ε, τον, στον ορισμό αυτής της περιχαράκωσης και εδώ έρχεται το δεύτερο κουδουνάκι του συναγερμού μου ε, το καμπανάκι του συναγερμού ακούγοντα τον Παρνιέ σχηματίσα την εντύπωση ότι για κάποια δικαιώματα ε, ετοιμάζονται να τα διαπραγματευτούν στη δεύτερη φάση των διαπραγματεύσεων και ειδικότερο το ζήτημα της ελεύθερης κυκλοφορίας των πολιτών, των Βρετανών πολιτών στην Ένωση των 27. Ε, την κατάσταση των διασυνεριακών εργαζομένων, την αναγνώριση μιας σειράς ε, ε, πολιτικών και αυτό που διακρίνω είναι ένας κίνδυνος. Κάποια δικαιώματα να τα προστατεύσουμε χάρη στην συμφωνία αποχώρησης, αλλά τα υπόλοιπα δικαιώματα να μείνουν έξω. Και αυτά τα δικαιώματα θα συζητηθούν στο πλαίσιο των διαπραγματεύσεων για τις εμπορικές συμφωνίες. Αυτό είναι που με φοβίζει, ότι κάποια δικαιώματα θα τα αφήσουν να πάνε στη φάση 2, να συζητηθούν στη φάση 2. Οπότε κατά την απόψή μου, ακόμη και απόψη ορολογίας, πρέπει να πούμε ακριβώς τι είδους περιχαράκωση θέλουμε ring fencing. Θέλουμε όλα τα δικαιώματα να συμπεριληφθούν στην συμφωνία αποχώρηση ακόμη και αυτά που αυτοί αυτή τη στιγμή προσπαθούν να τα αφήσουν για τη δεύτερη φάση των διαπραγματεύσεων. Η αυτό να έχει ήδη συζητηθεί σήμερα και να μην ήμουν εδώ και να μιλάω εκτός θέματος τώρα, αλλά είναι κάτι που με ανησυχεί ιδιαίτερα αυτός ο ακριβής ορισμός του ring fencing της περιχαράκωσης. Θέλει κάποιος ε, και κάποιο άλλος, ε, άλλοι βουλευτέ να μιλήσουν. Ο Χέλμουτ, παρακαλώ. Ευχαριστώ, κυρία Πρόεδρε. Ήθελα να επανέλθω στην παρατήρηση της Μερσέντες, όταν είπατε πέραν όλων των νομικών ζητημάτων που πρέπει να αναλύσουμε και να λάβουμε υπόψη το ότι θα έχουν επιτύχει τα πραγματευτικέ ομάδε κτλ. κτλ. Εμεί ω Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο θα πρέπει να αποσκοπούμε σε μια πολιτική διακήρυξη, μια πολιτική συμφωνία που θα λέμε σαφώς από πλευράς μας ποιο θα είναι το benchmark, ε, αν σας κατάλαβα καλά. Το σημείο αναφοράς δηλαδή ότι πέραν των διαπραγματεύσεων χρειαζόμαστε και μια πολιτική διακήρυξη, μια πολιτική δήλωση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου που θα συνοδεύει δύο πλευρές ε, ίσως να μην είναι επαρκή, γιατί αυτές διαπραγματεύονται μεταξύ τους το κοινοβούλιο θα πρέπει να πει με μεγάλη ακρίβεια ότι στη φάση 1 που αφορά τα δικαιώματα των πολιτών τα δικαιώματα των πολιτών πρέπει να έχουν προτεραιότητα να μην τα πετάμε δεξιά και αριστερά και να τα αφήνουμε έρμεο του κάθε συμφέροντος να υπάρξει δηλαδή μια πολιτική θέση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και να παίξει ε, σημαντικό ρόλο ώστε να συμφωνήσουν και οι δύο πλευρές. Όπως είπατε υπάρχουν, ακούμε αυτά τα, τα κουδουνάκια που μας προειδοποιούν. Πρέπει να επιταχύνουμε να καταλάβουμε τι συζητάμε όταν συζητάμε για αυτή την κόκκινη γραμμή που εκφράζουμε στο ψήφισμά μας το 2016. Και κάτι άλλο που θεωρώ σημαντικό ο ορισμός της επαρκούς προόδου θα πρέπει να διασαφινιστεί νομικά. Μπορούμε να ζητήσουμε λοιπόν από την νομική μας υπηρεσία να μας ε, δείξει τι θα πει επαρκής πρόοδος που είναι πολιτικός όρος να μας πούν λοιπόν σε ποιο βαθμό σχετίζεται με, την, ε, με τις ε, γραμμές που έχουμε υθετήσει στο ψήφισμά μας ως Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο όσον αφορά τις διαπραγματεύσεις για τον Brexit. Ναι, Χέρμοντ. Δεν νομίζω ότι υπάρχει νομικός ορισμός της επαρκούς πρόοδου. Θα αποτελέσει αντικείμενο πολιτικής απόφασης. Όπως και να έχει. Θα ήθελα να δώσω το λόγο στις προσκεκλημένες μας. Σας ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε. Σας ευχαριστώ για την υποστήριξη που εκφράσατε εδώ σήμερα. Είμαστε ευγνώμονες για αυτήν μετά από τις συναντήσεις που είχαμε τις τελευταίες εβδομάδες. Κρίσιμο είναι ότι εκφράσατε τις ανησυχίες σας σχετικά με τη διαπίστωση της επαρκούς πρόοδου. Και η ε, οργάνωση τα 3 εκατομμύρια και British in Europe ε, δεν ε, θα θέλαμε να δούμε να ε, εφαρμόζονται τελικά οι προσφορές που έχουν δοθεί αυτή τη στιγμή και από τις δύο πλευρές, ε, οι προτάσεις που έχουν δοθεί και από τις δύο πλευρές του διαπραγματευτικού τραπεζιού. Ε, σημειώνουμε αυτά που είπατε για το ring fencing, την, την περιχαράκωση, την απομόνωση των θεμάτων αυτών και το ερώτημα είναι Εάν τα πετύχουμε όλα αυτά, θα πρέπει να έχουμε άμεσα δικαιώματα που να έχουν κάποιο νόημα. Αν απλά έχουμε ε, ε, άμεση πρόσβαση στο δικαστήριο, αυτό είναι καλύτερο από το τίποτα, ιδιαίτερα σε περίπτωση ε, μη επίτευξης συμφωνίας, αλλά δεν είναι αρκετό. Θέλουμε λοιπόν διαφύλαξη όλων των δικαιωμάτων. Τον Μάιο είδαμε την πρόταση της Ευρωπαϊκής Ένωσης ε, και διαπιστώσαμε ότι αυτό θέλαμε και αυτό συνεχίζουμε να θέλουμε και θα ήθελα να κλείσω λέγοντας ότι κατοικώ στο Λουξεμβούργο, προέρχομαι από την Βόρεια Αγγλία και έχουμε το εθνικό σύνθημα ότι θέλουμε να παραμείνουμε ως έχουμε. Και νομίζω ότι ακριβώς αυτό θέλουμε να πετύχουμε και ελπίζουμε να το πετύχουμε αυτό με την υποστήριξη του Κοινοβουλίου. Σας ευχαριστώ. Ευχαριστώ, Φιώνα. Να πω απλά ότι στηρίζω απολύτως αυτά που είπε η Φιώνα. Οι ζωές μας διακυβεύονται τώρα. 122-123.000 πολίτες της Ευρωπαϊκής Ένωση, υπηκόοι τη Ευρωπαϊκής Ένωση, έχουν εγκαταλείψει το Ηνωμένο Βασίλειο μετά το δημοψήφισμα. Νομίζω ότι τα νούμερα μιλάνε από μόνα του. Πολλοί άνθρωποι όταν ε, αποχωρούν ε, δεν επιστρέφουν απαραίτητα στις πατρίδες τους. Άλλωστε ε, δεν έχει νόημα κάτι τέτοιο. Κάποιος που έχει μείνει στο Ηνωμένο Βασίλειο επί 35 χρόνια, εκεί έχει πια το σπίτι του. Ε, πολλοί θέλουν να συνεχίσουν ε, να ζουν ε, το ευρωπαϊκό εγχείρημα. Επίσης, πολλοί κόσμοι που αποχωρεί από το Ηνωμένο Βασίλειο παίρνει μαζί τους και τις δουλειές τους, τις επιχειρήσεις τους. Και αυτό αποτελεί μεγάλη απώλεια για το Ηνωμένο Βασίλειο. Και βλέπουμε και περισσότεροι Βρετανοί να εγκαταλείπουν το Ηνωμένο Βασίλειο. Δεν εγκαταλείπουμε μόνο εμείς οι Ευρωπαίοι το Ηνωμένο Βασίλειο. Πολλοί Βρετανοί λοιπόν νιώθουν ότι είναι και Ευρωπαίοι πολίτες και θέλουν να ζήσουν στην Ευρώπη. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ πολύ. Η Τζέιν. Απλά να προσθέσω ότι υποστήριζω τόσο όσα είπαν η και η Φιώνα και ήθελα για άλλη μια φορά να επαναλάβω αυτά που είπαμε ε, για τους εργαζομένους οι οποίοι πήγαν και έφτιαξαν τις ζωές τους βάσει της ευρωπαϊκής ηθαγένειας. αποκτήσαμε όλα αυτά τα δικαιώματα και τα επεκτείναμε πέρα από ότι ε, ήταν η πρόθεση των αρχικών δημιουργών τους. Ε, έχουμε ζήσει όχι σε μία χώρα παρέτα, αλλά και σε πολλές χώρες και όλοι θεωρούμε τους αυτούς μας Ευρωπαίους. Αυτό ήθελα να παραλάβω. Ευχαριστώ. Ευχαριστούμε. Κλείνουμε το θέμα εδώ. Να σας ανακοινώσω τις επόμενες συνεδριάσεις. Τακτική συνεδρίαση 3η 28 Νοεμβρίου στις 9 μέχρι τις 12.30 και μετά το απόγευμα από τις 2.30 μέχρι τις 6.30. Ε, ε, σας αποχαιρετώ.